everybody to the European Parliament. Καλώς ορίσατε κυρίες και κύριοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων 2018. Θέλω να σας ζητήσω παρακαλώ να λάβετε τις θέσεις σας. Ladies Κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη χαρά μου που σας καλωσορίζω στη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Επιχειρήσεων για το 2018. Ε, ξέρετε, η παγκόσμια γλώσσα της ε, μουσικής ε, μας ενώνει. Θέλω λοιπόν να σηκωθούμε όλοι και να ακούσουμε τον Ευρωπαϊκό ύμνο. Ευχαριστώ. Και τώρα, με ιδιαίτερη χαρά, θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού επιχειρηματικού ε, οργανισμού που εκπροσωπεί 20 εκατομμύρια επιχειρήσεων, εκ των οποίων πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Κρίστοφ Φλάιτεν.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 756 συμμετέχοντες. Τόσοι είμαστε που μαζευτήκαμε σήμερα εδώ και φυσικά θέλω θερμά να καλωσορίσω και τις κυρίες που είναι ανάμεσά μας, διότι οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι μια από τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης. Ich begrüße die Teilnehmerinnen. Και βεβαίως καλωσορίζω και τις συμμετέχουσες και συμμετέχοντες από 34 διαφορετικές χώρες, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέρος της κοινότητάς μας, που ανήκουν σε αυτή την ευρωπαϊκή οικονομία. Από πολιτικής άποψης ε, υπάρχει πολλή δουλειά πρέπει να γίνει ακόμη, πάντως οικονομικά είμαστε ενωμένοι και δεν είναι πρώτη φορά που η οικονομία προπορεύεται σε σχέση με την πολιτική. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που σας έχω σήμερα όλους εδώ. Είμαι περήφανος για την παρουσία σας εδώ, διότι έχουμε όλοι προσδοκίε, Έχετε και εσείς προσδοκίες, φιλοδοξίες, επιθυμίες που θέλετε να εκφράσετε και σήμερα θέλουμε να παρουσιάσουμε την Ευρώπη της οικονομίας και θέλετε κι εσείς να τα συζητήσετε όλα αυτά, να καταλήξετε σε αποφάσεις οι οποίες στη συνέχεια θα δώσουν ένα προσανατολισμό στο Ευρωεπιμελητήριο. Θέλουμε να σας ακούσουμε, θέλουμε να ακούσουμε το μήνυμά σας προς τα πού πρέπει να κινηθούμε και να κατευθυνθούμε. Εσείς θα μας το πείτε. Επιτρέψτε μου όμως πριν από όλα να χαιρετήσω όλους όσοι δεν παρευρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας. Τα μέλη από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι θέσεις σας είναι κενές σήμερα. Όμως μπορώ να σας διαβεβαιώσω για ένα πράγμα. Αν επιθυμείτε να επιστρέψετε, η αγκαλιά μας θα μείνει ανοιχτή, καθώς και η καρδιά μας. Ας ελπίσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις ε, σχετικά με το Brexit θα μας οδηγήσουν έτσι σε κάποια πρόοδο, έτσι ώστε να μην υπάρξει ρήξη, να μην, υπάρχουν, να μην υπάρξουν κραδασμοί και τελικώς να καταφέρουμε να μιλήσουμε για το κοινό μας μέλλον. Και για να μπορέσουμε να συναποφασίσουμε, και το λέω, το τονίζω, συναποφασίσουμε, διότι είναι σημαντικό για εμάς και στην οικονομία, είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, μας, ε, αφορά το Brexit. Θέλουμε οπωσδήποτε να ελαχιστοποιήσουμε τις ε, βλάβες και να συνεχίσουμε με την Ενωμένη Ευρώπη. Ε, καλωσορίζω επίσης και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Ταγιάννη, ο οποίος θα έρθει ανάμεσά μας σε λίγα λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ που μας θέσατε στη διάθεσή μας το ημικύκλιο και είμαι ιδιαίτερος ευτυχής που διαπιστώνω ότι ε, τελικώς ε, συνεργάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Ευρωεπιμελητήριο πάρα πολύ στενά και εκπροσωπούν και το Ευρωεπιμελητήριο όταν πηγαίνουν στην Ευρώπη σε κάποια άλλη χώρα ή και αλλού στον κόσμο. Αυτό μας δίνει πολύ κουράγιο, πολύ θάρρος και τον ευχαριστούμε τον κύριο Ταγιάννη γιατί εμπλέκεται προσωπικά σε όλο αυτό. Αυτός ο οίκος είναι το σύμβολο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και ένα σύμβολο των ευρωπαϊκών αξιών. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια φάση ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων συστημάτων διακυβέρνησης. Κάποιες ε, χώρες είναι ιδιαίτερα περήφανες σήμερα διότι θεωρούν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πιο αποδυναμωμένο ρόλο ε, θεωρούν ότι είναι καλύτερο να παίρνουν ε, αποφάσεις που δεν συνάδουν απαραίτητα με τη βούληση των λαών όμως είναι πολύ σημαντικό να ακούμε τους πολίτες, είναι σημαντικό να ακούμε τα μηνύματά τους και να εντάσσουμε τα μηνύματά τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εμείς γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι, για την δημοκρατική αυτή αρχή που μας διέπει και είμαστε επίσης υπερήφανοι διότι όσον αφορά την πολιτική έχουμε μία θέση η οποία τελικώς προκύπτει από τον σεβασμό της πολιτικής προς την οικονομία. Γιατί εμείς, η οικονομία, δημιουργούμε θέσεις απασχόλησης. Εμείς δίνουμε δουλειά σε 120 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη. Εμείς δημιουργούμε, εκπαιδεύουμε ταλέντα στην Ευρώπη. Εμείς πληρώνουμε ε, φόρους στην Ευρώπη έτσι ώστε η πολιτική ακριβώς να μπορεί να ενισχύει τα κοινωνικά συστήματα και γι' αυτό είμαστε επίσης πολύ υπερήφανοι. Αλλά αφού καταφέρουμε να κάνουμε όλα αυτά για την κοινωνία, αναμένουμε βεβαίως και τον απαραίτητο σεβασμό. Να σέβονται δηλαδή και τις συνθήκες πλαίσιο που έχουμε, έτσι ώστε και στο μέλλον να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε το ρόλο μας. Και επίσης είμαι πολύ ευτυχής που διαπιστώνω ότι στο μέλλον θα έχουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε να συνεχίσουμε να ε, σχεδιάζουμε από κοινού το μέλλον της Ευρώπης. Έχουμε πολλές αμφιβολίες, πολλά ερωτηματικά. Κάποιοι απελπίζονται με τόσα, ε, με τόσα ερωτηματικά, αλλά όχι οι εταιρείε, οι επιχείρησεις, γιατί σε κάθε κρίση βρίσκουμε ότι υπάρχει κάποια ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Υπάρχουν θετικά ευνοϊκά πράγματα που κρύβονται πίσω από μια κρίση και εμείς πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτές τις δυνατότητες, να είμαστε δημιουργικοί για να μπορέσουμε και εμείς να σχηματίσουμε το μέλλον της Ευρώπης, να βοηθήσουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να ενθαρρύνουμε τους Ευρωπαίους να μην φοβούνται το μέλλον, αλλά να έχουν το, το, το θάρρος ε, να κινηθούν προς ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον και θα πρέπει να μπορούμε βεβαίω να υπολογίσουμε και να ποντάρουμε και στην νεολαία μας και χαίρομαι που βλέπω εδώ νέου ανθρώπου ανάμεσά μας γιατί εσείς είστε οι νέοι που θα ζήσετε αύριο. Εσείς πρέπει μαζί να δουλέψετε με εμά για να σχεδιάσουμε το αύριο. Μαζί σας πρέπει να συνεργαστούμε, πρόκειται για το δικό σας μέλλον και θέλουμε να είμαστε περήφανοι για εσά, όταν αποφασίζετε για το μέλλον σα και δεν επιβιώνετε απλά αλλά αποφασίζετε για τον τρόπο ζωής σας, για την προσωπική σας ικανοποίηση και χαιρόμαστε ιδιαίτερα και είναι μια ευθύνη που έχουμε απέναντί σας πολύ σοβαρά, σοβαρή. Αγαπητοί εκπρόσωποι της οικονομίας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σήμερα θα ασχοληθούμε με τρία βασικά θέματα. Με το εμπόριο, Εξάλλου το μέλλον ή η ανάπτυξη της Ευρώπης Και όσον αφορά το εμπόριο, θα λέγω ότι υπάρχουν τρεις άξονες. Καταρχάς, είμαστε η πιο ισχυρή εμπορική δύναμη στον κόσμο. Το λέω, το ξαναλέω και το ξαναλέω. γιατί υπάρχουν πολλοί σχολιαστές οι οποίοι εξακολουθούν να μην το γνωρίζουν αυτό, να το αγνοούν. Είμαστε η πιο ισχυρή εμπορική δύναμη στον κόσμο και υπ' αυτή την έννοια θέλουμε να ασκήσουμε επιρροή και όχι να είμαστε ε, θύματα άλλων εμπορικών δυνάμεων. Θέλουμε να προσαρμόσουμε το εμπόριο στη βάση της, ε, των ελεύθερων ε, ανταλλαγών. Θέλουμε ευημερία, πλούτο και θέλουμε και χρησιμότητα για τον κόσμο, για τις κοινωνίες. Να δημιουργήσουμε μια αξία σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούμε το εμπόριο ως όπλο εναντίον κάποιου άλλου, αλλά είναι μια, μια γέφυρα ακόμη και τα πολιτικά συστήματα που δεν έχουν τις ίδιες αξίες με ε, το δικό μας, πρέπει να δημιουργήσουμε μια, ένα σύνδεσμο, μια γέφυρα. Πέρα από την ελεύθερη απαλλαγή, ανταλλαγή υπάρχει και το fair trade, το δίκαιο εμπόριο. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι τίποτα δεν θα γίνει χωρίς να σεβόμαστε κάποιες συγκεκριμένες αξίες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουμε στην κατάρτιση των ανθρώπων. Πρέπει όλοι οι Ευρωπαίοι να έχουν προσόντα και δεξιότητες. Αν καταφέρουμε να δώσουμε σε όλους δεξιότητες, τότε θα έχουμε πλήρη απασχόληση στην Ευρώπη. Εάν είχαν όλοι προσόντα και δεξιότητες, αν όλοι οι νέοι στην Ευρώπη είχαν δεξιότητες, το μέλλον θα ήταν πολλά υποσχόμενο. Αυτό λοιπόν πρέπει να δουλέψουμε περαιτέρω. Αλλά προσοχή. Οι εμπορικές σχέσεις θα πρέπει να είναι βιώσιμες και γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε το εμπορικό σύστημα του μέλλοντος, διότι η καινοτόμα ε, ανταγωνιστική δημιουργική Ευρώπη πρέπει να υπάρξει. Σκεφτείτε λιγάκι το, το βραβείο Νομπέλ. Πρόσφατα ε, είδαμε, ο, ε, αλλάζει ο τρόπος ζωής, έχουμε την κυκλική οικονομία. Η κυκλική οικονομία, ας πούμε, είναι στην καρδιά του προβληματισμού μας. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα με σαφείς ξεκάθαρους στόχους, μια ιδέα πρόοδου, αλλά πάντα με αλληλεγγύη απέναντι σε εκείνους που δεν έχουν αποκτήσει το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης. Να, ας πούμε, μία από τις αρμοδιότητες, ε, ένα από τα καθήκοντά μας. Πρέπει να το πάρουμε σοβαρά υπόψη. Έχουμε ένα business model όπως, όσον αφορά την ψηφιοποίηση, οπωσδήποτε, αλλά έχουμε νέα μοντέλα επιχειρησιακά ε, στο περιβάλλον, στην ε, οικονομία, στη χρήση των πόρων και όλα αυτά ε, στηρίζονται και στις εταιρικές σχέσεις με οργανώσεις, με συστήματα που μας συμπληρώνουν. Χρειαζόμαστε εταιρικές σχέσεις και κυρίως με την Αφρική. είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που εδώ μπορούμε να συζητήσουμε και για την Αφρική χωρίς να σκεφτόμαστε αναγκαστικά κάθε φορά τις ε, σωστικές λέμβους, αλλά να σκεφτούμε, να σκεφτούμε στην Αφρική με την έννοια του πώς θα αναπτύξουμε εταιρικές σχέσεις με τις ε, αφρικανικές χώρες. Έπειτα, το μέλλον της Ευρώπης Ξέρουμε γιατί είναι ασθενής η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Διότι του παρόντος δεν είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε αρκετά γρήγορες αποφάσεις. Συχνά παίρνουν άλλοι τις αποφάσεις στη θέση μας και δεν ε, είναι πάντα οι κατάλληλε και δεν συνάδουν πάντα με τις αξίες μας και με τα δημοκρατικά μας συστήματα. Αλλά οι άλλοι παίρνουν πιο γρήγορα τις αποφάσεις. Άρα και εμείς πρέπει να βρούμε τον τρόπο να διατηρήσουμε έτσι την πίστη στις αξίες μας, όντας ταυτόχρονα αποτελεσματικοί με τη λήψη αποφάσεων. Μερικές φορές οι διαδικασίες ε, ε, είναι μακροσκελείς, είναι ε, χρονοβόρες. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε και όχι να αντιδράσουμε. Και σίγουρα δεν πρέπει να παραμείνουμε ακίνητοι αναμένοντας απλώς άλλους να λάβουν αποφάσεις στη θέση μας. Χαίρομαι που έχουμε συνάψει ήδη με την Ιαπωνία την Συμφωνία Ελεύθερης, Ελεύθερων Συναλλαγών, αλλά ξέρετε αυτό χρειάστηκε 20 χρόνια για να γίνει. Τι, 20 χρόνια θα περιμένουμε, δεν είναι δυνατόν. Και ελπίζω ότι η Συμφωνία Ελεύθερων Ανταλλαγών ε, που θα περάσει με τι χώρε του Μερκοσούρ θα είναι, ε, θα, δεν θα χρειαστεί τόσο χρόνο. Και όλα αυτά τα οποία δημιουργούν προσκόμματα στην Ευρώπη, που παραλύουν την Ευρώπη, είναι αυτή η υποχρέωση για την ομοφωνία. Εντάξει, να το ξεφορτωθούμε. Γιατί έχουμε κοινοβούλιο, γιατί έχουμε δημοκρατία, για να ε, υπάρχουν ε, διάφορα επιχειρήματα, διάφορες αιτιολογίες, συζητήσεις και στο τέλος των ε, συζητήσεων να υπάρχει ψηφοφορία και να λαμβάνεται απόφαση. Αυτό είναι η δημοκρατία. Άμα ψάχνουμε ομοφωνία, τελείωσε, μπλοκάραμε. Και εφόσον δημιουργήσουμε αυτό, το, το, το μπλοκάρισμα, τότε διακυβεύουμε το μέλλον των νέων. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ως Ευρωεπιμελητήριο πρέπει να συνεισφέρουμε με τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Δημιουργήσαμε εξάλλου και ένα εργαστήριο ε, σχετικά Πώ μπορούμε να συμβάλλουμε σε μια θετική εξέλιξη τη Ευρώπη στο μέλλον. Ε, σε λίγους μήνες θα έχουμε τις ευρωεκλογές, θα έχουμε ένα, μια νέα σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε, να ταινίσουμε το ε, μέλλον. Πώς θα είναι η Ευρώπη σε πέντε χρόνια. Εδώ τίθεται θέμα στην απόφαση. Πρέπει και εμείς να της δώσουμε ένα πρόσωπο τη Ευρώπης και ελπίζω ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα δώσει κάποιες απαντήσεις σήμερα. Σας εύχομαι λοιπόν μια επικοδομητική συνάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Κρίστοφ Λάιταρ. Ε, θα δώσω τώρα τον λόγο στον εκπρόσωπο ε, της Προεδρίας του Εξαμήνου για το, του, ε, Συμβουλίου του κύριου Άντρο Πρέκτορ από την Αυστρία, ο οποίος και ε, έχει το βήμα. Ε, παρακαλούμε. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ε, αγαπητέ κύριε of Λάιτα, εξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί εκπρόσωποι των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, με τιμή μου και αισθανόμενος ε, ιδιαίτερο προνόμιο ε, προσέρχομαι εδώ στην πέμπτη αυτή συνεδρία ε, των, του Κοινοβουλίου για τις Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις που συγκερνά 575 επιχειρηματίες άνδρες και γυναίκες που προέρχονται από πάνω από 30 ευρωπαϊκές χώρες. με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι βρίσκονται εδώ συγκεντρωμένοι επιχειρηματίες και έχουν την ευκαιρία να έστω για μια μέρα να αισθανθούν μέλη του Κοινοβουλίου ε, για να ψηφίσουν και να αποφανθούν επί των πιο ακαθοδών θεμάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Μια ιδέα η οποία πήρε σάρκα και οστά στους κόρπους ε, της ε, καταπληκτικής αυτής διάσκεψης που είχε να κάνει με το κατά πόσο τελικά υπάρχει Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Επιχειρήσεων. Ήταν η επαρχία αυτής της πρωτοβουλίας. Για μένα πρόκειται αυτό να ε, ε, είναι αυτή μια ζωντανή απόδειξη για τη δυνατότητα των πολιτών και ειδικά των επιχειρηματιών να βρεθούν κοντά ένα στον άλλο. Αυτοί που είναι οι κύριοι ε, προωθητές της ευημερία και του πλούτου στην Ευρώπη είναι κάτι που πραγματικά αποτελεί επιτυχία. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας τις απόψεις και τις θέσεις της Ευρω... Αυστριακής Προεδρίας για το πώς η Ευρώπη θα μπορέσει να, δημορφώσει το μέλλον. Από το Ινσμπρουκ, το... την πατρίδα μου, σε άτυπη συνάντηση που είχα με τους αρμοδίους είχαν συζητήσεις που εστιάστηκαν γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς και για την αντίληψη που το ευρύτερο κοινό έχει περί των ευρωπαϊκών εμπορικών συμφώνων. Ε, θα το δούμε αυτό στην δεύτερη συνεδρία μας σήμερα. Πρέπει όλοι να έχουμε σαφές ότι δίκαιες και καλά ισορροπημένες εμπορικές συμφωνίες ωφελούν όλους και στο σημείο αυτό επικαλούμε τον κύριο Ζων Κλοντ Γιούνκερ πρόεδρο της Επιτροπής που την περασμένη Παρασκευή σε ομιλία στο Αυστριακό Κοινοβούλιο ε, συζήτησε λέγοντας ότι οι εμπορικές συμφωνίες είναι που κάνουν την Ευρώπη μεγάλη όπως είναι προσωπική μου άποψη είναι ότι σήμερα η διεθνή εμπορική ε, πολιτική αντανακλά ε, με πολύ εύγλωτο τρόπο την τρέχουσα συγκυρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μια πλευρά θέλουμε να είμαστε κρατεότεροι, ε, πολύ πιο ενωμένοι, πολύ πιο διεκδικητικοί. Από την άλλη πάλι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε πώς θα το πετύχουμε αυτό. Πόσο μάλλον καθώς ο χρόνος μας πιέζει μια και οι προκλήσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ε, επιμικρύνεται σε χρόνο και επιτείνονται σε ένταση. Ε, βλέπουμε να αυξάνουν τα χάσματα μεταξύ των κρατών μελών, κάτι που οδήγησε σε μια δραστική συρρήκνωση τη εμπιστοσύνη σε κυβερνήσει και, στους πολιτικούς. στου πολιτικού. Για το λόγο αυτό ακριβώ η Αυστριακή Προεδρία θέλει να κάνει τη διαφορά ε, να προτοθεί εκ νέου εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αμοιβαιότητα στην εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και εμπιστοσύνη και προ την Ένωση. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, δεν αρκούν ε, οι εύσχημοι λόγοι. Ε, σίγουρα χρειαζόμαστε δράσεις, χρειαζόμαστε ενέργειες και αυτό ακριβώς είχε κατά νου ο Όρμπερτ Σούμαν όταν είπε ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να γίνεται μια μέρα στην άλλη πραγματικότητα θα δομηθεί μέσα, και, ε, μέσα από συγκεκριμένα επιτεύγματα και ε, κατακτήσεις. Ακριβώς ε, την οικονομία και τους επιχειρηματίες είχε στο μυαλό του αυτούς που δίνουν την επιτυχία στην προσπάθεια για ευρωπαϊκή ενοποίηση. Για να επιτευχθεί αυτό η Αυστριακή Προεδρία επιλέγει ως έμπνευσή της στην αρχή της επικουρικότητας. Μας ενδιαφέρει να εντοπίσουμε τομείς πολιτικής όπου χρειάζεται ενέργεια σε ενωσιακό επίπεδο και να ενισχυθούν αυτοί οι τομείς. Και θα θέλουμε επίσης να ταυτοποιήσουμε τους τομείς εκείνης της πολιτικής που θα πρέπει να συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη ή ακόμα και σε επίπεδο περιφερειών. Ακόμα καλύτερο είναι αυτό για να δραστηριοποιηθούμε και να λάβουμε αποφάσεις. Βασική ε, έννοια πίσω από την ε, ε, ε επικουρικότητα είναι αρχές που από την αρχή διαπνέουν το, την Πάλι ποτέ ευρωπαϊκή κοινότητα. Αλλά την τελευταία φορά που σωστά συζητήθηκε αυτό ήταν στα πλαίσια τη προηγουμενη Αυστριακή Προεδρία του 2006 και πιστεύω ότι το Brexit ή τα θέματα τη μετανάστευση είναι εξαίρετε αφορμέ για να αρχίσει εκ νέου η συζήτηση αυτή. Ε, τώρα πλέον οι Βρυξέλλες πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τη φωνή και τι ανησυχίε των πολιτών και των κρατών μελών γενικότερα. Με τον λόγο αυτό η Αυστριακή Προεδρία θα διοργανώσει σε υψηλό επίπεδο διάσκεψη του Bregenz ε, γύρω στα μέσα Νοεμβριού ακριβώς για να ενισχυθεί ε, η κοινή κατανόηση ε, της αρχής της επικοροτικότητας. Έχουμε ήδη δομήσει μια ομάδα δράσης, μια task force για το λόγο αυτό. Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα μπορέσουμε όλοι να έχουμε μια Ευρώπη κρατεότερη πιο δυνατή απέναντι στα κοινά μας ζητήματα με καλύτερη ασφάλεια και πιο στεναρή αμυντική πολιτική στους τομείς εκείνους όπου και τα κράτη-μέλη αλλά και οι περιφέρειες είναι σε θέση να λάβουν αποφάσεις και μόνες τους όπως προανέφερα δεν είναι μόνο ότι αντιμετωπίζουμε πολλαπλές προκλήσεις αλλά παρατηρούμε να υπάρχουν ε, χάσματα, ρογμές και βαθιές διαιρέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Η Προεδρία λοιπόν θέλει να είναι η γέφυρα, θέλει να χτίσει γέφυρες ώστε να φτάσει μέχρι τον τελευταίο πολίτη να ακούσει όλες τι γνώμες. Ε, θέματα επί των οποίων μπορούμε όλοι να δουλέψουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και να προχωρήσουμε. Ε, σκόπιμα έχουμε επιλέξει ως ε, ρητό μα και σύνθημά μας μια Ευρώπη που προστατεύει οι πολίτες δεν περιμένουν μόνο να έχουμε μια Ευρώπη ε, βήμερη ε, και μια Ευρώπη ε, ε, προχωρημένη, αλλά θέλουμε και μια Ευρώπη ασφαλή. Για να υπάρξει αυτό χρειάζεται σταθερότητα και ευημερία σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό θα το πετύχουμε όχι μόνο ε, μέσα από εσωτερικέ δράσει, αλλά και με ενίσχυση συνόρων μα. Επίση, ε, για να επιμείνω περαιτέρω στα διάφορα θέματα που διαπνέουν την ε, ε Αυστριακή Προεδρία. Ασφάλεια και καταπολέμηση παράνομη μετανάστευση. Προστασία του Ευρωπαίου πολέτη πρέπει να είναι ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων μα. Για να μπορούμε λοιπόν να το έχουμε αυτό, πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχουμε τα εξωτερικά μα σύνορα. Σίγουρα ε, από το 2015 και μετά έχουμε χάσει τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων μα, κάτι που ε, έχει σε αποτέλεσμα την υπονόμευση τη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον πολίτη. Για το λόγο αυτό, η Αυστριακή Προεδρία χαιρετίζει την ανακοίνωση από πλευρά του κ. Γιούνκερ και τη Κομισιόν για ενίσχυση τη Frontex και για την για σχετική απόφαση του Συμβουλίου ήδη από Ιουνίου φέτο. Αλλά η ασφάλεια των εξωτερικών ε, συνόρων δεν είναι το μόνο μέτρο για να αντιμετωπίσουμε την παράνομη μετανάστευση. Η πραγματική λύση για την Ευρώπη τελικά βρίσκεται στην Αφρική. Εκείνη η απάντηση, γι' αυτό πρέπει να είναι πιο ενεργή και ισχυρή η Ευρώπη, ε, έτσι ώστε εκπρόσωποι από χώρες προέλευσης και διαμετακόμιση να συμμετέχουν στο διάλογο, να στηριχθούν αυτέ οι χώρε, να δοθούν νέε προοπτικέ για τη νέα γενιά εκεί. Θέλουμε νέε συμμαχίε με την Αφρική, νέε επενδύσει για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία. Πρέπει να ξεκινήσουν νέε ευκαιρίε για τι οικονομίε μα. Για το λόγο αυτό, η Αυστριακή Προεδρία θα διοργανώσει από κοινού με την Αφρικανική Ένωση ε, και την επιχειρηματική κοινότητα υψηλής, ε, υψηλού επίπεδου ε, διάσκεψη επιχειρηματιών στη Βιέννη το Δεκέμβριο. Σκοπός είναι να υπάρξει μακροπρόθεσμη οικονομική συνεργασία στεναρή και πολλά υπασχόμενη με τον βιομηχανικό και ε, οικονομικό κλάδο της Αφρικής για το μέλλον. Κατά δεύτερο λόγο, η Αυστριακή Προεδρία εστιάζει σε θέματα διασφάλισης της ευημερία. Ο αυτοματισμός, η ψηφιοποίηση και δημιουργία οικονομίας πλατφορμών ε, κάτι που θα αλλάξει θεμελιωδό στον κόσμο που σήμερα ζούμε. Εάν πετύχουμε να είμαστε ε, οι προτεργάτες στον τομέα αυτό, τότε θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις νέες ευκαιρίες και θα εξακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ηγέτης παγκοσμίω. Τα πάντα πρέπει να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι στο μέλλον ε, μεγάλες εταιρείες του χώρου του διαδικτύου δεν θα έχουν πια έδρα μόνο της ΕΠΑ ή την Κίνα όπως σήμερα ζούμε, αλλά θα επανέλθουν και πάλι στην Ευρώπη. Επίσης να αναλογιστούμε ποιο είναι το μέλλον της, ε, του βιομηχανικού κλάδου στην Ευρώπη ε, με τον μεταπητικό ε, κλάδο να ηγείται αυτή τη νέα ε, σειρά ευκαιριών. έτσι είναι που οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει θα δημιουργήσουν σαφώ ε, προτιθέμενη αξία. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώ έχει τα συστατικά εκείνα που θα τη επιτρέψουν να αποτελέσει ε, παγκόσμιο πρωταθλητή σε αυτή την ομάδα ε, ε, επιλέκτων της οικονομίας. Οι εξαιρετικές μας υποδομές μας, το έμψυχο υλικό μας υψηλά εξειδικευμένο και με πάρα πολλά προσόντα, με μια νέα αγορά τόσων εκατομμυρίων ανθρώπων, σίγουρα μπορούμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκε πλαίσιο εντός των οποίων η υψηλή τεχνολογία θα ηγηθεί στην Ευρώπη και όλοι μαζί θα έχουν δίκαιο πεδίο ε, ανταγωνισμού μέσα και από τις τιμαριθμικές ε, προσαρμογές. Ε, μέσα δε και από την διασφάλιση αυτής της ευημερίας, εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είμαστε πιο διεκδικητικοί, πρέπει να είμαστε πιο διεκδικητικοί παγκοσμίω. Η Ευρώπη δεν θα αρκείται πλέον στο ρόλο ενός σχολιαστή ή θεατή του παγκόσμιου γίγνεσθε. Η Ευρώπη πρέπει να είναι ενεργός ε, αρχιτέκτον και πρωτεργάτης ε, του νέου κόσμου. Ε, πρέπει να είμαστε ε, αυτοί που θα λειτουργούν ως συντελεστές, όχι μόνο ως δεύτεροι παίκτες. Αυτό σημαίνει να είμαστε ενεργοί και δραστηροί και έχει στη γειτονιά μας η Ευρώπη παράγει και εξάγει και στη γειτονιά της. Μόνο αν διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ασφάλεια στη γειτονιά μας θα είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε μακροπρόθεσμη ευημερία και σταθερότητα εντός τη Ευρώπης. Έχουμε την επιλογή μεταξύ της εξαγωγή σταθερότητα ή εισαγωγή αστάθεια. Μια είναι πολύ κοντά στην καρδιά μας σαφώς είναι η εισαγωγη ασταθειας μια περιφερεια που ειναι πολυ κοντα στην καρδια μας σαφω ειναι Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τότε μόνο θα θεωρηθεί πλήρη όταν έχουν ε, όλα τα βαλκανικά κράτη γίνει κομμάτι της Ενωμένης ΕΕ. Ευρώπης. Αυτά τα κράτη όχι μόνο αξίζουν να έχουν μια ευρωπαϊκή προοπτική, αλλά ακόμα καλύτερα ε, έχουν κερδίσει με το αίμα τους το δικαίωμα να είναι μέλη της Ένωσης και τέλος να συμπληρώσω, να τονίσω τη συνεισφορά της Αυστρίας στον όλο διάλογο σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα κορυφωθεί με την άτυπη ε, συνοδοκορυφή στο Σύμπιου ε, το Μάιο ε, του χρόνου στα πλαίσια της Ρουμανικής Προεδρίας. Η ρουμανική κρίση μας δείχνει ότι η Ευρώπη δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί ως σχέδιο. Με τον, ε, ως προς αυτό λοιπόν και με τους μετανάστες στο μυαλό μας ε, έχουμε ε, πολλά ακόμα να κάνουμε με τις διόδους που έχουμε ανοίξει έχουμε σαφώς επιλέξει την επικουρικότητα ως ε, την αρχή που θα διαπνεύσει αυτό το ευρωπαϊκό ε, σχέδιο για μια επανασυμφιλίωση ε, με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης η επικουρικότητα είναι εργαλείο συνεργασίας και όχι, Έχει, όχι ένα μέσο διαίρεσης η αρχή αυτή λοιπόν δεν πρέπει να αξιοποιείται για να διαλύει την αναξελίξη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ή οτιδήποτε άλλο καλό έχει επιτευχθεί μέσω της ε, ολοκλήρωσης. Η επικουρικότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα μέσο για μια επανενεργοποίηση του ευρωπαϊκού σχεδίου. Ολοκληρώνω, επικαλούμενο τον μόνο τον YouTube που πολύ σωστά είπε η Ευρώπη σήμερα είναι μια αφηρημένη ιδέα που χρειάζεται να γίνει συνέστημα. Με αυτά σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή επιτυχία στη συζήτησή μας ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Επιχειρήσεων και ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε τον κύριο Γκρουπρέτα. Θα ήθελα στη συνέχεια να σας δώσω κάποιες τεχνικές πληροφορίες όσον αφορά την διαδικασία της συζήτησης που θα ακολουθήσει. Η πρώτη πληροφορία είναι ότι ε, τη στιγμή αυτή μας εκπέμπουν ζωντανά από το Europe Satellite. Δορυφορικά λοιπόν ανά τον πλανήτη εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων παρακολουθούν ε, εν δυνάμει αυτό το ε, γεγονός ζωντανά σε όλο τον κόσμο, αυτή η οργάνωση. Αυτό μας παρέχει τη δυνατότητα να θέσουμε ζητήματα και μέσω των μέσων κοινωνικής διεκτύωσης, μέσω του Twitter, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό από αυτό του ημικυκλίου εδώ σήμερα. Τρία ερωτήματα λοιπόν θα σας αναφέρω τα οποία θα μπορούσαν να μας απασχολήσουν και θα πρέπει να απαντηθούν και τις επόμενες ώρες και είναι τα εξή. Το πρώτο ερώτημα, ύστερα και από τα όσα αναφέρθηκαν κάτι διάρκεια των δύο παρεμβάσεων, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ε, ένα πρόγραμμα επιδότησης ολοκλήρωσης για τις μικρομεσαίες ώστε να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες μπορείτε να απαντήσετε ναι ή όχι ε, μπαίνοντα στο Twitter account του Eurochambers Δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με θέματα εμπορίου σε μια εποχή κλιμακούμενων εμπορικών αντιπαραθέσεων και ενός επιτυνόμενου εθνικισμού τόσο εντός όσο και εκτός ένωσης έχετε τη διάθεση να συνεχίσετε να είστε ενωμένοι κάτω από μια κοινή ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική και πάλι στο Twitter account μας μπορείτε να πείτε ναι ή όχι και το τρίτο ερώτημα είναι το εξή. σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης είναι αυτό τώρα ίσως να φανεί λίγο τεχνική υφής αλλά είναι πολύ κέριο ωστόσο ε, ο κύριος Λάιτλ άλλωστε το ανέφερε και προηγουμένως και είναι το εξή. τα ψηφίσματα στο Συμβούλιο θα πρέπει να γίνονται με πλειοψηφία ή με ομοφωνία εφόλων των τομέων πολιτικής και πάλι στο Twitter account μπορείτε να ψηφίσετε ναι ή όχι, αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε δηλαδή. Στη συνέχεια θα πάρετε το βήμα. Θα σας ζητηθεί να μιλήσετε και να κάνετε τις παρεμβάσεις σας. Να σας υπενθυμίσω αγαπητοί συνάδελφοι ότι υπάρχουν κάμερες οι οποίες ακολουθούν τον ομιλητή αμέσως μόλις πατήσει το κουμπί του μικροφόνου του. Σας ζητώ λοιπόν, μόλις ακούσετε το όνομά σας, να σηκώνεστε από τη θέση σας, να πατάτε το κουμπί του μικροφόνου για να ζητηθεί το βήμα και η κάμερα θα εστιάσει αυτομάτως επάνω σας. Θα έχετε 60 δευτερόλεπτα να μιλήσετε. Στην οθόνη ε, θα υπάρχει και ένα χρονόμετρο που με φθήνοντα τρόπο θα μετρά τα λεπτά που ε, τα δευτερόλεπτα που σας μένουν ακόμα διαθέσιμα και ζητώ από όλους τους παρεμβαίνοντες να σέβονται το χρόνο αυτό. Αν ξεπεραστούν τα 60 δευτερόλεπτα θα αναγκαστώ να σας διακόψω δυστυχώς κλείνοντας το μικρόφωνο και αυτό βέβαια το καταλαβαίνετε και εσείς και εγώ κάθε άλλο παρά ευχάριστο είναι ε, απλά θα σας δώσει μια γεύση α, της αυτηρότητας που διέπει τις διαδικασίες μας, αλλά πρέπει όλοι όσοι έχουν ζητήσει το βήμα και είναι πάνω από 100 να μπορέσουν να παρέμβουν. Οπότε ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός. Τελευταίο και λιγότερο σημαντικό, τα... έχουμε ειδικό εκπρόσωπο διοργάνωσης, εκπρόσωπο των ε, ευρωπαϊκών ε, θεσμικών οργάνων ε, που θα μπορούσε να είναι από την Κομισιόν ή από το Κοινοβούλιο είναι ένα συμπεριογνώμων ο οποίος θα ρυθμίσει εδώ τα διαδικαστικά μας θα μας πει κάποια θέματα διαδικαστικά θα μιλήσετε εσείς, θα υπάρξει ψηφοφορία και στη συνέχεια θα υπάρξει και η παρέμβαση ατόμου που εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά όργανα που πραγματεύονται τα διάφορα θέματα και θα πάρει το βήμα ε, και πάλι είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλε και όσε ερωτήσει τεθούν από πλευρά σα με τη παρέμβασή σα και το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία θα καταγραφούν και θα γνωστοποιηθούν επισήμω κατά τη διάρκεια των τριών συνεδριών. Ε, θα είναι όλα αυτά κομμάτι μια προσπάθεια επιρροή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων επί τη βάση τη έκβαση τη ψηφοφορία. Και αυτό βέβαια είναι κάτι που ε, θα αναλάβουν το Euro Chambers ε, που θα αναλάβει τις επόμενους εβδομάδες ή μήνες. Νομίζω ότι με αυτά ε, ολοκληρώσαμε τα προκαταρκτικά. Ας κάνουμε τώρα μια δοκιμή του συστήματος ε, ψηφοφορίας. Έχετε όλοι σας ένα badge, μια καρτούλα. Αυτή η καρτούλα που θα τη δείχνω τώρα είναι και κάρτα ψηφοφορίας. Βγάζετε την κορδέλα, τοποθετείτε την καρτέλα μέσα στη σχισμή μπροστά στη συσκευή ψηφοφορίας που έχετε μπροστά σας και αμέσως ψηφίζετε. Μπορείτε να ψηφίσετε ναι εάν πατήσετε το πράσινο κουμπί, αν πατήσετε το κόκκινο είναι αρνητική ψήφος και για το κεντρικό άστρο κουμπί είναι οι αποχές. Να κάνουμε μια δοκιμή λοιπόν για να δούμε αν όλα δουλεύουν καλά. Παρακαλώ όλοι με τις κάρτες στο χέρι. Ας βάλουμε ένα ερώτημα, τυπικό ερώτημα έτσι για τη δοκιμή δοκιμαστικό ερώτημα και θα το διαβάσουμε στην οθόνη αν μπορέσουμε πώς ε, οι νέοι κανόνες ε, του απορρίτου των πληροφοριών για, που η Ευρώπη έχει θέσει σε εφαρμογή μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά ε, τις ε, επιχειρήσεις. Ναι ή όχι. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε. Ισχύει ή όχι αυτό. Θα είναι δυσκολότερο για τις επιχειρήσεις αυτό το νέο σύστημα. Η κάρτα στη σχισμή, πράσινο το ναι, κόκκινο το όχι και το λευκό οι αποχές είναι στο κέντρο. Συνεχίστε να ψηφίζετε παρακαλώ. Έχουμε ακόμα 100 άτομα που δεν έχουν ψηφίσει. Παρακαλώ κάντε το τώρα. Δοκιμαστική ψηφοφορία είναι, δεν είναι κάτι κακό. Με την κάρτα σας στη σχισμή παρακαλώ και μετά πατάτε πράσινο για ναι, κόκκινο για όχι, λευκό για την αποχή. Η ερώτηση είναι αν και κατά πόσο οι νέοι κανόνες ε, περί της προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη είχαν αρνητικό αποτέλεσμα στην επιχείρησή σας. Προτείνω να περαιωθεί η ψηφοφορία τώρα, θα την κηρύξουμε ως περαιωθήσα δηλαδή, οπότε για να δούμε τι έχει συμβεί. Παρακαλούμε να εμφανιστούν στην οθόνη τα αποτελέσματα. Βλέπετε εδώ, έχουμε ψηφίσαντες 566, ε, γύρω στους 100 δεν φέρεσαν να ψηφίσουν ή δεν ψήφισαν. Αποτέλεσματα 308 ναι, ότι δηλαδή υπήρχε αρνητικό, αρνητική επίπτωση και 202 είπαν όχι, 56 αποχές. Προτείνω τώρα στο μεταξύ και προκειμένου να ε, σας προκαλέσω λίγο να κάνουμε ακόμα ένα τεστ με την ψηφοφορία με τις τρεις ερωτήσεις οι οποίες έχουν τεφυγεί από ψηφοφορία έτσι και αλλιώς μέσω των μέσων κοινωνικής ε, δικτύωσης για να δούμε λίγο να πάρουμε μια γεύση για το τι αίσθηση επικρατεί εδώ ως προς τα ερωτήματα αυτά. Θα ήθελα να σας ζητήσω να ψηφίσετε και ταυτόχρονα ε, θα ζητούσα, αλλά δεν γίνεται, να εμφανιστούν οι ερωτήσεις στην οθόνη. Περιμένω ε, σήμα. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, το ερώτημα λοιπόν το πρώτο. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ένα ειδικό ταμείο ολοκλήρωσης για τις μικρομεσαίες που να δώσει ευκαιρίες για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Παρακαλούμε ψηφίστε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Περαιούται η ψηφοφορία εδώ. Τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν ευθύ αμέσω στην οθόνη. Έχουμε λοιπόν ψηφίζοντε 562, εκ των οποίων 429 απεφάθησαν καταφατικά, 93 αρνητικά και 40 απήχαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δεύτερο ερώτημα τώρα. Η ψηφοφορία στους κόλπους του Συμβουλίου θα πρέπει να γίνεται με πλειοψηφία ή, ε, ε, και όχι με ομοφωνία εφόλων των τομέων της πολιτικής. Ξεκινάει η ψηφοφορία λοιπόν.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 Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η ε, ψηφοφορία στο σημείο αυτό για να δούμε μαζί ποια είναι η έκβαση αυτής της ε, ψηφοφορίας. Ψήφισαν 571, εκ των οποίων 393 υπέρ, 128 κατά και 50 πήχαν. Ευχαριστώ πολύ. τελευταίο ερώτημα που θα τεθεί στην ψηφοφορία και ε, θα με ενδιέφερε να δω ποια θα είναι η τελική έκβαση όταν θα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα αυτά με αυτά που θα προκύψουν από την ψηφοφορία μέσω του ίντερνετ. Ε, πρώτη ψηφοφορία λοιπόν σχετικά με το εμπορικό ζήτημα. Σε μια εποχή κλιμακούμενων εμπορικών αντιπαραθέσεων και ενός επιτινόμενου εθνικισμού εντός και εκτός Ευρώπης έχετε τη διάθεση να παραμείνετε ενωμένοι πίσω από μια κοινή εμπορική ευρωπαϊκή πολιτική. Ψηφίστε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Περαιούται ε, εδώ η ψηφοφορία και επί του ερωτήματος αυτού για να δούμε από κοινού ποια είναι η έκβαση της ψηφοφορίας. Ψήφισαν 586, εκ των οποίων 565 απεφάθησαν θετικά και 10 μόνο αρνητικά. Προφανώς και είναι ενθαρρυντική αυτή η έκβαση ε, πριν του ότι το ακροτήριο εδώ πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική θα πρέπει να συνεχίσει να είναι κοινή και στο μέλλον. Στη συνέχεια θα δούμε και θα διατυπώσουμε σχόλια στην καταληκτήρια συνεδρία σχετικά με την ενδεχομένως αντιστήχηση των αποτελεσμάτων τη ψηφοφορία αυτού του ακροτηρίου με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την ψηφοφορία μέσω των ε, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ε, που θα προκύψουν από την ε, συμμετοχή στην διαδικασία πλήθους ανθρώπων μέσω του Twitter. Περιμένουμε τώρα να προσέλθει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναμένεται ανα πάσα στιγμή. Μου είπαν ότι θα έπρεπε ήδη να είναι εδώ. Δεν ξέρω αν είναι ήδη στο κτίριο αν θα έρθει από πίσω ή από μπροστά. Δεν ξέρουμε ακριβώς από ποια είσοδο της αίθουσης θα έρθει, αλλά θα το ανακαλύψουμε που θα πάει. Is coming. Yeah. Καταφθάνει λοιπόν. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ στενός φίλος της επιχειρηματικής κοινότητας καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του και είναι και φίλος των μικρομεσαίων ιδιαίτερος ε, Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ, στο κοινοβούλιο μας. Για αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός, την πολύ σημαντική εκδήλωση, επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη. Η επικεφαλής κύριος Αντρέα Ρούτσπα και ο βασικός ε, σύμβουλος της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, ε, ο πρόεδρος του Ευρωπημελητηρίου και ο κύριος Σαμπρουτσίνη, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήρθατε. στο, ε, στην πέμπτη κοινοβουλευτική συνέλευση των επιχειρήσεων. Είναι πολύ σημαντικό είναι πολύ σημαντική η εκδήλωση αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους επιχειρηματίες. Πρέπει να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρέπει να ενδυναμώσουμε την πραγματική μας οικονομία. Πρέπει να ενδυναμώσουμε τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες, τις μεγάλες όλες. Χωρίς εσάς είναι αδύνατον να καταπολεμήσουμε την ανεργία και κυρίως την ανεργία των νέων. Γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δέσμευσή σας, όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε μέρα. Η ανάπτυξη λοιπόν κατά της ε, ανεργίας υπέρ της Ευρώπης, που είναι μια βιομηχανική ήπειρος, έχουμε 24 εκατομμύρια εταιρείες. Η χώρα μου έχει 4 εκατομμύρια επιχειρήσεις. Ξέρετε, είναι σημαντικό για την οικονομία μας. Χωρίς την πραγματική οικονομία είναι αδύνατον να υπάρχει προστασία κατά τις διάφορες ε, κρίσεις που βιώνει η οικονομία σας, είστε ο πιο ε, σημαντικός στυλοβάτης. Όταν ήμουν αντιπρόεδρος της Κομισιόν και ε, επίτροπος για τη βιομηχανία, Πάντα υπολόγιζα στη βοήθειά σας να με βοηθάτε στην ε, αποστολή μου για την ανάπτυξη, οπουδήποτε στον κόσμο. Υπήρξατε και συνεχίζετε να αποτελείτε μια πολύ καλή εικόνα της πραγματικής ευρωπαϊκής οικονομίας. Η δουλειά σας είναι πολύ σημαντική και για μένα αλλά και για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τώρα επιτρέψτε μου να εκφραστώ στη μητρική μου γλώσσα, στα Ιταλικά. Φέτος η οργάνωσή σας εορτάζει την 60η επέτειο από την ίδρυσή της και πραγματικά έχει μια ιστορία πολύ στενά συνδεδεμένη με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι το 1958 το Ευρωεπιμελητήριο ήταν, μέσα στη, ήταν στη φάση της ε, ενσωμάτωσης και από τότε μέχρι σήμερα η συμβολή σας υπήρξε σημαντικότατη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Ευρωεπιμελητήριο ανέκαθεν με συνόδευε μου για την ανάπτυξη στην Ασία, στη Μέση Ανατολή, στην Αμερική και ανέκαθεν υπήρξε ε, η σημαία των ευρωπαϊκών εταιριών. Το Ευρωεπιμελητήριο Ε, είναι μια πραγματικότητα ε, που βασίζεται στην ευημερία, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει και απασχόληση, εργασία. Είναι και ένα εργαλείο για την ενδυνάμωση των διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός αυτής ε, και εκτός από αυτά που κάνετε και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, χωρί επιχειρήσει δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχει απασχόληση. Το 85% των ε, θέσεων εργασία εξαρτώνται από εσά και το, τα 2 τρίτα τη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα επίση εξαρτώνται από εσά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σα επαναλαμβάνω ότι χωρί τη δική σα βοήθεια δεν υπάρχει ανάπτυξη. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύπτει όλο και περισσότερο τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Όπως σας έλεγα λοιπόν, χωρίς τη δική σας πραγματικότητα, η οικονομική ε, κρίση θα είχε καταστρέψει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες οι οποίες δεν είχαν έτσι ένα ισχυρό δίκτυο μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι αυτές οι οποίες υπέφεραν τα μάλα κατά τη διάρκεια της ε, οικονομικής κρίσης από το 2008 μέχρι το 2012-2013. Ευτυχώς ε, όταν αναφερόμαστε στο 2008 βλέπουμε ότι είχαμε ε, ε, ε, αύξηση των εταιριών, αύξηση της προσθέμενης αξίας κατά 18%, αύξηση της απασχόλησης του κατά 3%. Δηλαδή γίνονται πράγματα και πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε πράγματα για να διατηρούμε την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεών μας. Όσον αφορά το σημαντικό έργο που κάναμε τα τελευταία χρόνια στην Κομισιόν, ε, πρέπει να το συνεχίσουμε, πρέπει να έχουμε μια βιομηχανική πολιτική και όταν μιλάω για τη βιομηχανία δεν αναφέρομαι στην ε, μεγάλη κλίμακα βιομηχανία, αλλά αναφέρομαι σε όλα όσα έχουν να κάνουν με την πραγματική οικονομία και αυτό μας ε, καθιστά ικανούς να αναπτύξουμε μια σειρά επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών. Γιατί αν δεν υπάρχει βιομηχανία, δεν ε, υπάρχουν και υπηρεσίες. Ε, δεν υπάρχουν εταιρείε ε, υπηρεσιών. Η ψηφιακή πολιτική, η ενεργειακή πολιτική, όλα τέλο πάντων, οι διεθνεί εμπορικέ πολιτικέ πρέπει να παρέχουν εγγυήσει στι επιχειρήσει μα και πρέπει να δίνουν καλύτερε συνθήκε για να μπορούν να ανταγωνίζονται σε διεθνέ επίπεδο. Η Ευρώπη, θα είμαι σαφή, έτσι, δέχεται επίθεση. που σπουδαίοι όλου του κόσμου αν έβλεπαν ε, τι, τι, γίνεται με την εσωτερική αγορά μας, με την ικανότητά μας ε, να φτιάχνουμε ε, προϊόντα. Δηλαδή δεν εξάγουμε μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκτός. Αν τα βλέπαν όλα αυτά καλύτερα, ε, θα καταλάβαιναν και για την ποιότητα των προϊόντων μας, που τα προϊόντα αυτά είναι ανώτερης ποιότητας. άρα όλα αυτά πρέπει να υποστηριχθούν όμως με καλές εμπορικές πολιτικές. Τώρα, πρέπει να ανταποκριθούμε και στα, στις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ανταγωνιστικότητα ή με τον ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για σκεφτείτε λίγο και το dumping και τις σχέσεις με την Κίνα, με τη ΣΥΠΑ, σκεφτείτε την κλιματική αλλαγή, την προστασία των καταναλωτών και επίσης την πνευματική ιδιοκτησία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες έτσι ώστε να εκφράζετε καλύτερα την αριστεία και τις δυνατότητές σας. Πολλοί από εσάς έχετε ήδη πειραματιστεί και έχετε βιώσει τα ωφέλη της εσωτερικής αγοράς. Έχουμε 1.700 περιφερειακ... 1.700 περιφερειακά και τοπικά εμπορικά επιμελητηρία και ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζεστε δείχνει πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ε, ευημερία και ευμάρεια. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ίσως ε, ισότιμος ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει περισσότερη ε, οικονομική εναρμόνιση ε, πρέπει να αποφύγουμε τους φορολογικούς ε, παραδείσους, να τους ξεφορτωθούμε. Ε, δεν μπορεί, ας πούμε, εσείς να πληρώνετε περισσότερους φόρους από ότι κάποιες εταιρείες που δεν δημιουργούν καλύτερη ευημερία στην Ήπειρό μας και βγάζουν και δίνουν όλα τους τα κέρδη στην Κίνα. Όλες οι εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται και οι ευρωπαϊκές εταιρείες. Εντάξει, όταν δημιουργείς ευημερία πρέπει να πληρώνεις φόρους. Η ενεργειακή αγορά πρέπει να υποστηρίξει την ανάπτυξη επιχειρήσεων και αυτό που χρειαζόμαστε είναι επενδύσεις, όχι βοήθεια, όχι συνδρομή και κρατικές ενισχύσεις. Όταν μιλάμε για τα χαμηλότερα επίπεδα της ε, κρίσης, αυτά, πρέπει να, βγήκαμε από αυτά και πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη φάση της ε, ανάκαμψης, διότι αντιμετωπίζουμε άλλα διαφορετικά ε, ζητήματα. Έχουμε, ας πούμε, το σχέδιο ε, επενδύσεων Juncker, το οποίο είχε πολύ καλό αντίκτυπο και συνέπειες. Έχουμε περισσότερες επενδύσεις στον επικείμενο προϋπολογισμό. Τίποτα από αυτά όμως δεν θα είναι αρκετό από μόνο του. Τα κράτη, οι μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να δεσμευτούν προς αυτή την κατεύθυνση ότι οι επιχειρηματίες χρειάζονται κεφάλαιο. Είμαστε... Έχουμε την υποχρέωση να ολοκληρώσουμε και την τραπεζική αγορά έτσι ώστε να μπορέσουμε να, χρηματοδοτήσουμε, να χρηματοδοτούμε πιο εύκολα ε, την καινοτομία και τις νέες επιχειρήσεις. Ε, πρέπει να δώσουμε πίστη στις επιχειρήσεις και πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στις τράπεζες να δίνουν ε, δάνεια μέχρι και 1,5 εκατομμύριο ευρώ έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερη ρευστότητα, να έχουν ρευστό οι μικρομεσαίες. Αυτό είναι το μήνυμα της εμπιστοσύνης που ε, θέλουμε να το ανανεώσουμε. Έστω και αν υπάρχει κάποια αντίσταση, θέλουμε να αυξήσουμε, αν θέλετε, το, το κατόφλι στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ανέκαθεν εγκρίναμε μέτρα τα οποία ευνοούν ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ας πούμε η επανεξέταση του τραπεζικού πακέτου είναι ένα παράδειγμα. Και τώρα αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η δέσμευση των κρατών μελών, διότι σε ορισμένες χώρες η φορολόγηση είναι υψηλότατη και υπάρχουν καθυστερήσεις ε, ε, από διοικήσεις ε, τεράστιες καθυστερήσεις που προκαλούν, είναι, προκαλούν ε, το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων. Γι' αυτό λοιπόν η συγκεκριμένη οδηγία όσον αφορά την πληρωμή των καθυστερούμενων αποτελεί εγγύηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι θα υπάρχουν, υπάρχει μια δημόσια διοίκηση που ε, θα σέβεται και τις δικές της υποχρεώσεις και δεν θα είναι αυστηρή μόνο με τους πολίτες. Και το λέω αυτό στις αρχές της δικής μου χώρας επίσης. Γιατί εντάξει, όταν πρέπει να πληρώσουν ε, εταιρείε, το κράτο δηλαδή, είναι ο χειρότερο, είναι πολύ κακοπληρωτέ. Η Ιταλία ε, έλαβε έτσι ευελιξία στον προπολογισμό της ε, έτσι ώστε το, το, κράτος να καταβάλει τα χρωστούμενα στις εταιρείε, αλλά η ευελιξία αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε με τον σωστό τρόπο. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η χώρα μου, η Ιταλία, έπρεπε να λειτουργήσει σωστά, αλλά και άλλες χώρες που καθυστερούν χρήματα στις εταιρείες πρέπει να ακολουθήσουν αναλόγως. Το, επίσης χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις και για την έρευνα. Ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα φροντίσει να αφιερωθούν περισσότερα κονδύλια στον τομέα αυτών. Έχουμε 120 εκατομμύρια λίγο πολύ για επενδύσεις και έρευνα. Ε, πρέπει να εδραιώσουμε την ηγετική μας θέση στις επιστήμες και στην τεχνολογία. Τα προγράμματα έρευνας είναι πάρα πολύ καλά, είναι επιτυχημένα εδώ και 30 χρόνια, αλλά πρέπει να τα συνεχίσουμε και γι' αυτό στις 27 Νοεμβρίου θα φιλοξενήσω μία διάσκεψη για την Ευρωπαϊκή Έρευνα Θέλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες μας πόσο βελτιώθηκαν οι ζωές μας χάρη στην έρευνα που χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την ε, ικανότητα να φροντίσουμε ώστε ο κόσμος της έρευνας και των επιχειρήσεων συνεννοούνται και συνομιλούν μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε καταστάσεις ε, κατά τις οποίες υπάρχει απώλεια των ε, καλύτερων νεαρών ερευνητών γιατί μπορεί, πάντα ε, βρίσκουν ε, δουλειά στο εξωτερικό, στον Καναδά ή στη ΣΥΠΑ, στην, στο Ισραήλ και την Ιαπωνία γιατί δεν μπορούν να καλυφθούν από, εμάς. Είναι μια πραγματική πολιτική αυτό που πραγματικά δημιουργεί δεσμούς μεταξύ νέων επιστημόνων και και, και, έρευνας. Αυτοί οι νέοι εγγυώνται το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Ανυπομονώ λοιπόν να δω ε, τη δική σας σύμβολη και θέλω να καλέσω τώρα τους επικεφαλείς του Ευρωεπιμελητηρίου και σας όλους που μπορείτε να που μπορείτε να έρθετε και να συμμετάσχετε στις 27 Νοεμβρίου στη διάσκεψη γιατί η σχέση μεταξύ έρευνας και επιχειρήσεων είναι σημαντική. Δεν μπορούμε να ε, δουλεύουμε ξεχωριστά. Πρέπει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργάζονται γιατί το ένα είναι αναπόσπαστο τμήμα του άλλου. Και καθημερινά αντιμετωπίζετε τις αγορές. Ξέρετε πολύ καλά πόσο σημαντικές είναι οι δεξιότητες έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Δυσκολεύεστε να βρίσκεστε ειδικευμένους καταρτισμένους εργαζόμενους που ε, ε, καλύπτουν τις ανάγκες σας και έτσι ερχόμαστε στο θέμα της κατάρτισης. Δεν μπορούμε να έχουμε νέους ανέργους στις εταιρείε μας οι οποίοι δεν έχουν ε, πρόσβαση σε δεξιότητες. Έχουμε μία συνάντηση για την προσφορά και τη ζήτηση και εγώ Μοιράζομαι βεβαίως την ιδέα του εράσμου για τους νέους επιχειρηματίες και του Europass και του Eures. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ε, ε, λέει ότι 56 εκατομμύρια άνθρωποι θα κάνουν δουλειές που τώρα δεν υπάρχουν. Το 33% των Ευρωπαίων εργαζομένων έχουν βιώσει κάποιες τεχνολογικές αλλαγές που άλλαξαν τη ζωή τους. Κάποιος ξεκινά να δουλεύει με τον άλφα τρόπο και μετά αυτός ο τρόπος αλλάζει. Θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση ε, για την κατάρτιση, την εκπαίδευση και δεν θέλουμε κανείς να μείνει πίσω. Η διαβίου κατάρτιση είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους τους ανθρώπους και για τις επιχειρήσεις όμως. Θα πρέπει όλοι να ε, συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. η κοινωνική οικονομία της αγοράς μπορεί να οδηγήσει σε ε, ευημερία. Η Ευρώπη είναι γνωστή για τη δημιουργικότητά της και για τα προϊόντα της παγκοσμίω, για την ποιότητά του συγκεκριμένα. 30 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη εξαρτώνται από τις εξαγωγές. Είχαμε το ότι συνεργασία με, το, με τη Σιγκαπούρη, τον ε, Καναδά και θέλουμε και άλλες συμφωνίες. Χιλή, Μερκοσούρα, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τις εταιρείες, κυρίως τις μικρότερες εξ αυτών, να μπορούν να εξάγουν περισσότερο, να τις περασπιστούμε ε, κατά του αθέμητου ανταγωνισμού, να προστατεύουμε ε, τα τα, τα, σήματά τους, να προστατεύουμε το περιβάλλον. Ε, θέλουμε ελεύθερο εμπόριο με σαφείς κανόνες και με ε, δίκες συνθήκες. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αγωνιστεί ε, για τους κανόνες αντι-dumping κατά της Κίνας και άλλων χωρών οι οποίες πράγματι κάνουν dumping σε πολλούς τομείς. Δεν μπορούμε δηλαδή να, δεχτούμε ότι υπάρχει το, το δικό τους θέμα το, του πλεονάσματος πέφτει στους δικούς μας όμως ε, και μας βαρύνει. Μέτρα λοιπόν αντι-dumping και το κοινοβούλιο ε, έχει αγωνιστεί για όλα αυτά, παρόλο που αντιμετωπίζει και αντίδραση και αντίσταση από τα κράτη-μέλη και από την Κομισιόν. Εν κατακλείδη, χρειαζόμαστε μια Ευρώπη η οποία ε, θα αποτελεί όλο και περισσότερο φύλλο στενό των επιχειρήσεων. Η νομοθεσία πρέπει να απλοποιηθεί και να γίνει λιγότερο γραφειοκρατική. Πρέπει να δούμε λιγάκι τον εαυτό μας, να κάνουμε μια ενδοσκόπηση και να έχουμε περισσότερους πόρους ε, για τις εταιρείες και τις ε, μικρομεσαίες και τις καινούριες. Έχουμε ευρωεκλογέ σε λίγους μήνες. Εξετάζουμε τις τάσεις που επικρατούν. Βλέπουμε πως κάποιοι απορρίπτουν. Εγώ είμαι περήφανος που είμαι Ιταλός. Η Ιταλία είναι το σπίτι μου. Αλλά επειδή είμαι Ιταλός, αισθάνομαι και Ευρωπαίος. Εγώ γεννήθηκα στη Ρώμη. Και βεβαίως αισθάνομαι Ευρωπαίος. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης υπάρχουν πράγματα τα οποία μου υπενθυμίζουν την πόλη μου. Σε όλη την Ευρώπη. Χάρη στην εξαίρετη δουλειά ε, των νομικών ε, εμπειρογνωμών από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Το δικό μας δίκαιο ε, διέπει τις καθημερινές μας λειτουργίες. Και αυτό το οφείλουμε στους νομικούς ιστορικούς της Γερμανίας και της Γαλλίας. Άρα το να είσαι πατριώτης σημαίνει ταυτόχρονα ότι είσαι και Ευρωπαίος. Αν είσαι καλός Ευρωπαίος, είσαι και Ιταλός, είσαι και Γάλλος, είσαι και απ' όλα. Δεν θα χρειάζεται να ψάχνουμε εξυλαστήρια θύματα. Αυτοί οι οποίοι βασίζονται πάρα πολύ έτσι στην... Ε, ε, ε, στην εθνική κυριαρχία. Αυτοί ψάχνουν τα εξηλαστήρια θύματα. Αλλά εγώ δεν χρειάζομαι κάτι άλλο, δεν χρειάζομαι άλλο σήμα από αυτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω και αν είμαι Ιταλό. Ε, δεν θα πρέπει να κατηγορούμε την Ευρώπη για τα πάντα. Σαφώ και πρέπει να αλλάξει, σαφώ και πρέπει να βελτιωθεί, ε, να έχει λιγότερη γραφειοκρατία, να εφαρμόσει καλύτερε πολιτικέ, να υπάρχουν πολιτικοί ε, συνομιλητές οι οποίοι θα μπορούν να υιοθετούν πολιτικές που οδηγούν την Ευρώπη σωστή κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε πολιτικές και εσείς χρειάζεστε πολιτικές που θα δίνουν συγκεκριμένες απαντήσεις ε, στις ε, ανάγκες σας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Πρέπει εσείς είστε αυτοί. Πρέπει να σας υποστηρίξουμε γιατί χωρίς εσάς δεν υπηρετούμε του ανθρώπου τη Ευρώπη, του Ευρωπαίου πολίτε. Έχετε ένα θεμελιώδη ρόλο στην κοινωνία μα, γιατί χωρί δουλειά δεν υπάρχει αξιοπρέπεια. Χωρί δουλειά χάνεται την αξιοπρέπεια, χάνει ο κόσμο την αξιοπρέπειά του. Άρα λοιπόν, όταν χάνει την αξιοπρέπειά σου, χάνει και την ελευθερία σου. Και εσεί, επειδή δημιουργείτε θέσει εργασία, είστε υποδείγματα αξιοπρέπεια και ελευθερία. και γι' αυτό εδώ και χρόνια έχω δεσμευτεί να υποστηρίζω το έργο σας και το κάνω με πλήρη συνέστηση και με ζήλο γιατί θεωρώ ότι είναι το σωστό που να σας βοηθάμε να κάνετε αυτό που κάνετε και να καταστήσουμε την Ευρώπη μια ελεύθερη ε, πλούσια ήπειρο όπου ο καθένας, ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα έχει το δικαίωμα να αναπτύσσεται. Και χωρίς επιχειρήσεις αυτό δεν μπορεί να γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. καλώ ορίσατε και σας εύχομαι καλές εργασίες σήμερα. Now after these inspiring Μετά από αυτά τα λόγια γεμάτα έμπνευση, με χαρά ε, κυρίζω την έναρξη της ε, πρώτης ε, συνεδρίας. Θέλω να καλέσω δύο εκπροσώπους, τη Μαρτίνα Λαμπαγιώβα και το Μπράντο Μπενιφέρη, uh, an Ωραία. Ε, θέλω να σας παρουσιάσω ένα βίντεο ως εισαγωγή, το οποίο θα μας ε, δώσει έτσι λίγη τροφή για σκέψη όσον αφορά το θέμα συζήτησης ε, σε αυτή τη συνεδρία. Τώρα, ο λόγος στη Μαρτίνα Νταμπλαγιόβα με μία πρόταση. Χωρίς δεξιότητες, game over. Τελείωσε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι δύσκολο να παίρνει κανείς το λόγο μετά από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου. Θα προσπαθήσω να μιλήσω αγγλικά, γιατί μόνο στα ιταλικά θα μπορούσα να είμαι τόσο συναισθηματική, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ και με τα αγγλικά. Είμαι η Μαρτίνα ε, Ντλαμπατζόβα, είμαι μέλος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το, Ευρωπα... το Ευρωεπιμελητήριο με καλεί πάντα στην εκδήλωσή του και χαίρομαι ιδιαίτερα. Είναι πολύ χρήσιμο και για μένα και για σας. Είναι καλό να βρισκόμαστε μαζί στην Ολομέλεια εδώ στο ημικύκλιο και ξέρετε πριν από πέντε χρόνια θα καθόμουν εκεί μπροστά. Γιατί πριν έρθω στο κοινοβούλιο ήμουν επιχειρηματίας και θα ε, καθόμουν στη θέση σας εκεί και θα άκουγα κάποιους βαρετούς πολιτικούς, αλλά τώρα οι κανόνες έχουν αλλάξει. Αισθάνομαι ακόμη περισσότερο επιχειρηματίας παρά μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιο πολύ δηλαδή ε, στη δουλειά παρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο και για σας. Όμως, θεωρώ ότι όταν το Ευρωεπιμελητήριο σταματήσει να με καλεί εδώ, θα, θα σταματήσω να είμαι επιχειρηματέ και θα γίνω μόνο πολιτικό. Ελπίζω να, να μην συμβεί ποτέ αυτό. Ξέρετε, οι δεξιότητε και το τέριασμά τους με την απασχόληση, με την ανεργία των νέων. Όλα αυτά είναι θέματα που με έχουν απασχολήσει πολύ ε, πριν γίνω μέλος του Ευρωκοινοβουλίου και τώρα περισσότερο από ποτέ συνειδητοποιώ ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι ένας κόσμος γρήγορων αλλαγών. Χαρακτηριζόμαστε από την ψηφιοποίηση, την παγκοσμιοποίηση, τη διασύνδεση, τους νέους τρόπους εργασίας, των νέων τύπων εργασιακών συμβάσεων. Δεξιότητες που διδάσκουμε στα σχολεία σήμερα μπορεί αύριο να μην υφίστανται. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα και τι μπορούμε να αλλάξουμε. Πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι ε, ριζωμένο στο τρέχον εκπαιδευτικό ε, πρόγραμμά μας και πρέπει και στην εκπαίδευση να έχουμε κοινωνική ευθύνη όπως έχουν οι επιχειρήσεις, ε, οι εταιρείε. Πρέπει να βοηθήσουμε τα, τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα να μην έχουν πρόβλημα να προσαρμόζονται στην, στις ανάγκες της σημερινής και μελλοντικής αγοράς εργασίας. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι κάποια σχολεία δεν μπορούν να προσφέρουν τι απαραίτητε δεξιότητε στου νέου ανθρώπου, έτσι ώστε ε, να αντιμετωπίσουν του μελλοντικού εργοδότες του. Άρα εσεί, ω εργοδότε, πρέπει να του βοηθήσετε να προσφέρουν τις σωστές δεξιότητες ε, στου νέου ανθρώπου. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά καλά παραδείγματα στην Ευρώπη, εξαιρετικά παραδείγματα συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, κυρίως ε, σε κάποια κράτη-μέλη έχουν πολλά καλά παραδείγματα, ωστόσο δεν υπάρχει ένα σύστημα, δεν υπάρχει μια συστηματικότητα, λείπει από την Ευρώπη. Ε, σήμερα ε, ε, έχουμε διαπιστώσει ότι 40% των επιχειρήσεων αγωνίζονται να βρουν καταρτισμένο προσωπικό. Ενώ 40%, 40 των νέων ανθρώπων δουλεύουν σε διαφορετικό τομέα από αυτόν για τον οποίο σπούδασαν. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια στρέβλωση. Το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων είναι ακόμη πιο ανησυχητικό, διότι άτομα 18 με 25 στην Ευρώπη ε, μαστίζονται από την ανεργία. Σε κάποια κράτη-μέλη έχουμε και 50% ανεργία. Σε κάποιες περιφέρειες, κυρίως στην Νότια Ευρώπη, αυτό το ποσοστό αγγίζει και το 60%. Και αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερος. Ξέρουμε ότι υπάρχουν νέες τάσεις όσον αφορά δεξιότητες κλειδιά που απαιτούνται, ε, ζητούνται όλο και περισσότερες έτσι, χειρονακτικές δεξιότητες και ε, αναλυτική σκέψη, καινοτομία, δημιουργικότητα, ε, στρατηγικές ε, ενεργούς εκμάθησης. Υπάρχει και αύξηση όσον αφορά τα λεγόμενα soft skills, τι απαλέ δεξιότητε. Και πάντα γελάω αυτό. Γιατί τι λέμε έτσι. Αυτέ είναι πιο δύσκολε να αποκτήσει κανεί. Ε, δεν είναι έτσι πολύ απαλέ και εύκολε. Ε, σύμφωνα με τον Όσα, το 19% των ε, θέσεων εργασίας θα εξαφανιστεί εντελώς εξαιτία της ε, ρομποτικής ε, και της ψηφιοποίησης. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη σας από αυτό, διότι γνωρίζουμε ότι θα αλλάξουν οι δουλειές, θα αλλάξουν τα επαγγέλματα, θα προκύψουν νέα επαγγέλματα και ο κόσμος θα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτος, θα πρέπει να υπάρχει μια προσαρμοστικότητα όσον αφορά την επαγγελματική καριέρα. Όλες αυτές είναι σημαντικές αλλαγές και δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Πρέπει να σκεφτούμε και να προνοήσουμε, να προετοιμάσουμε και το εργατικό δυναμικό και την αγορά εργασίας για αυτές τις αλλαγές, γιατί οι αλλαγές επίκειται και θα εξαρτάται από εμά αν θα είναι καλές ή κακές. Οι εργοδότε στην Ευρώπη υλοποιούν, εφαρμόζουν διαφορετικές ε, πρακτικές προτιμούν να προσλαμβάνουν νέο μόνιμο προσωπικό αντί να επενδύουν στην επανακατάρτιση του τρέχοντος προσωπικού. Άλλοι προτιμούν τον εξοπορισμό. Υπάρχουν σίγουρα διαφορετικές προσεγγίσεις και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε για τις δικές σας καλές πρακτικές, γι' αυτό είσαστε και εδώ ε, να εξετάσουμε όλες τις στρατηγικές και τον καλύτερο δυνατό τρόπο συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, θεσμών και πανεπιστημίων. Κάθε φορά που συζητώ, που μιλώ με επιχειρηματίες, κάθε φορά το μείζον ζήτημα και το μείζον πρόβλημα είναι το θέμα των ε, δεξιοτήτων και η προσαρμογή για τη μελλοντική αγορά εργασίας. Είναι ένα θέμα που το συζητάμε διαρκώς με τους επιχειρηματίες. Πιστεύω λοιπόν ότι ο τρόπος με τον οποίο ανταλλάσσουμε ευέλτιστες πρακτικές, δηλαδή μαζί σας, σίγουρα είναι σημαντικό για όλους προκειμένου να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές και πρέπει αυτές τις αλλαγές να τις μετατρέψουμε σε ευκαιρία. Όπως σας είπα, μία λύση θα ήταν να μεταρρυθμίσουμε τα τρέχοντα εκπαιδευτικά συστήματα. Ξεκίνησαμε αυτή την ιδέα ήδη από πριν από τρία χρόνια να ξεκινήσουμε ένα είδος κοινωνικής εταιρική ευθύνη για τα σχολεία και τα, τα, εκπαιδευτικά ιδρύματα. Γιατί οι επιχειρήσεις θα πρέπει ε, να ε, είναι κοινωνικά υπεύθυνε. τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα σχολεία θα πρέπει επίση να είναι υπεύθυνα. Γιατί είναι υπεύθυνα αυτά τα ιδρύματα για τι δεξιότητε που προσφέρουν στι νέε γενιέ και στου ε, μελλοντικού εργαζόμενου. Το τελευταίο σημείο μου αφορά την ε, εκπαίδευση περί επιχειρηματικότητας. Δηλαδή, αν δεν μιλήσουμε εδώ για επιχειρηματικότητα και για εκπαίδευση σχετικά, ε, μαζί με εσάς, πού θα μιλήσουμε. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα γίνουν επιχειρηματίες και θα ανοίξουν επιχειρήσεις. Απλώς πρέπει ο καθένας να γίνει καινοτόμος, να λύνει προβλήματα, να σκέφτεται ελεύθερα, να παίρνει ρίσκα. Η επιχειρηματικότητα είναι και μια στάση ζωής. Πώς να είσαι δραστήριο στη ζωή. Αυτό ε, είναι κάτι που πρέπει να το προωθήσουμε και στα σχολεία μας. Φυσικά, εδώ βρισκόμαστε σε μια ομάδα ανθρώπων που προσπαθεί και συνήθως πετυχαίνει και σκέφτεται έτσι εκτός, έξω από κουτάκια. Δηλαδή δεν ακολουθεί την πεπατημένη. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο να κάνουμε πράγματα. Μοιραστείτε λοιπόν τις ιδέες σας μαζί μας και σας υπόσχομαι ότι έχουμε έρθει εδώ να σας ακούσουμε. Ξέρετε, η πρώτη μου εκδήλωση ως πολιτικός μέλος του Ευρωκοινοβουλίου πριν από τέσσερα χρόνια ε, ήταν με ανθρώπους από τις επιχειρήσεις. Το 2014 εδώ στις Βρυξέλλες ε, ανέβηκα στο βήμα να μιλήσω και ο, πολύ, ξέρετε, εγώ επιχειρηματίας τώρα πήρα το λόγο να βγάλω λόγο, πετάχτηκα στην πολιτική και πρέπει να, αναφερθώ, να, να απευθυνθώ σε επιχειρηματίες. Τους είπα λοιπόν σε όλους, λέω, τι θέλετε να, να από μένα, τι θέλετε από μένα. Πώς ένας πολιτικός μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, ξέρετε τι μου απάντησαν. Με κοίταξαν και μου είπανε μην κάνεις τίποτα, απλά άκουσέ μας. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εδώ μέσα, εδώ που καθόμαστε και που ψηφίζουμε στις Ολομέλειες, υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί οι οποίοι πραγματικά είναι πρόθυμοι να σας ακούσουν. Άρα μην τα παρατάτε. Συνεχίστε να μιλάτε στους πολιτικούς ηθήνοντες. μοιράζεστε τις ιδέες σας μαζί ε, Του Είναι εδώ για να σα ακούσουν. Σα ευχαριστώ πολύ και σα εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σα. Ευχαριστώ πολύ Μαρτίνα Ντορπαγιώβα. Τώρα, σειρά σα να διατυπώσετε σχόλια, να επιβάλλετε ερωτήσει να διατυπώσετε ε, παρατηρήσει. Ε, πολλοί είναι αυτοί που έχουν ζητήσει το λόγο. Θυμηθείτε 60 δευτερόλεπτα ο καθένα και μετά υποχρεωμένο να κλείσω το μικρόφωνο. Πρώτο από τη Γερμανία, αριθμό 150, κύριο Έρικ Σβάιτσα. Die Alba-Gruppe ist ein führendes europäisches Umweltdienstleistungs- und Recyclingunternehmen, unter anderem neben Europa auch in Asien tätig. Um unsere Tätigkeit, unser Unternehmertum aus. Εξάλλου δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στην Ασία. Για να μπορέσουν λοιπόν να προχωρήσουμε με τις δραστηριότητές μας, μας χρειάζονται εργατικά χέρια ικανά και εκπαιδευμένα. Ξέρετε ότι ήδη ασχολούμαστε με την εκπαίδευση του προσωπικού μας. Μια ε, σωστή επαγγελματική εκπαίδευση ανοίγει μεγάλες προοπτικές σταδιοδρομίες στους νέους, αντιμετωπίζουν επιτυχημένα τον κίνδυνο της ανεργίας που μηδενίζεται και μάλιστα στελεχωνόμαστε και από άτομα από το Πανεπιστήμιο. 30% των φοιτητών νέων τέλο πάντων που ξεκινούν μελέτε στη ε, σπουδές στη Γερμανία όμω τι εγκαταλείπουν. 40.000 άτομα ε, τον χρόνο στη Γερμανία εγκαταλείπουν τι σπουδέ του. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις τη δική τελικά χάνουν την προοπτική να προσλάβουν ειδικευμένου πολύ πολύ ικανούς επαγγελματίε. Μια σωστή επαγγελματική κατάρτιση θα πρέπει ε, έτσι να εντάσσεται στο, σε ένα ολοκληρωμένο, πραγματικά ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρώπης ε, πρέπει να αναγνωριστούν τα προνόμια αυτή τη προσέγγιση. Το Erasmus ε, καταβάλει προσπάθεια προ την κατεύθυνση αυτή, αλλά πρέπει και η Κομισιόν να λαμβάνει υπόψη τη πιο σοβαρά και περισσότερο τα συμφέροντα και τι επιδιώξει των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Ελλάδα στη συνέχεια, θέση 221. Ο κύριο Πλάτων Μαλαφέκα, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που είμαι σήμερα εδώ μαζί σα. Το όνομά μου είναι Πλάτανος Μαρλαφέκα, είμαι ιδιοκτήτη εταιρεία Lux, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία αναψυκτικών στην Ελλάδα. 180.000 απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα για να αναζητούν και να ζητούν εργασία σε άλλε χώρε τα τελευταία 8 χρόνια τη κρίση. Οι έρευνε δείχνουν ότι μέχρι και το 76% των εφήβων εξετάζουν το ενδεχόμενο ε, να σπουδάσουν και να εργαστούν στο εξωτερικό σε άλλες χώρες. Ενώ στις μεταπολεμικές δεκαετίες είχαμε μαζική μετανάστευση από την Ελλάδα, ε, η σημερινή κατάσταση είναι τελείως διαφορετική επειδή πρόκειται για μια πραγματική ποιοτική αποστράγγιση. Είναι νέοι και οι πιο εκπαιδευμένοι άνθρωποι με νέες δεξιότητες που χρειάζονται και για την τέταρτη τεχνολογική επανάσταση αυτοί λοιπόν εγκαταλείπουν την ελλάδα προ όφελο άλλων χωρών παραδείγματο χάρη ηνωμένο βασίλειο γερμανία και άλλε που δεν έχουν πληρώσει ούτε ένα ευρώ για την εκπαίδευσή του. η διαρροή εγκεφάλων έχει τεράστιε αρνητικέ επιπτώσει στην ελληνική οικονομία. ποια μέτρα στοχεύουν να πάρει η ευρωπαϊκή ένωση για να ανατρέψει την τάση αυτή στην ελλάδα αλλά και σε άλλε χώρε όπω ακούσαμε που παρατηρεί το ίδιο φαινόμενο. ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με το Βέλγιο. Αριθμός 10. Κριστιαν Duro. Γεια σας. Η εξέβραση ε, ειδικευμένου και ικανού προσωπικού δεν είναι εύκολο πράγμα. Ε, το να τους προσλάβουμε και να τους εκπαιδεύσουμε σωστά είναι ακόμα πιο δύσκολο. 10% μόνο των ατόμων αυτών τελικά θα μπορέσουν να έχουν μια καλή έκβαση. Πρέπει να υπάρχουν σίγουρα και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην όλη διαδικασία και για μένα η γλώσσα είναι ένας από αυτούς τους παράγοντες. Η γλώσσα έχει σημασία όχι μόνο για, το, για την εργασία και την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο. Καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες και βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα που έχει δρομολογήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό και συγκεκριμένα για μια σωστή εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων στους, ε, σε επίπεδο των επιχειρήσεων. Θα μπορούσε ίσως η Ευρώπη να κάνει ακόμα περισσότερο ε, πέρα από αυτά που ήδη καταβάλλονται ως προσπάθειες στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε την Αυστρία. Φέση 5 Μάρτα Σούλτς. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αγαπητοί αντιπρόσωποι κυρίε και κύριοι, είμαι επιχειρηματία από την Αυστρία. Ε, δραστηριοποιούμε στον χώρο του τουρισμού και των υπηρεσιών γενικότερα. 800 είναι οι εργαζόμενοι ε, στο δυναμικό μας Είμαι επίσης πρόεδρος της ε, Επιτροπής Skills δεξιοτήτων του Eurochambers. Δεν με εκπλήσει το ότι το θέμα των ικανοτήτων και προσόντων είναι υψηλά στην ατζέντα μας σήμερα. Το βλέπουμε άλλωστε ότι από, την τον οικονομικό απολογισμό και μόνο η έλλειψη των ικανοτήτων είναι η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Αυστρία, τη χώρα μου, αυτή είναι μια από τι πιο μεγάλε προκλήσει που αντιμετωπίζουμε έτσι κι αλλιώ. Στους κόρπους της Επιτροπής μας στους Euro συζητούμε με τους ειδήμονες, ιδίω ε, και με το δίκτυο των ε, εμπορικών επιμελητήριων. Μιλούμε για τις εξελίξεις και τις ενδεχόμενες προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην κάλυψη αυτού του κενού σε δεξιότητες. Έχουμε έλλειψη σε αυτές. Προσπαθούμε να βρούμε τις καλύτερες πρακτικές και να τις αξιοποιήσουμε παντού όπου είναι αυτές διαθέσιμες στην Ευρώπη. Όπου υπάρχει τέτοια πρόκληση, βλέπουμε ότι υπάρχουν μέτρα που προσανατολίζονται προ την αγορά εργασία μέσω των διαφόρων συστημάτων επαγγελματική κατάρτιση και ιδίω τη ε, πρακτική εκμάθηση. Κατάρτιση επιτόπου στον χώρο εργασία, δουλεύοντα, χάρη στην οποία προσέγγιση οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ε, δεξιότητε ε, που χρειάζεται η επιχείρηση. Είναι λοιπόν η μαθητεία μεγάλη, πολύ σημαντικό κομμάτι ε, στη Βουδαπέστη θα έχουμε μια διάσκεψη για το θέμα αυτό, αλλά ο τομέα αυτό ε, των ε, δεξιοτήτων και προσόντων ε, θα μα απασχολήσει και στη Βιέννη τη διάσκεψη τις επόμενες εβδομάδε. Ελπίζω να συνεχίσουμε την προσπάθεια εξέβραση λύσεων και ότι θα μπορέσουμε πραγματικά να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στο μέλλον χάρη και σε αυτήν την εκδήλωση που η Αυστρία ετοιμάζει. Ευχαριστώ πολύ. Σα υπενθυμίζω ότι 60 δευτερόλεπτα αυστηρά έχει ο καθένας. Λουξεμβούργο στη συνέχεια θέση 452 Στάνι Βερικόφσκι. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρήσουν ή και να ανακτούν τι δεξιότητες και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να συνεργάζονται με το οικονομικό περιβαλλον προκειμένου να υπάρχει ικανή πρόθεση της εκμάθησης των τεχνολογικών αντιλήψεων πέρα ακόμα και από το προϊόν. Αυτές οι γνώσεις περνούν και από την μαθητεία επί της ε, γλώσσας, προγραμματισμού. Αυτές οι δεξιότητες επιτρέπουν ε, και τη δημιουργία και την επικύρωση λογισμικών που ανά την Ευρώπη μπορούν να αναπτυχθούν επί τη βάση ανοιχτών πηγών που θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν από όλε τι διαδικασίε που μα ε, απασχολούν έτσι κι αλλιώ. Η αυτονομία των πολιτών και του οικονομικού κόσμου περνάει από τον έλεγχο των χρησιμοποιούμενων λογισμικών και τα καλύτερα εχέγγυα για τον έλεγχο αυτό παρέχονται μέσα από την αξιοποίηση λογισμικών, ο κωδικός πηγής των οποίων είναι ανοιχτό σε όλους. Καλό θα ήταν να ενθαρρυνθεί η εκμάθηση και η αξιοποίηση αυτών των ανοιχτών ελεύθερων λογισμικών και να παροτρινθούν οι επιχειρήσει αλλά και η δημόσια διοίκηση να ζητούν τέτοιε λύσει και να τι απαιτούν προκειμένου για τις προκηρύξεις ε, εκδήλωση ενδιαφέροντο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με την Ιταλία. 2.32 Κλάου Αλτζέρι. Κλάους Αλτζιέρη, Ατζέρτη από την Κοζέντσα, από το εμπορικό επιμελητήριο συγκεκριμένα. Είναι έτοιμη άραγε η Ευρώπη να ανταποκριθεί στην πρόκληση της αγοράς εργασίας, να κυβερνούμε και να ζητούμε την ε, αλλαγή δεν αρκεί. Ε, πρέπει το, το όπω όπως το δικό μας να ε, μπορεί να ενθαρρύνει αυτή την προσπάθεια για την δημιουργία των μέσων αλλά και των τρόπων ανταπόκριση στην ψηφιοποίηση. Αυτό δεν συνδέεται και με του τοπικούς τομείς και κλάδους και σίγουρα αυτό θα εξυπηρετήσει όλους ε, με γνώμονα βέβαια και διακύβευμα τη δημιουργία ενός σωστού δικτύου που θα υπερβαίνει τα εδαφικά όρια. Προς το παρόν βλέπουμε να είναι περιορισμένες οι ανταποκρίσεις ε, στις ε, τεχνολογικές προκλήσεις. Πρέπει να βρούμε σωστά, σωστές Τεχνολογικέ προσεγγίσεις και η Ευρώπη να αποκτήσει νέα στοιχεία συνθετικά. Ευχαριστούμε η Ισπανία στη συνέχεια, αριθμός 617, Ελένα Άλβαρεθ. Ε, μεταξύ των δεκιβευμάτων που έχουν επιχειρήσεις είναι και αυτή της δημιουργίας των ικανοτήτων ε, των ορισμένων. Είναι ένα θέμα που ανακύπτει διαρκώς. Σίγουρα χρειαζόμαστε τρόπους να αντιμετωπίσουμε τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Ε, πραγματικά είμαστε σε μια στιγμή που πρέπει, αν διασυνδέσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα με τι ανάγκε που οι επιχειρήσεις έχουν για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Η επαγγελματική κατάρτιση θα πρέπει να βοηθήσει στην απάμβληση του προβλήματο με την δημιουργία εκπαιδευμένων και σωστά καταρτισμένων εργαζομένων και σωστή διασύνδεση επιχείρηση και ε, εκπαιδευτικού συστήματο. 74% ε, των νέων σήμερα ε, ναι, μεν έχουν πάρει δρόμου κατάρτιση, αλλά έχουμε ακόμα αρκετό έλλειμμα. Το χώρο των επιχειρήσεων, ανάλογα και τα δεδομένα της, ε, του επιμελητηρίου, 60% των επιχειρήσεων στην Ισπανία δεν έχουν ευκαιρία διασύνδεση με το κρατικό σύστημα. Ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δημιουργήσει ε, του τρόπου εκείνου και τι ευκαιρίε που θα μπορέσουν να προάγουν και να ενθαρρύνουν την δυσήμαντη επαγγελματική κατάρτιση. Η συμμετοχή των εμπορικών και επαγγελματικών επιμελητηρίων θα έχει ζωτική σημασία για την προώθηση αυτής της πρωτοβουλίας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you We continue with Croatia. Ευχαριστώ πολύ. Κροατία, αριθμός 18, Μαρίνκο Ντόσεν. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι επικεφαλής ε, ηγετικής ε, στη χώρα μου επιχείρηση στο χώρο ε, των πλαστικών που τροφοδοτεί την αυτοκινητοβιομηχανία. βιομηχανία. μας στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων μεταξύ των οποίων προκύπτει άλλωστε και αυτή η διαπίστωση της ανάγκης για κατάρτιση και για απόκτηση δεξιοτήτων σε διαρκή βάση. Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες η ακαδημαϊκή κοινότητα και ο πραγματικά ο οικονομικός ε, τομέας, εκεί όπου η επιχείρηση πάλεται, δεν έχουν κάλυψη ε, δεξιοτήτων. Συμβαίνει στη χώρα με αυτού για να βελτιωθεί η κατάσταση στο επίπεδο αυτό και να μπορέσει το εκπαιδευτικό σύστημα να αποδώσει αποτελεσματικά. Το δικό μας επιμελητήριο δρομολόγησε ένα σύστημα δυσήμαντης εκπαίδευσης, δηλαδή και θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης. Με βάση τα δεδομένα αυτά, περιμένω να μάθω η Ευρώπη πώ βλέπει να στηρίζει τέτοιου είδου πρωτοβουλίε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με το σημείο 2, το 4, Ευάγγελος Μυρσινίας, Ινσουλό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί συνάδελφοι, το όνομα μου είναι Ευάγγελος Μυρσινιάς, είμαι πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λέσβου από την Ελλάδα και αντιπρόεδρος του Ινσουλέρ του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νησιωτικές επιχειρήσεις αναφέρουν όλο, όλο ένα ε, και πιο μεγάλες δυσκολίες ε, για ορισμένες βασικές δεξιότητες, εν απουσία μάλιστα συντονισμένη δράση. Οι νησιωτικέ επιχειρήσει αναφέρουν επίση ότι μπορεί να είναι δυσκολότερη η πρόσβαση στην κατάρτιση σε τοπικό επίπεδο και όταν αυτή είναι διαθέσιμη μπορεί να είναι αρκετά ακριβή τα ποσοστά ανεργίας είναι υψηλότερα στις νησιωτικές περιφέρειες από ό,τι στους εθνικούς μέσους όρους και σε ορισμένες περιπτώσεις σε σημαντικό βαθμό. ωστόσο ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας είναι η διατήρηση και προσέλκυση ανθρώπων σε ηλικία εργασία. ενώ υπήρξε έντονη πληθυσμιακή ανάπτυξη που οφείλεται στην εσωτερική μετανάστευση αυτό συμβαίνει συνήθω σε ηλικίε 65 ετών και άνω. το πρόσφατο πρότυπο της εσωτερικής κυρίως μετανάστευσης έχει ενισχύσει τη μετακίνηση μεγαλύτερων ηλικιών προς τα νησιά μας και έχει δημιουργήσει έλλειμμα εξειδικευμένων ατόμων σε ηλικία εργασίας ιδιαίτερα στην ηλικιακή ομάδα 15 έως 39 ετών. Υπάρχει στη σκέψη των ηθινόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόθεση να λάβουν μέτρα για να αναστραφεί αυτή η τάση για τα ευρωπαϊκά νησιά που αποτελούν και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλτα. Αριθμό 526, ε, David Trerab. Κύριε Πρόεδρε, μικρόφωνο παρακαλούμε. Ε, μικρόφωνο παρακαλούμε. Μικρόφωνο παρακαλούμε, δεν μπορεί να υπάρξει διερμηνία χωρί μικρόφωνο. Sorry. Ζητώ συγγνώμη, παρακαλώ ε, ξεκινήστε από την αρχή γιατί δεν είχατε μικρόφωνο κύριε. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα από, το, από την επιχειρηματική κοινότητα της Μαλτά. Διάφορα δημοκρατικά φαινόμενα και οι τεχνολογικέ εξελίξει ταχαίω μεταρρυθμίζουν τι κοινωνίε και την αγορά μα. Νέε τεχνολογίε εμφανίζονται σε, με ρυθμού ασύλληπτου και τα εκπαιδευτικά συστήματα δεν μπορούν να κρατήσουν, να τηρήσουν το ρυθμό αυτό και να τον παρακολουθήσουν. Για να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, θα πρέπει οπωσδήποτε και από εκεί εξαρτάται οι, οι ανθρώπινοι πόροι μα να μπορούν να ανταπεξέλθουν στι προκλήσει αυτέ, ειδικά στι περιφερειακέ αυτέ ε, ζώνε όπου που ζούμε. Πρέπει να προσαρμοστούμε αποτελεσματικά σε αυτές τις εξελίξεις για να είναι ανταγωνιστικές οι περιοχές μας. Οι βασικοί μας ανταγωνιστές ε, ως Ευρωπαίων ε, είναι άνθρωποι και επιχειρήσει οι οποίοι ε, ε, δημιουργούν μεγάλη πρόοδο στους διαφορου τομείς Από την άλλη πλευρά βιώνουμε αποστράγγιση εγκεφάλων. Υπάρχουν όμως μεγάλες ευκαιρίες το ανθρώπινο αυτό δυναμικό που τόσο πολύτιμο είναι και που το χάνουμε να μπορέσει να αξιοποιηθεί και να επανέλθει μέσα από μια ε, σίγουρα φιλόδοξη επένδυση. Περαιτέρω ζητούμε να προσπαθήσουμε να το βοηθήσουμε αυτό και επίσης να ενισχύσουμε την υποχρεωτική εκπαίδευση και κατάρτιση. Τέτοιου είδου πρωτοβουλίε σίγουρα θα μας βοηθήσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ε, δεξιότητες να διατηρήσουμε και ε, άλλες να αποτρέψουμε από το να φύγουν. Όπω άλλωστε και ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόλι προηγού μα, είπε, ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να ε, εφαρμόσει πολιτικέ θαραλέε που θα μπορέσουν να, να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις αυτές. Τα, ζητούμε από τα Άνα την Ευρώπη επιμελητήρια να συνεχίσουν να ενισχύουν την προσπάθεια για διασύνδεση του κρατικού χώρου και, της, ε, και των επιχειρήσεων. Γαλλία, 161, ολυγέ Ζουλγκού. Καλή σας ημέρα. Ολιβιά Γκυλγκό. Είμαι επικεφαλής ε, ε, γαλλικής εταιρείας ε, που ασχολείται με την παρασκευή βιολογικών καλλιντικών. Είμαστε παρόντες και σε ένα δίκτυο απευθείας πωλήσεων με 1.500 πολιτές με εγκαταστάσεις που αριθμούν πάνω από 200 άτομα προσωπικό σε διάφορες μάρκες αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι υψηλές προδιαγραφές παραγωγής και ποιότητας μας ε, κάποτε γίνονται προσκόμματα και εμπόδια. Κάποιες φορές ε, τα βλέπει κανείς ως εγγύηση ποιότητας, ωστόσο και εγώ θα ήθελα να παραμείνουμε υψηλά ιστάμενοι στις προδιογραφές, αλλά για να μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους άλλους στο μέλλον θα πρέπει κάτι να γίνει ε, σε πρόσφατη ε, συμμετοχή μου σε ε, ασιατική διάσκεψη μάθαμε ότι η Κίνα κάνει πράγματα διαφορετικά από εμάς αξιοποιούν τις δεξιότητες και λόγω της ενδογνωστικότητάς τους μας απειλούν πρέπει λοιπόν να αυξηθεί η ενδογνωστικότητά μας να επιταθεί η απασχολησιμότητα των νέων μας αλλά με μια μεγαλύτερη ευελιξία στις προδιαγραφές για να μπορούμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε σε ένα προκλητικό παρόν και μέλλον Δύο ερωτήματα λοιπόν Πώς θα διευκολύνουμε την πρόσβαση σε ε, κονδύλια κατάρτισης ε, ε, από την τροπία του de ε, βοηθήματος και κατά δεύτερο πώς θα ενθαρρύνουμε τη μαγειμενική κινητικότητα με προγράμματα όπως το Erasmus ε, έτσι ώστε να υπάρξει μια διευρωπαϊκή πλατφόρμα στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Πορτογαλία υπαριθμό 504 Μπερνάρντου Αγιάρ. Στην εταιρεία μου παροχή συμβουλευτικών επιχειρήσεων ασχολούμαστε κυρίως με όλους τους τομείς της ε, αλυσίδας αξίας των αυτοκινήτων. Ζητούμε ένα πρόγραμμα όπως το Erasmus Plus που συγκερνά 24 ε, εταίρου από 11 χώρες και ασχολούνται όλοι μαζί με την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν την αλυσίδα αυτή. Ο χώρος της, ε, ε, του αυτοκινήτου χρησιμοποιεί προσωπικό με 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ανά την Ευρώπη. Στην Ευρώπη, Σε Πορτογαλία με συγχωρείτε, 230 εταιρείε, 51.000 θέσεις εργασίας και 5% του καθαρίστου εθνικού προϊόντος. Λοιπόν, δύο σύντομα μηνύματα. Χρειαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις προκλήσεις που τίθενται. Η προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ε, είναι τεράστια για την παραδοσιακή μα βιομηχανία. Παρακαλούμε αυτά να τα έχετε τα δύο κατά νου όταν διαπραγματεύεστε το επόμενο πολιετέ χρηματοοικονομικό πλαίσιο. Δεύτερον, όσον αφορά τι δεξιότητε του μέλλοντο, παρακαλούμε να ζητήσετε τρόπου αμοιβαία αναγνώριση και επιστοποίηση των δεξιότητων εκείνων που θα έχουν θεμελιώδη σημασία για την ανάπτυξη των βιομηχανίων. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια η Βουλγαρία, αριθμός 25, Ρώσαν Δασκάλοφ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, ονομάζομαι Ρώσαν Δασκάλοφ, κόμμανι Σίμκαρ. ε, Βουλγαρία. Είναι, είμαστε στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Βουλγαρία. Ξέρουμε ότι οι δεξιότητε είναι τεράστια σημασία. Παιδιά, εκπαίδευση, δουλειά, λέξει κλειδιά ε, μιλώ σαν γονιό και σαν επιχειρηματία και ξέρω ότι πρέπει να ετοιμάσουμε την νέα γενιά των νέων ανθρώπων για τι προκλήσει τη πραγματική ζωή. Να του παρέχουμε τι καλύτερε δεξιότητε εκ των προτέρων. Προ την κατεύθυνση αυτή κινούμενη, η Βουλγαρία πετύχε ήδη να εφαρμόσει τα πλαίσια του παιδικού συστήματο ε, ε, πολύ καλέ ε, δομέ επαγγελματική κατάρτιση. Δεδομένη τη πρώην καριέρα μου ω επαγγελματία οδηγού ράλι, μπορώ να σα πω ότι το σύστημα τη εκπαίδευση, όχι μόνο στη Βουλγαρία, αλλά σε όλη την Ευρώπη, θα πρέπει να περιλάβει και το θέμα τη ασφάλεια στο, στον τομέα τη οδήγηση αυτοκινήτων. Είναι κάτι σημαντικό. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώ όλα αυτά ε, μπορούν να συγκεραστούν σε μια προσέγγιση επιβίωση στη ζωή και τον δρόμο. Ζητώ από τι ευρωπαϊκέ χώρε να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση και να παρέχουν στα παιδιά μα τι βασικέ δεξιότητε για να μπορούν να επιζήσουν και στο τιμόνι και στο δρόμο. Σώστε το μέλλον μα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Germany. Η Γερμανία 200. Hans Peter Volsheimer. Γεια σα. είμαι ο Hans Peter Volsheimer, είμαι από την Κολονία και είμαι επικεφαλής ε, μιας ε, εμπορικής εταιρείας. Έχουμε βεβαίως ε, καταρτισμένους εργαζόμενους και χρειαζόμαστε περισσότερους. Πρέπει να, θέλουμε να επενδύσουμε σε αυτούς, θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους νέους ανθρώπους να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται και θέλουμε να ενισχύσουμε αυτές τις δεξιότητες και να τους βοηθήσουμε στις δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να βιώνουν. Θέλουμε επίσης να βοηθήσουμε και νέους που προέρχονται από άλλες χώρες Επίσης, είναι είναι ένα υψηλά ποιοτικό επίπεδο κατάρτιση το οποίο χρειαζόμαστε μέσα από το Εράσμους και μέσα από, το, από τα προγράμματα ISF+. Plus. Έτσι μπορούμε να ενισχύσουμε την επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση. Μέσα, πρέπει να δημιουργήσουμε συμβουλευτικά συστήματα που θα βοηθήσουν να καλύψουμε τα κενά μεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης και του κόσμου ε, της ε, εργασίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με την Πολωνία. 501, ο Γιαρόζο Φόροκ. Η αυτοκινητοβιομηχανία χρειάζεται ε, διαβίου μάθηση επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό είναι μια σύνοψη όσων ελέγχθησα νωρίτερα. Το μαθαίνω κάνοντας θα πρέπει να αποτελέσει το μέλλον της επαγγελματικής κατάρτισης το μέλλον καθώς και των προγραμμάτων κατάρτισης. Τέτοια μαθήματα, πρακτικά ουσιαστικά, θα πρέπει να αφιερώνονται ε, στους ακαδημαϊκούς, στους εκπαιδευτές, στους φοιτητές, ε, στους μαθητές και θα πρέπει να αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της μεταφοράς ε, τεχνογνωσίας από τον ένα κόσμο στον άλλο. Οι εκπαιδευτές και οι ακαδημαϊκοί θα πρέπει να μάθουν από τους εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας τι είδους γνώση και δεξιότητες χρειάζονται περισσότερο. Θα πρέπει οι εμπειρογνώμονες να μάθουν πώς οι ανάγκες τους θα μετατραπούν σε ένα ε, αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα. Πιστεύω ότι για να δημιουργήσουμε έτσι μια μακρά σχέση συνεργασίας αυτό είναι απαραίτητο και έτσι ώστε να αναπτύξουμε και αμοιβαία κατανόηση. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Η Κύπρος, το νούμερο 2, ο Μάνθος Μαυρομάτης. We all expect the Euro... Όλοι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ε, ισχυρή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα φοβόμαστε όλοι ότι οι ε, κενές θέσεις ε, θα αυξηθούν και δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις θέσεις. Χρειαζόμαστε εκπαιδευτικά προγράμματα και επαγγελματική κατάρτιση για να αντιμετωπίσουμε τις νέες ε, ανάγκες τις νέες οικονομίες. Ζητάμε από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να συμπεριλάβουν ε, επιχειρηματικούς εκπροσώπους ε, σε αυτή την πολυδιάστατη προσπάθεια σχεδιασμού κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κατάρτισης για το μέλλον. Με τον τρόπο αυτό θα είμαστε σε θέση να ε, δώσουμε την ευκαιρία στην επιχειρηματική κοινότητα να δημιουργήσει την ευημερία που όλοι χρειαζόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Η Τσεχία, 14, ο Ιαν Ρόμπα. Χαίρετε. Είμαι διευθύνων σύμβουλος μιας ε, startup ε, από την Τσεχία να πω δύο πράγματα. Αν η Ευρώπη θέλει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μέλλον, να είναι ανταγωνιστική και καινοτόμα στο μέλλον, τότε πρέπει να αλλάξουμε την παιδεία, την εκπαίδευση. Και αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρέπει να εκπαιδεύουμε όχι εμ, επιχειρηματικούς εργαζόμενους, αλλά ε, ιδρυτές νέων εταιριών, γιατί αυτοί είναι εκείνοι που θα δημιουργήσουν το χώρο εργασίας και πρέπει να ε, εκπαιδεύσουμε και πραγματικά πραγματικούς υπερασπιστές έτσι, της ανάπτυξης που αναπτύσσουν δηλαδή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Σλοβακία. Η Σλοβακία 4,75 η Ρενάτα Κουρντουλιακόβα. Good afternoon. Χαίρετε. Είμαι από το Σλοβακικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Είμαστε μια μικρή χώρα. Όμως, νομίζω ότι έχουμε πολύ ισχυρή αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε δεν είναι υψηλά καταρτισμένο προσωπικό, με μορφωτικό επίπεδο υψηλό, αλλά χρειαζόμαστε εργάτες ε, με πιστοποιητικά τεχνικής γνώσης. Και η ερώτησή μου είναι πόσο μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας βοηθήσει ε, να υλοποιήσουμε αυτό μας το σχέδιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Σας καλώ λοιπόν να βάλετε το το μπάτζο δεν είναι εκπιστωτική. Μην φοβάστε ότι θα σας σηκώσει χρήματα από το λογαριασμό. Θα βάλετε λοιπόν στο μηχάνημα την κάρτα και θα περάσουμε μια σειρά ερωτήσεων. Ερώτηση 1. Η επιχειρηματική κοινότητα ε, ε, συμμετέχει αρκετά στην πολιτική εκπαίδευση, ε, όπως είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων. Ψηφίστε. infatti. infatti. Thank you very much. Ευχαριστούμε. Λήξη της ψηφοφορίας. Λοιπόν, αποτέλεσμα. 537 ψήφισαν, 112 ναι, αρκετά συμμετέχει, 406 άτομα είπατε όχι, ευχαριστούμε πολύ. Δεύτερη ερώτηση. Είναι δυσκολότερο να προσλάβει κανείς προσωπικό με τις σωστές δεξιότητες σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια. Άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ ψηφίστε. It's green. There's no one Thank you. Ευχαριστούμε. Λήξη ψηφοφορίας. 532 ψήφοι, 408 ψήφοι ναι. Είναι δυσκολότερο να προσλάβουμε ανθρώπους με σωστές δεξιότητες. Ερώτηση 3. Θα πρέπει η απασχολησιμότητα των αποφύτων να αποτελεί το πιο σημαντικό κριτήριο στην, στην βαθμολόγηση των επιδόσεων για, τους, ε, για τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης. Ψηφίστε. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Λήξη της ψηφοφορίας. Τα αποτελέσματα. 534 ψήφοι. 427 ε, άτομα πιστεύουν ότι η αποσχολησιμότητα των ε, αποφύτων θα πρέπει να είναι ένα κριτήριο έτσι, βαθμολόγησης της εκπαίδευσης των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ερώτηση 4. Θα πρέπει η εκμάθηση που βασίζεται στην εργασία να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όλων των αρχικών επαγγελματικών ε, προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης. Ψηφίστε. Tutto verde. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Λήξη της ψηφοφορίας. 534 ψήφισαν. 505 πιστεύουν ότι ναι, θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι σε όλα τα προγράμματα επαγγελματική κατάρτισης και εκπαίδευσης. Ερώτηση 5. Το κόστος αποτελεί ένα σημαντικό πρόσκομα στις επιχειρήσεις για να προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης ή εργασίας σε πρόσφυγες και μετανάστες. Ψηφίστε. Thank you very much. Ευχαριστούμε. Λήξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν 524, 168 είπαν ναι, 268 είπαν όχι. 88 αποχές. Ευχαριστούμε. Τώρα, θα δώσουμε το λόγο στον... στους ανθρώπους μας που θα απαντήσουν. Έχουμε τον Μπράντο Μπενιφέη ανάμεσά μας ο οποίος θα μιλήσει. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε ανάμεσά σας. Είμαι ο Μπράντο Μπενιφέη, είμαι μέλος ε, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως και η συνάδελφός μου η Μαρτίνα. Συνεργαζόμαστε, μερικές φορές συμφωνούμε, άλλες διαφωνούμε. Είμαστε ένα κοινοβούλιο όπου ακούγονται διάφορες ιδέες, διάφορες προτεραιότητες, πολλές ιδέες εκπροσωπούνται. Βασικά ο ρόλος μας είναι να ε, λαμβάνουμε όλα όσα προκύπτουν από το δικό σας κόσμο και να τα συνδυάζουμε με άλλες απόψεις που τίθενται επιτάπητος όταν συνεργαζόμαστε πάνω σε διαφορετικά θέματα και να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία ώστε να προχωρήσει και για ε, να προσφέρουμε αποτελέσματα στις επιχειρήσεις, στους πολίτες, στους εργαζόμενους. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Με συγχωρείτε γιατί κάποια στιγμή ίσως μπορεί να αλλάξω και να μιλήσω και στα ε, Ιταλικά, έτσι και για να τιμήσω και τους ε, συμπατριώτες μου που είναι σήμερα παρόντες, καθώς και για το Union Camera, το επιμελητήριο, το οποίο γνωρίζω πολύ καλά. Ε, θέλω όμως επίσης να πω ευχαριστώ στο Eurochamber, και σε όλες τις εθνικές ε, οργανώσεις ε, των ε, εμπορικών επιμελητηρίων, γιατί ακριβώς αυτό που λέω, ότι δουλεύουμε πολύ καλά μαζί, συνεργαζόμαστε πολύ στενά. Προσπαθούμε να προωθήσουμε τις δικές σας προτεραιότητες εντός των διαφόρων έτσι, φακέλων. Προσωπικά εγώ δουλεύω για τις ψηφιακές δεξιότητες. Το δουλεύουμε αυτό στην, της, στο πλαίσιο της νέας ατζέντα ε, της ε, Κομισιόν. Ακούμε τις προτάσεις σας, δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Συνεργαζόμαστε απευθείας με τις επιχειρήσεις που χρειάζονται εκπαιδευμένο, καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, κυρίως ε, στα πλαίσια των ψηφιακών δεξιότητων. Προσφάτως, συνεργαστήκαμε και στο ε, θέμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης που είναι ένα σημαντικός φάκελος και βεβαίως ε, με την προοπτική του νέου ε, πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου μιλάμε για 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να διατηρήσουμε τέτοιες δράσεις και για την απασχόληση και για την πρακτική εξάσκηση Ξέρετε ότι αγωνιζόμαστε πολύ προκειμένου να συμπεριλάβουμε και τον επιχειρηματικό τομέα και την κοινωνική οικονομία και τα εμπορικά επιμελητήρια σε αυτό το project. Γιατί ξέρετε, το να δημιουργήσουμε μια πιο συνοχική ε, και δίκαιη Ευρώπη είναι μεγάλη ευκαιρία για όλους τους οργανισμούς και συνεργαζόμαστε και πάνω στα ευρωπαϊκά ταμεία και με το κόσμο, αλλά και για την πρόσβαση στην ε, πίστοση και θα προσπαθήσω εδώ να θίξω και κάποια από τα ζητήματα που αναφερθήκατε με το Ταμείο Κόσμη, με το ε, νέο σχέδιο Juncker για τις επενδύσεις. Έχουμε συνεργαστεί στενά προκειμένου να ε, προσφέρουμε περισσότερες ευκαιρίες χρηματοδότησης για νέα σχέδια από τον επιχειρηματικό κόσμο και επειδή και πρέπει να σας πω ότι συνεργαζόμαστε και στενά και με τους νέους επιχειρηματίες, νεαρούς δηλαδή. Υποστήριξη λοιπόν για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ε, μικρομεσαίων, αλλά και με το Εράσμος για τους νέους επιχειρηματίες. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα και η Μαρτίνα και εγώ Είμαστε ε, πρέσβεις αυτού του προγράμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσπαθούμε να ε, διαδώσουμε αυτή την ιδέα και στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να φέρουν όλο και περισσότερους νέους επιχειρηματίες να συμμετάσχουν σε αυτά τα σχέδια κινητικότητας. Γιατί διακούσαμε από εσάς, κάποιοι το είπατε, ότι δουλεύετε με αυτά τα ταμεία και για να ενισχύσετε τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, αλλά και για να ανταλλάξετε δεξιότητες. Ακούσαμε π.χ. Ε, τη δουλειά που γίνεται για την ανταλλαγή δεξιοτήτων στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας ε, βάσει ευρωπαϊκών ε, σχεδίων και ο ίδιος προσωπικά έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλά σεμινάρια και εδώ στο Κοινοβούλιο και εκτός και νομίζω ότι αυτού του είδους η ανταλλαγή είναι πάρα πολύ σημαντική γνωρίζοντας ότι εν μέρει αυτή η προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί και από τα εθνικά κράτη-μέλη και από τις περιφέρειες που σε πολλές χώρες είναι, αν θέλετε, οι ε, επιχειρησιακές αρχές για τα ε, ευρωπαϊκά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που είναι πολύ σημαντικό για, για, για την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. Ε, δεύτερη ερώτηση. Είδαμε μια θερμή απάντηση και λέτε ότι σας λείπουν ακόμη ε, οι εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι. Τώρα το δουλεύουμε και εμείς ηγητής, εγώ για την πολιτική ομάδα μου, για τους σοσιαλδημοκράτες. Η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι. Δουλεύουμε λοιπόν για το ECT το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, δηλαδή ΣΥΝ, και εστιαζόμαστε πολύ στην διαβίου μάθηση των εργαζομένων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για σας δηλαδή να έχετε τη δυνατότητα να έχετε ένα εργατικό δυναμικό το οποίο είναι ενημερωμένο σχετικά με τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και την αλλαγή ως προς τις απαιτήσει που προέρχονται από τη βιομηχανία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σίγουροι ότι τα ευρωπαϊκά χρήματα κατευθύνονται με τον καλύτερο δυνατό ε, τρόπο στη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει και η ε, πρωτοβουλία για την εγγύηση για τον νέο, ότι υποστηρίζουμε δηλαδή ε, την κατάρτιση και την απασχόληση νέων ανθρώπων σε εταιρείε. Από την πλευρά μας πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το κάθε ευρώ και το κάθε ε, ευρωπαϊκό ε, ευρώ χρησιμοποιείται για να χρηματοδοτήσει ποιοτικά σχέδια, για να προσθέσει αξία και για σας και για τις περιοχές τις οποίες να σταματήσουμε αυτό το brain drain, αυτή την ερήμωση ε, και εδώ χρειαζόμαστε λοιπόν κινητικότητα, πρέπει να την ενισχύσουμε έτσι ώστε ο, ο κόσμος να βγαίνει και να αποκτά εμπειρία στο εξωτερικό, αλλά μετά αυτές τις εμπειρίες να τις φέρνει μέσα πάλι. Ό,τι έμαθα ο καθένας να ε, το μεταφέρει στη χώρα του. Οι άνθρωποι που έχουν συμμετάσχει στο Εράσμους, ανταλλαγές αυτές και στο εράσμο των νέων επιχειρηματιών βλέπουμε ότι είναι πιο ανθεκτικοί, βλέπουμε ότι έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους ε, εργοδότες, ε, βλέπουμε ότι ξεκινάνε καλύτερα την επιχείρησή τους όταν γίνονται επιχειρηματίες από την άλλη πλευρά. Ε, υπάρχει κακή κινητικότητα αυτή, η οποία αφορά εκείνους που φεύγουν διότι δεν βρίσκουν ευκαιρίες στη χώρα τους. Και για αυτούς λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μας για μια καλύτερη οικονομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να ανακάμψουμε σε κάποιες χώρες. Ακούσαμε κάποια παραδείγματα στις παρεμβάσεις. Να εξακολουθούμε να ε, χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις από το ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να οδηγήσουμε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Η προσέγγιση μου και νομίζω ότι συμφωνούμε ε, ως προς αυτό και με τους ε, συναδέλφους ότι τα κίνητρα είναι πολύ σημαντικά δουλεύουμε πάνω σε εργαλεία για να το διευκολύνουμε όλο αυτό, αλλά αν η οικονομία έχει πρόβλημα, αν δεν υπάρχει αύξηση των θέσεων εργασίας, νέες θέσεις που θα προέρχονται από μια αλλαγή της κατάστασης σε μακροοικονομικό επίπεδο, τότε όλα τα κίνητρα, όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν πρόκειται να έχουν αποτελέσματα και πολιτικές επίσης δραστηριοποίησεις για τη διαβίου μάθησης. Αυτά, ξέρετε, στο τέλος κινδυνεύουν να γίνουν απλά ε, φτωχά επιδόματα για κάποιες μεταβατικές περιόδους. Πρέπει λοιπόν ανταυτού να έχουμε έναν ουσιαστικό οικονομικό ρόλο για να σταματήσουμε την εγκατάλειψη των ε, νέων από τις χώρες τους. Πρέπει επίσης να προσελκύσουμε περισσότερους νέους ανθρώπους από άλλα μέρη του κόσμου στις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν ε, είναι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες σε θέση να καλύψουν τις ε, θέσεις τους και χρειάζονται επαγγελματίε και επιχειρηματίες από άλλες χώρες. Τώρα το τελευταίο κομμάτι θα το πω στα Ιταλικά, όπως σας είπα προς τιμήν των συμπατριωτών μου. Λοιπόν, άρα πραγματικά ασχοληθήκαμε επίσης με το θέμα της ε, ενσωμάτωσης, της ένταξης του σχολείου και τη μετάβαση από το σχολείο στη δουλειά. Αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό θέμα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι θεσμοί ε, υποστηρίζουν το διτό αυτό σύστημα. Είναι ένας τρόπος κατάρτισης, όπως για παράδειγμα στην Ιταλία, δηλαδή η χώρα μου, έκανε κάποιες μεταρρυθμίσεις πέρσι προς ε, μια εκμάθηση που θα βασίζεται περισσότερο στην πρακτική, διότι πρέπει να φέρουμε πιο κοντά τον κόσμο της μάθησης με τον κόσμο των επιχειρήσεων και θα πρέπει να προσφέρουμε ε, ικανοποιητικές ευκαιρίες. Δεν σας λέω ότι όλα είναι τέλεια, ότι είμαστε καλύτεροι στον κόσμο. Πάνω σε αυτό το, το σημαντικό θέμα θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή δέσμευση, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία ε, του περάσματος από σχολείο στη δουλειά. Χρειαζόμαστε κοινέ προσπάθειες όλες της επιχειρηματικής κοινότητας να φροντίσουμε ώστε αυτή η μετάβαση γίνεται με ποιότητα και αποτελεί μια ευκαιρία που δίνει τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να εισέλθουν σε αυτό το διτό σύστημα εκπαίδευση, να έχουν εμπειρίες που τους εκπαιδεύουν και που είναι χρήσιμες στον οικονομικό κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν οι θεσμοί πρέπει να δουλέψουν πάνω σε αυτό, αλλά και ο κόσμος των επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι η ανταλλαγή καλών πρακτικών ε, μεταξύ των χωρών είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό να υπάρξει μια ανταλλαγή, είναι χρήσιμο ε, για όλες τις χώρες Κάποιες χώρες ε, δούλεψαν αυτά τα θέματα τα τελευταία χρόνια προκειμένου να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε ε, δουλέψει. Είναι πολύ σημαντικό για τους νέους ανθρώπους, είτε είναι εργαζόμενοι είτε επιχειρηματίες. Και ένα άλλο θέμα είναι η αναγνώριση των ε, πτυχίων Έχουμε ενιαία αγορά για, για αγαθά, για ανθρώπους, για την αγορά. Δεν έχουμε μια ενιαία αγορά για την αμοιβαία αναγνώριση των ε, πιστοποιητικών ε, και πτυχίων και δεξιοτήτων. Τα κράτη-μέλη πρέπει να βοηθήσουν το ένα το άλλο και μερικές φορές ε, θα πρέπει να, δεν πρέπει να φοβούνται να δώσουν τη δυνατότητα να έχουν προκειμένου να έχουν αποτελέσματα. Αν κατακλείδει, ε, θα αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και το συζητήσαμε. Ο επιχειρηματικός κόσμος υπό το ρόλο του έτσι προσδιορισμού ευρωπαϊκών πολιτικών με το Euro, ε, Euro Chamber κάνουμε πολλή δουλειά μαζί αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα κυρίως όταν χρησιμοποιούμε τα ευρωπαϊκά ταμεία τα οποία τα αποφασίζουμε εδώ. Όταν αυτά ασχολούνται με αυτά τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και διαχειριστικές αρχές ε, σε πολλούς τομείς πρέπει να, να διατηρούν για όλα τα ταμεία και κυρίως για αυτά που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη ε, ε, ένα διάλογο. Πρέπει να υπάρχει διαρκής διάλογος με τον κόσμο της παραγωγής. Ε, κινηθήκαμε πολύ προς αυτή την κατεύθυνση ε, εδώ στους θεσμούς, αλλά πρέπει να εκμεταλλευτούμε και το ε, νέο πλαίσιο. Πρέπει και να απλοποιηθεί η πρόσβαση στα κονδύλια, αλλά πρέπει να υπάρξει Ε, ε, να υπάρξει μεγαλύτερη συνέπεια και σε περιφερειακό επίπεδο. Χρειάζεται λοιπόν μια κοινή προσπάθεια για να το καταφέρουμε αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πραγματικά ο θεσμός εκείνος ο οποίος είναι πιο κοντά στις ανάγκες των ανθρώπων και ε, των γεωγραφικών περιοχών. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να είμαι σήμερα μαζί σας. Άκουσα όλα όσα είπατε και τα έχω σημειώσει. Ωραία, θα κλείσουμε με μια πρόταση από την Μαρτίνα Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να σας κρατήσω. Ξέρω ότι πρέπει να πάτε τώρα να φάτε. Απλώς ε, μόνο μία απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις που θέσατε κατά τις παρεμβάσεις σας. Όλοι σχεδόν αναρωτιέστε τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για εμάς. Λυπάμαι που θα σας πω το μυστικό, αλλά όλοι είμαστε Ευρώπη. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε όλοι μαζί έχει σημασία. Όλο αυτό που κάνουμε, αυτό θα γίνει. Δηλαδή, όχι ότι η Ευρώπη θα το κάνει για μας. Εμείς είμαστε η Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα έχουμε διάλειμμα για φαγητό. Ε, μία ώρα. Σας ζητώ λοιπόν να επιστρέψετε στην ώρα σας στις 2 και 20 για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Ευχαριστώ.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

Mm-hmm. Mm-hmm.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 Ladies and gentlemen, I invite you to take your seat, please. Κυρίες και κύριοι, οι εργασίες μας θα επαναληφθούν αμέσως μόλις έχετε όλοι πάρει τις θέσεις σας. Γι' αυτό και σας παρακαλώ, καθίστε.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 ισκομίσετε οτιδήποτε υγρό στην αίθουσα, μπουκάλια νερού ή καφές θα πρέπει δυστυχώς να μείνει εκτός της αίθουσας. Please. Παρακαλούμε να λάβετε τις θέσεις σας λοιπόν για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. das kommt sitzen, nicht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 ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το εμπόριο Σεσίλια Μάλστρόμα και τον πρόεδρο ε, του ε, τμήματος εμπορίου του Κοινοβουλίου, τον κύριο Μπέντ Λάγκα. Ζητώ και από τους δύο να έρθουν κοντά μας στο βήμα. Now we can... Μπορούμε λοιπόν ευθύ αμέσω να ξεκινήσουμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για την συνεδρία αφιερωμένη στο εμπόριο. το βήμα στο μέρος του Κοινοβουλίου ε, κύριο Μπέρτ Λάγκε. Να σας υπενθυμίσω ότι στην προηγούμενη του καριέρα ήταν ε, βάσκαλος. Κάποιο ειδικό τρόπο θα έχει να μας ε, μιλήσει για το εμπόριο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι εδώ πλέον είμαστε αντιμέτωποι με μια διτή κατάσταση όσον αφορά το εμπόριο. Από τη μια πράγματι θα το παραδεχτούμε ότι υπάρχει πολιτική και οικονομική ανάγκη για περισσότερο εμπόριο, ιδίω εν ώψη της εξέλιξης της παγκόσμιας αλυσίδας αξίας, πάνω από 100% του παγκόσμιου εμπορίου δεν συνδέεται με αυτή την παγκόσμια αλυσίδα αξία. Όπως επίσης όλοι γνωρίζουμε, έχει γίνει πια συνείδηση ότι το εμπόριο δεν έχει να κάνει μόνο με δασμούς, έχει να κάνει και με πρότυπα, με προδιαγραφές, με νομοθετικά πλαίσια, με συνεργασία, με προστασία του καταναλωτή, με εργασιακά δικαιώματα, με την τήρηση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών και την προστασία του κλίματος. Με άλλα λόγια, έντονη διαγράφεται η ανάγκη για περισσότερο διεθνοποιημένο εμπόριο, με τρόπο όμως ρυθμισμένο. Και η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι η αυξανόμενη τάση που βλέπουμε να αναπτύσσεται βάσει της οποίας ε, έχουμε τον κύριο Τραμπ ο οποίος έρχεται και ακυρώνει πολλές διεθνείς συμβάσεις που μέχρι σήμερα ίσχυαν δίνοντάς μας σαφή ένδειξη της επιθυμίας του να παραμείνει πιστός στην αρχή της ε, δύναμης, της απόλυτης ισχύω που σημαίνει δεν δέχεται το κράτος δικαίου και ε, θέλει να έχει την ευχαίρεια να ασκεί πίεση όχι μόνο στους εμπορικούς του εταίρους αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη μέσα από την επιβολή δασμών για τον χάλιβα και για το αλουμίνιο με περαιτέρω περικοπές στον ορίζοντα και δεσμεύσεις. Είναι μέτρα, και και να μας αρέσει ο όρος, προστατευτικά Δύο λοιπόν πλευρές του νομίσματος είναι αυτές ε, που αναπτύσσονται και εξελίσσονται με τρόπο τελείω ξέχωρο. Από τη μια μεριά βλέπουν ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ρύθμιση, περισσότερο κράτος δικαίου και περισσότερο ε, ε, ισχυροποιημένο νομοθετικό πλαίσιο και από την άλλη όλο και αυξανόμενη είναι η τάση λήψης προστατευτικών μέτρων ανά τον κόσμο. Και τι να κάνουμε, αυτή είναι η συγκεκριμένη πρόκληση που έχει μπροστά της Ευρωπαϊκή Ένωση είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η δικό μας καθήκον είναι πράγματι να είμαστε επικοδομητικοί σε προσπάθειες ε, υπερκερασμού αυτής της δεύτερης πλευράς του νομίσματος και αυτό προς το συμφέρον των επιχειρήσεων ανά την Ευρώπη, προς το συμφέρον ε, της αηφορίας της ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και προκειμένου ε, το εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη να κατοχυρούται. Είναι απόλυτα σαφές ότι το εμπόριο αποτελεί τον κινητήρα, τον μοχλό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, υψηλότερων αμοιβών, με 60% παραπάνω των μισθών που έχουμε προκειμένου για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εξαγωγικό τομέα. Με άλλα λόγια πρέπει να είμαστε πραγματικά επικοδομητικοί, ευρηματικοί και στηρίζουμε την δέσμευση που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθεια αυτή που κινείται σε δύο κατευθύνσεις. Αφενός, προφανές άλλωστε είναι, να προσπαθήσει να σταθεροποιήσει ε, το ε, πολύπλευρο εμπορικό σύστημα με σκοπό την αναθεώρηση του ΠΟΕ και ειδικά όσον αφορά την τάση αυτή της, ε, του προστατευτισμού που βλέπουμε να διαχέεται είναι σημαντικό να προχωρήσουμε με αυτή την προσπάθεια και το παλιό μας κουρασμένο πλοίο να μπει πάλι ξανά στη ρότα του, γιατί κάπου έχει ξενερίσει. Νομίζουμε ότι είναι αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο παγκόσμιας οργάνωσης εμπορίου και όσον αφορά τις μέχρι τώρα πρακτικές στον ΠΟΕ είμαι πεπισμένος ότι σαφώς τα εκκρεμεί ζητήματα όσον αφορά την ε, διασφάλιση περισσότερων στοιχείων ανάπτυξης ε, στην ΠΟΕ πρέπει οπωσδήποτε ήδη από τώρα να τεθούν επιτάπητος όπως επίσης χρειαζόμαστε και νέα στοιχεία, νέες πτυχές όπως αναφορά ε, το συγκερασμό της ψηφιοποίηση, η οποία όλο και προχωρεί. Έτσι σίγουρα το ηλεκτρονικό εμπόριο πρέπει να τεθεί στην ατζέντα του ΠΟΕ ε, σίγουρα τα θέματα της φτώχειας που κυκλοφορεί και διάφορα θέματα. Χρειαζόμαστε επίσης να καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργεί ε, και ο η δευτεροβάθμια βαθμίδα εκδίκασης υποθέσεων στην ε, ΠΟΕ έχει να κάνει με τις ΙΠΑ αυτό. Ένα κομμάτι αυτού, του, αυτής της δομής δεν ανταποκρίνεται στην αποστολή της και πρέπει να βρεθούν λύσεις σίγουρα αν πρόκειται να παραμείνει στη θέση του ΕΟΠΟΕ και βέβαια η ιστορική δομή του όλου έργου του ΠΟΕ με ιδιαίτερη έμφαση στην μεταρρύθμιση του ρόλου του Γενικού Γραμματέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβηκε με πρόταση μεταρρύθμισης και θα συζητηθεί στην ΟΤΑΒΑ πολύ προσεχώς όταν γίνει η επερχόμενη συνάντηση. Ίσως αυτή η προσέγγιση να αποτελέσει τη γέφυρα στην όλη διαδικασία, ένας τρόπος για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά, έτσι ώστε αυτός ο οργανισμός που τόσα πολλά έχει προσφέρει να συνεχίσει να προσφέρει. Κατά δεύτερο λόγο, η διμερή μας ατζέντα, και ως προς αυτό είμαι πεπισμένος ότι μέσα σε αυτό το πνεύμα α, αβεβαιότητας θα είναι καλό να έχουμε διμερείς ε, συμφωνίες επίσης μακρέ και κάποτε δύσκολε οι συζητήσεις που είχαμε με τον Καναδά κι όμω να που σήμερα ο Καναδά έχει ήδη ζητήσει εδώ και ένα χρόνο να συμπεριληφθεί στις συνεννοήσεις μας για εξαγωγές ειδικά με, για μηχανήματα και το μέσα αυτός εφελείται πάρα πολύ όχι μόνο αυτός αλλά και άλλοι και άλλοι τομείς επίσης ωφελούνται άρα ε, αναφέρουμε πρόοδο και σε επίπεδο διμερών συνεννοήσεων ανέφερα τον Καναδά και επί τη ευκαιρία να πούμε ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επέλθει και η επικύρωση της συμφωνίας με την Ιαπωνία. Έχουμε συμφωνία και με το Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ. Ε, είναι αυτές ε, ήδη Αναμενόμενε και αναμένεται η υπογραφή τους να σταθεροποιήσει περαιτέρω το γενικότερο κλίμα μαζί με διάφορες άλλες διμερεί που όπως ανέφερα ανταποκρίνονται στην ανάγκη για την λήψη μέτρων που να διασφαλίζουν καλέ εμπορικές συναλλαγές. Έχω την πεποίθηση ότι έχει μεγάλη σημασία και καθήλη εφαρμογή όλων αυτών, η εκτέλεση των όλων των συμβάσεων. Ε, βλέποντας το θέμα της, ε, ε, των δικαιωμάτων χρήσης ε, πρέπει να προσέξουμε την εκτέλεση των όρων της σύμβασης ειδικά έτσι μικρομεσαίας έχει μεγάλη σημασία αυτό έχουμε πολλές και διάφορες συμβάσεις που αφορούν κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη δημιουργία ενιαίων θηρίδων συναλλαγής one stop shop δικτυακών τόπων αλλά δεν αρκεί όλο αυτό σίγουρα για τις μικρομεσαίες ε, υπάρχουν ακόμα προσκόμματα όσον αφορά την αξιοποίηση των διαφορών προτεραιμάτων που απορρέουν από τις εμπορικές συμφωνίες. Οπότε καλό θα είναι να δουλέψουμε και στο επίπεδο αυτό. Μα ακόμα και ο Καναδάς που ανέφερα προηγουμένως. Οι εθνικές αρχές δεν ήταν πραγματικά έτοιμες να παράσχουν απερίφραστη υποστήριξη στις επιχειρήσεις για να αξιοποιήσουν τα προτερήματα ε, που απορρέουν από τις εμπορικές συμφωνίες. Ένα παράδειγμα, μια εταιρεία που κατασκευάζει μοντέρνα συστήματα θέρμανσης και θέλει να εισέλθει στην καναδική αγορά, ε, αντιμετωπίζει τον φορέα πιστοποίησης, ε, δεν ήταν έτοιμο να χορηγήσει το πιστοποιητικό που απαιτείται προκειμένου να κυκλοφορήσουν τα προϊόντα αυτά στην καναδική αγορά. Ωστόσο εγώ έχω την πεποίθηση ότι αυτό που κυρίως καλούμαστε να κάνουμε, το πιο κρίσιμο είναι να παρακολουθήσουμε την εκτέλεση των όρων των συμβάσεων εμπορίου που έχουμε συνάψει ήδη σήμερα όσον αφορά την Κολομβία και το Περού. Ε, είμαστε στη φάση αυτή, το κάναμε και με την Κορέα, παρακολουθούμε δηλαδή την εκτέλεση αυτή για να βελτιωθεί ο βαθμός υλοποίησης αυτών των όρων των συμβάσεων αυτές οι συμβάσεις οι οποίες ε, οδηγούν στη δημιουργία των προδιαγραφών για μελλοντικές πολύπλευρες συνεννοήσεις. Να πούμε και για την Ιαπωνία. Το θέμα της Ιαπωνίας είναι πρότυπο, ένα πρότυπο σύγχρονου συμφώνου εμπορικών συναλλαγών με το οποίο καλύπτουμε γύρω στο 1 τρίτο του παγκόσμιου ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, 40% του παγκόσμιου εμπορίου και αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη περί του τι είναι σύγχρονη εμπορική συναλλαγή. Έτσι και όχι μόνο άσκηση ισχύω. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λάγκε. Το βήμα τώρα σε εσάς. Περιμένουμε να ακούσουμε τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Σας υπενθυμίζω ότι έκαστος ή έκαστη έχετε 60 δευτερόλεπτα που πρέπει να τηρήσετε αυστηρά προκειμένου όλοι να μπορέσουν να λάβουν το λόγο. Είχε μεγάλη σημασία να κτηρούμε το χρόνο εδώ. Ισπανία πρώτη, θέση 554. Μανουέλα Λαμπάρ, Φερνάντεθ Καβάλια. εξιότιμη αντιπροσωπή εκπροσωπώ την τέκνικα Ρεουνίδα, ισπανική επιχείρηση που ειδικεύεται στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την ενέργεια. Υπογράφουμε συμβάσει σε όλε τι χώρε του κόσμου, με μηχανικούς και εργαζόμενου διαφορών επικοτήτων, Ευρωπαίου και μη. Είμαστε στου ε, κορυφαίους 10 του κόσμου στον τομέα μα. Με την προοπτική λοιπόν είμαστε υπέρμαχοι ε, απερίφραστα της αλληλεγγύης μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών ε, όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση, την ψηφιοποίηση, τις ελεύθερες και απρόσκοπτες αγορές και μια ε, εμβάθυνση της ε, διεθνούς ε, ένομης τάξης. Είναι αυτές βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μας κάνει δυνατούς. Οτιδήποτε αντιβαίνει στις αξίες αυτές, οτιδήποτε προωθεί εθνικούς εγωισμούς, οτιδήποτε είναι προστατευτισμός, απισχνεί την Ευρώπη, την αποδυναμώνει. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι τι επόμενε εκλογέ του Ευρωκοινοβουλίου έχει μεγάλη σημασία να ψηφίσουμε σωστά. Ελπίζω αυτό το κοινοβούλιο να έχει πολλού φίλο Χρειαζόμαστε περισσότερο άνοιγμα, ε, ε, ε, φιλελευθερισμό, δικαιοσύνη κοινωνική για να μπορέσουμε να προάγουμε την ευημερία του κόσμου μας και να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε το ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με την Τουρκία. 693 Χακάν Ουλικέν. Hello, my name is... Ονομάζομαι Χακάν Χουλκέν, έρχομαι από την Τουρκία. Όσον αφορά την καθήρη εφαρμογή υπάρχουν ιστορικά ε, προσκόμματα όσον αφορά τις τουρκικές ε, μικρομεσαίες ειδικά προκειμένου για συναλλαγές με τους Ευρωπαίους ομολόγους μας ε, Χειριστέ μεταφορές επίσης είναι ένα ζήτημα δύσκολο που θέτει προσκόμματα στην ελεύθερη κίνηση, διακίνηση με των ρευμάτων από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε άραγε κάποια πρόταση για το πώς θα λυθεί το θέμα τη της βίζας για τις μικρομεσαίες και όσον αφορά τις ποσοστώσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με τη Γερμανία. 2-4-0 Wolfgang Γκρένκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, συνέστησα μια επιχείρηση. Τρέγκερ Αγκα είναι κοντά ε, στο Αμβούργο και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Έχει να κάνει με συστήματα leasing και χρηματοοικονομική υποστήριξη μέσα από τραπεζικά προϊόντα και τραπεζικές λύσεις. Ε, κατά συνέπεια είμαστε παρόντες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Θέλουμε να αρθούν όλα τα προσκόμματα για το εμπόριο και για να είμαστε πιο ενταγωνιστικοί αφενός, αλλά και για να έχουμε όσο πιο πολύ κέρδος έχουμε διασφαλισμένο για τους πελάτες μας. Για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοια που να ασκεί διεθνές εμπόριο επί τη βάση κανόνων. Έχουμε ανάγκη λιγότερα προσκόμματα και εμπόδια για το εμπόριο, όχι περισσότερα, όπως επίσης χρειάζεται οπωσδήποτε να αρθούν άλλα εμπορικά ε, προσκόμματα όπως είναι η τελωνικοί δασμοί. Διευκολύνεται το εμπόριο, θα κάνει κάτι η Ευρώπη για μας και κυρίως να αρθούν τα εμπόδια τα οποία τίθενται στις μικρομεσαίες. Έτσι θα μπορέσει να υπάρξει ένα δίκτυο εμπορικό που θα μπορέσει να αντέξει σε οποιαδήποτε προστατευτική προσπάθεια. Ε, η ανταγωνιστικότητα ε, σε ισότιμους όρους δεν πρέπει να υπονομεύεται από εμπόδια που τίθενται μεταξύ άλλων και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ευχαριστώ πολύ. Ιταλία παρακαλούμε. 2.8.0 Μάριο Πότσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ως πρόεδρος ε, της, του Επιμελητηρίου του Βένετο ε, και ως επιχειρηματής σας χαιρετίζω. Θα ήθελα να ενισφέρω στην συζήτηση αυτή με την ιδιότητά μου ως εκπρόσωπος. Βλέπω τα προβλήματα που υπάρχουν σε επίπεδο του εμπορίου και με μεγάλη προσοχή τα προσεγγίζω γιατί το ίδιο με ενδιαφέρουν και δημιουργές ε, συμβάσεις που η Ευρώπη ε, υπογράφει και πόσο δύσκολο αποβαίνει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται και ταυτόχρονα να ακούγεται τη φωνή τους στις διαπραγματεύσεις πόσο μάλλον καθώς πολλές φορές υπάρχει έλλειμμα διαφάνειας. Πρέπει να δούμε τώρα πού είναι η αξία. Προφανώς αυτές οι συμβάσει προσφέρουν δυνατότητες όπως επίσης έχουν και επίπτωση επί του εθνικού ανταγωνισμού. Η έλλειψη πληροφοριών και μέσων ενημέρωσης είναι πρόβλημα στο θέμα αυτό και οι επιχειρηματίες ε, πρέπει να εξοικειωθούν με το νέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα πρέπει να αναπτυχθεί μια λυσίδα αξίας ήδη με αφετηρία το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Διαφορετικά θα πρέπει να υπάρχουν ενδιάμεση, επιπλέον ε, επιμελητήρια κτλ. Αυτό ζητάμε από τους ευρωπαϊκούς φορείς σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Γαλλία, 2.07 η θέση, Jean Χρυσάρ. Καλησπέρα σας, Jean Χρυσάρ από την και Ναζέρ. Ε, είμαι δημιουργό ε, ψηφιακής εταιρεία. εταιρείας. Ε, μια παρατήρηση στα όσα προηγουμένως αναφέρθηκαν. Μπορείτε να στηριχθείτε στα δίκτυα παντού στην Ευρώπη των επιμελητηριών για να υπάρχει ενημέρωση επί των συμφώνων ελεύθερων συναλλαγών. Αυτό εν είδη προκατακτική παρατηρήσεω και το ερώτημά μου. Σε έναν κόσμο που έχουμε απόλυτη ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει βελτίωση του βαθμού της ε, κοινωνικής και κοινοτικής υπευθυνότητας, εταιρικής υπευθυνότητας των ε, εταιριών μας για να μειωθεί η επίπτωση στο περιβάλλον γενικότερα. Δεν πρέπει τα κριτήρια του Εράσμου να ενταχθούν στις δημόσιες προκηρύξεις διαγωνισμών για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Σουηδία 594 Ματς Johansson. κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, μέσα από διάφορες δραστηριότητες παντού να σας πω ότι εδώ και 15 χρόνια εγκαταστάθηκα στη Ρωσία και το προσωπικό μου στην Σουηδία φοβήθηκε μήπως και χαθούν θέσεις εργασίες και όμως σήμερα πολλαπλασιάσαμε τον αριθμό του προσωπικού μας στην ε, Σουηδία 400 άτομα ε, όμως κάτι τέτοιο δεν είναι κάτι που είναι οικονομικό. Χρόνος, χρήμα, προσωπικό, το κόστος αυτό πρέπει σίγουρα να ληφθεί υπόψη. Για το λόγο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε περισσότερες μικρομεσαίες που έχουν την τόλμη να πάνε στο εξωτερικό ακριβώς για να διαδρυνθεί το δίκτυο πωλήσεων μα σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά μα χρειάζεται και ένα οικονομικό σύστημα χρηματοοικονομικό το οποίο λειτουργεί. Οι τράπεζε μα ε, σήμερα δεν μα παρακολουθούν στην πορεία μα αυτή και την προσπάθεια. Ε, οι διάφοροι κανόνε και τα εχέγγυα που μα ζητούν να προσκομίσουμε μα δυσκολεύουν τη ζωή και οι τράπεζε δεν είναι έτοιμε να λάβουν το κίνδυνο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει αυτή την ε, προσπάθεια για εγκατάσταση στην Αλοδαπή και αυτό το άνοιγμα και θηγατρικών όπου μπορούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με την Ουκρανία. 7-04. Τσίσνικοφ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συμμετέχοντες, καταρχήν χαιρετισμού από τον επιχειρηματικό κόσμο της Ουκρανίας. Η Ουκρανία υπέραψε ε, τέσσερα χρόνια πριν μια σύμβαση ελεύθερη συναλλαγή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αποφελή και για τι δύο πλευρέ. Ε, κάποια επιτεύγματα που έχουμε αποκομίσει. Καταρχήν, ε, μεταξύ Ουκρανίας και ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνει το εμπορικό ισοζύγιο με τεράστιες εξαγωγές ε, 25% αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων ε, στην ε, Ουκρανία που εξάγουν πλέον στην Ευρώπη. Και μια πρόταση. Σύντομα, με βάση αυτά θα ήθελα να τονίσω την σημαντική συνεισφορά ε, του, αφού του Σουεδίου ή Ανατολή και Δύση ε, για την εμπλοκή και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στι εμπορικέ αλλαγέ ένθεν και ένθεν. Μα ενδιαφέρει η ανάπτυξη και των ε, πρωτοβουλειών που ήδη έχει αναλάβει το επιμελητήριο στην Ουκρανία. Στηρίζουμε την καθήλη εφαρμογή των όρων των εμπορικών συμφώνων που έχουμε υπογράψει και μας ενδιαφέρει προκειμένου να ανταποκριθούμε και εμείς στην ανάγκη ε, της ευρωπαϊκής αλυσίδας περισσότερη υποστήριξη σε όλους τους τομείς. Χαιρετίζουμε την θέσπιση ε, πιο ευαρύτων εργαλείων προκειμένου για την αντιμετώπιση των ε, ποσοστώσεων και δασμών FTA και τέλος ε, τονίζουμε την σημασία ε, να υπάρχουν ευρωπαϊκά ταμεία ειδικά για τους Ουκρανούς επιχειρηματίες και ελπίζω γενικά για όλους όσους συμμετέχουν στην ε, εταιρική σχέση με την Ανατολή. Να συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε Πορτογαλία 563 Σέρζιου Σίλβα. Εκπροσωπώ τη μεγαλύτερη ιστοποιία στην Πορτογαλία και είμαι πρόεδρος και του Πορτογαλικού Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου ε, Βιετνάμ και Πορτογαλία. Μιλώ για την ε, σύμφωνο εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ένωση και Βιετνάμ. Από το 2015, μετά από 14 κύκλου διαπραγματεύσεων υπεγράφει αυτό, η επιχειρηματική κοινότητα θέλει τώρα πλέον αυτό να εκτελεστεί στην πράξη. Ελπίζουμε πράγματι ότι το FTA θα μπορέσει να τεθεί σε ισχύ όσο νωρίτερα γίνεται. Διαφορετικά, οι ευρωπαϊκέ μικρομεσαίε θα χάνουν κάθε μέρα και πιο πολύ μερίδιο στην αγορά έναντι των απευθεία ανταγωνιστών μα. Ε, πρέπει τις βασικές αξίες να τις δούμε να εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η, στενή συνεργασία με, την, με το ε, Διεθνές Γραφείο Εργασίας και με το Βιετνάμ είναι ένα, κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να το κατοχυρώσουμε και αυτές οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κατοχυρούνται γενικά. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ιρλανδία 446 Paul Nolan. Καλησπέρα σα. Ε, χαίρομαι που είμαι εδώ με του συναδέλφου από τα διάφορα επιμελητήρια. Λέγομαι Πον Νόλαν, είμαι από, τον, από την ομάδα Donmates, οικογενειακή ε, εταιρεία μεταποίηση κρέατο ε, προβάτου και μόσχου. Ε, εξάγουμε σε πάρα πολλούς από τους ε, γείτονες μας στην Ευρώπη. Με υπερηφάνεια είμαστε τμήμα της ψηφιοποιημένης βιομηχανικής οικογένειας της Ιρλανδία, που ε, μεταλαμπαδεύει τα κέρδη τη σε ολόκληρη την κοινότητα, τοπικά και περιφερειακά. Αναγνωρίζουμε την σημασία των εμπορικών συμφωνιών, ειδικά προκειμένου για την άρση οποιονδήποτε δασμολογικών και μη προσκομμάτων. Ε, αναγνωρίζουμε ότι το σύμφωνο με την Ιαπωνία έχει αποδώσει πολύ για τον ο, τομέα των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν πάβουν υπάρχουν και κίνδυνοι για το χώρο της, ε, των τροφίμων, ειδικά σε θέματα ασφάλειας. Καταλαβαίνουμε ότι και η γεωργία πρέπει να είναι κομμάτι τη συμφωνία, αλλά ειδικά για το βόλιο κρέα να είμαστε προσεκτικοί. Ε, πρέπει ε, η πρόσβαση να δίνεται με τρόπο ε, δίκαιο, ακριβοδίκαιο με συγχωρείτε. Πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφέ ισότιμε και ένθεν και ένθεν να τηρούνται οι ίδιε προδιαγραφέ σε επίπεδο αμοιβαιότητα. Πιστεύουμε ότι ε, δεν θα πρέπει να ανεχόμαστε ε, οι αντισυμβαλόμενοι να μην τηρούν του όρου που εμεί τόσο ευλαβικά τηρούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λουξεμβούργο 458. Μόιμπερτο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συμμετέχοντε. καταρχήν θα ήθελα να σα ευχαριστήσω ε, ως, ε, για την πρόσκληση που με έχετε απευθύνει να είμαι εδώ. Το Κοινοβούλιο είναι παρόν και το χαιρετίζω. Αυτή η ευκαιρία Μα δίνουμε την ευκαιρία όλοι να καταλάβουμε τι έκανε και κάνει η Ευρώπη προκειμένου να ενδυναμώσει την ευρωπαϊκή οικονομία και βιομηχανία και ιδίω τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Η εταιρεία μα έχει αναπτύξει τεχνολογία μηχανημάτων συμπιεσμένου αέρα που ενδιαφέρουν όλου ε, για βιομηχανικέ και μη εφαρμογέ, για καθαρή κινητικότητα και για αναπαθήκευση ενέργεια. Το βιομηχανικό μας μοντέλο στηρίζεται στην καθήλη εφαρμογή ενός δικτύου μικροεργοστασίων σε όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μας ενδιαφέρει άμεσα να υπάρχει μια ανοιχτή αγορά. Ως επιχειρηματίας που εστιάζει στην ανάπτυξη αυτής της ε, δραστηριότητάς του, αυτό το δρόμενο του ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου των Επιχειρήσεων μου δίνει την ευκαιρία και να καταλάβω τις δυνατότητες που, παρέχω, που παρέχουν οι συνθήκες που τώρα διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλους μας. Αυτές οι συνθήκες πρέπει να άρουν τα προσκόμματα, ε, τους τελωνικούς δασμούς και να ε, κινητοποιηθεί η όλη δραστηριότητα εφαρμογή των κανόνων. Ε, χάρη, ευχαριστώ το ε, Λουξεμβούργιο Επιμελητήριο για την ευκαιρία που μου παρέσχει να είμαι εδώ κοντά σας σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε. Γερμανία, θέση 300, Μαρκ Σέχακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί επιχειρηματίες και επιχειρηματίες και των δύο γενών. Είμαι ε, πρόεδρος και δηλωθείων σύμβουλος ε, επιχείρησης η οποία μεταπολεί αυτοκίνητα με 70 ε, άτομα στο μισθολογιό μας. Ω πολίτη και επιχειρηματία, ασκώ κριτική απέναντι στο διεθνέ εμπόριο που ασκείται. Είμαστε πραγματικά στον αέρα και αυτό γιατί εξαρτώμαστε από τι κοινοβουλευτικέ εκλογέ του χρόνου που ελπίζουμε να οδηγήσουν σε ένα κοινοβούλιο που θα δείξει σοβαρότητα. Θέλω μια πολιτική σοβαρή ώστε όλοι να μπορέσουν να αποφεληθούν από το πλούτο που ε, δημιουργείται. Ισχύει και τον κόσμο, αλλά ισχύει και την Ευρώπη και βέβαια για τη δική μα συγκυρία για να γιατί όλοι οι πολίτες συνεισφέρουν στη δημιουργία του πλούτου, οπότε εκείνοι πρέπει να απολάβουν πρώτοι τα θετικά αποτελέσματα της παραγωγής και του εμπορίου. Ε, Ιδίω όσον αφορά το χώρο του αυτοκινήτου, πρέπει να δώσουμε προσοχή. Εδώ και τρία χρόνια, ω εμποροί, πραγματικά αντιμετωπίσαμε μεγάλα προβλήματα απέναντι στου πελάτε μα και ιδίω ε, προκειμένου για τι τιμολογιακέ μα πολιτικέ είναι και με τις συμβάσεις που υπογράφουμε με τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων κατήγγυλαν όλες τις συμβάσεις που είχαν υπογράψει με μας και μας επέβαλαν νέες συμβάσεις που είναι λεόντιες, πολύ πιο δεσμευτικές. Μην ξεχνάμε ότι οι πολιτές και οι μεταπολιτές ε, οχημάτων έχουν συγκεκριμένο πρόβλημα ε, έκκληση μην ξεχνάτε επίοικείς και ισότιμους κανόνες για όλους στην Ευρώπη και ειδικά για τους ε, μισθωτούς μας συνεργαζομένους. Ευχαριστώ. Βέλγιο, θέση 33, Μαρκ Βανκύλο. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η εταιρεία μου Hartekan Flanges ε, παρασκευάζει μηχανικά ε, ε, εξαρτήματα για την ε, βιομηχανία. Ως επιχείρηση χαιρόμαστε ιδιαίτερα ε, για τις ε, εμπορικές συμβάσεις που υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτό μας παρέχει εύκολη πρόσβαση στις ξένες αγορές και διασφαλίζεται η συμμόρφωση των ξένων αγορών με τα γενικότερα κριτήρια και προδιαγραφές. Όσον αφορά την παραγωγή μας υπάρχουν διαφορές και μάλιστα οξύνονται. Ένα παράδειγμα, στην Ευρώπη έχουμε πολύ αυστηρό περιβαλλοντικό νομοθετικό πλαίσιο και είναι καλό και ένα πολύ ε, αυστηρό σύστημα κοινωνική ασφάλιση. Όλα αυτά βέβαια σημαίνουν τεράστιο κόστο που φέρουν τα προϊόντα μα. Επί τη ευκαιρία αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουμε δει να έρχονται σοβαρέ επενδύσει στη μεταλλουργία, τι εξορίξει μεταλλευμάτων και τα μηχανικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερώτηση. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντισταθμίσει αυτή την κατάσταση, να αναστρέψει την πορεία και να διασφαλίζει ότι οι νέοι, οι εισερχόμενοι στον χώρο τη παραγωγή αντιμετωπίζουν ίδιο κόστο και ίδιε προδιαγραφέ και κανόνε και μπορούν να τεθούν τα ε, de minimis, όροι αλλά και οι de maximis όροι. Δηλαδή για τα κράτη-μέλη να υπάρχουν τα μέγιστα και τα ελάχιστα με τρόπο ισότιμο για να έχουν όλοι λίγο πολύ το ίδιο πλαίσιο για προδιαγραφές ανταγωνισμού μεταξύ τους. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε τη Δημοκρατία της Τσεχίας. Θέση 39. Τόμας Πλούαρικ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε. Όταν μου ζητήθηκε την πρώτη φορά να σχολιάσω την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, λέω όχι άλλες ρυθμίσεις, ε, όχι άλλη παρέμβαση. Πάντως μετά με διόρθωσα και λέω δημιουργήστε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εποφελές, να επενδύουμε στις μικρομεσαίες. Είναι μια επιλογή για ε, ε, κλιμάκωση. Πρέπει να μοχλεύσουμε τα FTA, πρέπει να φροντίσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις, να τις διευκολύνουμε. Into the, uh, into και σας ζητώ λοιπόν ουσιαστικά να γίνετε λίγο πιο δημιουργικοί. Να γίνετε όπως ε, εμείς καθημερινά πρέπει να είμαστε, δηλαδή δημιουργικοί εμείς στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ιταλία τώρα, 3.37, Φερούτσο Νταρντανέλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα τηρήσω το χρόνο που μου διατίθεται. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ, σε μια Ευρώπη η οποία επενδύει και δημιουργεί αξία. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε περισσότερες ευκαιρίες να συζητάμε τα προβλήματά μας. Ευχαριστώ. Εγώ εκπροσωπώ το οικονομικό σύστημα του Πιεμόντα. Είμαι ο πρόεδρος της ε, Ένωσης αυτής της σημαντικής περιφέρειας στην Ιταλία και το διεθνές εμπόριο μας ε, ε, είναι αυτό που έχει καταστήσει επιτυχημένα τα ευρωπαϊκά κοινωνικά ε, και πολιτικά πρότυπα. Ε, είναι σημαντικές οι διμερείς σχέσεις. Σε αυτή την περίοδο της εμπορικής ενσωμάτωσης, αλλά και σε αυτές τις σημαντικές στιγμές του προστατευτισμού, οι αξίες θα πρέπει να προωθηθούν με αποφασιστικότητα οι εξαγωγές θα είναι το σημαντικότερο κομμάτι των δραστηριοτήτων μας και θα είναι πολύ σημαντικές για την παραγωγικότητά μας. Και στο Πιεμόντε είμαστε δυναμικοί, είμαστε καινοτόμοι, έχουμε τεχνογνωσία η οποία ε, είναι πολύ παλιά, είναι μακριά στο παρελθόν. Ε, και είναι σημαντικό αυτή η αριστεία ε, να προστατεύεται όταν υπογράφουμε διεθνεί εμπορικέ συμφωνίε. Η Ευρώπη πρέπει να καταβάλει μια προσπάθεια προ αυτήν την κατεύθυνση. 2.73 Ελλάδα, ο Παύλο Ραβανής. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ συναδέλφες επιχειρηματίε, αγαπητοί συνάδελφοι επιχειρηματίε, είμαι πρόεδρο του Βιοτεχνικού Μελητηρίου τη Αθήνα. Θεωρούμε ότι τα λιμάνια αποτελούν μια κινητήρια δύναμη τη οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από τα λιμάνια των κρατών μελών της και για το εμπόριο εντός της Ένωσης αλλά και εκτός της Ένωσης. Βάσει της Eurostat το 75% του εξωτερικού εμπορίου γίνεται από τα λιμάνια και το 33% του εσωτερικού εμπορίου. Περισσότερο από 25 σημαντικοί εμπορικοί λιμένες λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τέσσερι από του οποίου έχουν χαρακτηριστική από την Ευρωπαϊκή Ένωση ω λιμένε στρατηγικού ενδιαφέροντο και έχουν ενταχθεί στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών ως βασικές διασυνδέσεις της διόδου Orient East Med. Αυτοί οι τέσσερις ελληνικοί Orient East Med λιμένες είναι τα λιμάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Ιγουμενίτσας και της Πάτρας. Πώς θα ήταν αδυνατόν να αναπτύξουμε και τα άλλα λιμάνια της χώρας της Ελλάδος, αλλά επίσης και της Ιταλίας και των άλλων χωρών που βρίσκονται στη Μεσόγειο, αν ε, θα αποκτήσουν και αυτοί στρατηγικό ενδιαφέρον. Και εκείνο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι κάθε φορά που υπογράφει η Ευρώπη οποιαδήποτε συμφωνία με οποιοδήποτε κράτο θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνε ασφαλεία των εργαζομένων και ιδιαίτερα για το, περιβάλλον, η προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Thank you very much. Romania. Η Ρουμανία 267. Αουρέλιαν Γκουγκουλέσκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι μερικές ιδέες και κάποιες παρατηρήσεις από την πλευρά του Ρουμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες και τη σημασία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και για τον αντίκτυπο στη Ρουμανία και στην Ευρώπη. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι η Ρουμανία βασίζεται κατά 76% στο ενδοκινοτικό εμπόριο και θεωρούμε ιδιαίτερο σημαντικό να υποστηρίξουμε την αντατικοποίηση των διαδικασιών διαπραγματεύσεις ε, στη βάση των ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Αλλά χάρη και στα πολλά ωφέλη που επιφέρουν αυτές τις συμφωνίες. Από τις 600.000 ευρωπαϊκές μικρομεσαίες που εξάγουν και πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο 6.500 είναι ρουμανικές και μόνο ένα μικρό κομμάτι των μικρομεσαίων ουσιαστικά επωφελείται από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ε, διεθνή αγορά. Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει τις σχέσεις της ε, με τις ε, οργανώσεις υποστήριξης, επιχειρηματικής υποστήριξης, έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τον αντίκτυπο αυτών των ε, συμφωνιών. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να τονίσω ότι η προώθηση της ε, διεύρυνσης της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της επίτευξης των ευρωπαϊκών στόχων για την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων και για τη δημιουργία του κατάλληλου νομικού πλαισίου για το νέο επιχειρηματικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Πολωνία, 507. Μάργκο Τζέτα, Κρυσόφσκα. Κυρίες και κύριοι, είμαι δικηγόρος, είμαι ιδρυτικό μέλος μιας ε, δικηγορικής εταιρείας διεθνούς δικαίου. Ε, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε κοινούς στόχους στα πλαίσια της επίτευξης της ε, κοινή εξωτερικής πολιτικής και αυτό βοηθά στην αύξηση της ασφάλειας στα κράτη-μέλη, δημιουργεί την εικόνα μιας ισχυρότερης Ευρώπης με μεγαλύτερη συνοχή και προλαμβάνει βεβαίως διενέξεις και πολέμους ε, μεταξύ των χωρών. Απ' την άλλη πλευρά, υπάρχει ένας πολύ στενός δεσμός μεταξύ της ε, πολιτικής έντασης και της οικονομικής ανάπτυξης. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκείνη η οποία πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο ως προς την προώθηση των εμπορικών και οικονομικών δυνατοτήτων μας στο ε, διεθνές σκηνικό. Μία ε, δραστηριοποίηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δώσει στους επενδυτές μια αίσθηση μεγαλύτερης ασφάλειας και θα βελτιωθεί βεβαίως η οικονομική σταθερότητα. Όσον αφορά τις ε, το διεθνές σκηνικό υπάρχει μια ισχυρή οικονομία ε, που πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας. Σας ζητώ λοιπόν ε, να, βάλετε πάλι την κάρτα σας ε, στο μηχάνημα και περνάμε στην πρώτη ερώτηση, η οποία έχει ως εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει αρκετά προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά τα ευρωπαϊκά, τους κανόνες των ευρωπαϊκών FTA και τις υλοποίησής τους. The vote is... Λήξη της, πληρο... ψηφοφορίας. Ευχαριστούμε. 462 ψήφισαν. 35 είπαν ναι. 376 είπαν όχι. 51 αποχές. Ευχαριστούμε. Ερώτηση 2. Αισθάνεστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ηγετική θέση στο διεθνές ε, στερέωμα έτσι ώστε να βρίσκεται μπροστά στις ανοιχτές αγορές και στο πολυμερές ε, σύστημα εν ώψη ε, πρόσφατων εντάσεων με διεθνείς εταίρους. Ψηφίστε. Thank you very much. Ευχαριστούμε. Λήξη ψηφοφορίας. 462 ψήφισαν. 450 είπαν ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ηγεσία στο Διεθνές Πολυμερές Σύστημα. Ερώτηση 3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ θα πρέπει να ξεκινήσουν εκ νέου αυτές τις διαπραγματεύσεις που αφορούν τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, τα FTA. Ε, ε, άρχεται η ψηφοφορία. you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Λήξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν 463. 391 ναι. Όντω θα πρέπει να ξεκινήσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις. Question number Ερώτηση 4. Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του Brexit δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς της εσωτερικής αγοράς, έστω και αν είναι σε είναι επιβλαβές να ε, συναλλασσόμαστε εμπορικά με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ψηφίστε. Thank you very much. Ευχαριστούμε. Ψήφισαν 473. 411 απάντησαν ναι. 29 είπαν όχι. Last question. Τελευταία ερώτηση, ερώτηση 5. Θεωρείτε ότι η κάθε εμπορική συναλλαγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα ε, σχέδιο δράση υλοποίηση στην Ευρώπη έτσι ώστε να υπάρχει πιο εύκολη συμφωνία και να είναι πιο κοντά στους επιχειρηματίες και στις μικρομεσαίες. Ψηφίστε. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Λήξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν 471. 460 απάντησαν ναι. ναι ευχαριστούμε. Now it is my pleasure. Τώρα με ιδιαίτερη χαρά θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Επίτροπο Εμπορίου, την κυρία Σεσίλια Μόλστρομ. Και είπα στην αρχή θα ακούσουμε μία πρώην δασκάλα, τώρα όμως ακούμε μία συγγραφέα, σωστά. εντάξει, ήμουν και στο Πανεπιστήμιο λέκτορα. Εντάξει, ε, μερικά βιβλία, ναι, αλλά πάει πολύ καιρό. Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Σα ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα εδώ και που μου δίνετε την ευκαιρία να ακούσω κάποιε από τι ε, ενδιαφέρουσε παρεμβάσει. Είναι δουλειά μου να απαντήσω σε κάποιες ε, ερωτήσεις ε, πάνω στι οποίε ψηφίσατε κιόλα και να κάνω και κάποια σχόλια στο πρώτο θέμα, όσον αφορά τι μικρομεσαίε, σαφώ και δεν κάνουμε ποτέ αρκετά. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε να επικεντρωθούμε και αυτό αποτέλεσε μία από τις ε, μεγάλες προτεραιότητες τα τελευταία χρόνια για, το, για την πολιτική εμπορίου, να εστιαστούμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί όπως όλοι το ξέρετε και δεν χρειάζεται να σας πείσω γι' αυτό, εσείς αποτελείτε τη σπονδυλική στήλη τη δική μας. Το 99% των επιχειρήσεων ε, στην Ευρώπη είναι μικρομεσαίες, μη μικρές ή μεσαίες και θέλουμε λοιπόν να σας υποστηρίξουμε, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι εφόσον το επιθυμείτε θα επωφεληθείτε από τις εμπορικέ συμφωνίες τις οποίες διαπραγματευόμαστε. Συνεπώς συμπεριλαμβάνουμε σε πολλές εμπορικέ συμφωνίες κάποια ειδικά κεφάλαια που αφορούν τις ε, μικρομεσαίες, δημιουργούμε ειδικέ ε, ιστοσελίδες, έχουμε ειδικά σημεία επαφής για τις μικρομεσές και προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε με τα διάφορα επιμελητήρια, εθνικά, ευρωπαϊκά, έτσι ώστε να διαδώσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που είναι και πολλές, ε, υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας. Παρ' αυτά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες αυτές τις πληροφορίες απευθύνονται στους τους ανθρώπους, τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν πάντα το χρόνο να αναζητούν αυτές τις πληροφορίες και να τις ανασύρουν. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα σημείο έπαφη, ένα stop shop, στο οποίο θα μπορεί κανεί να βρίσκει όλε τι απαραίτητε πληροφορίε, ε, κανόνε, ε, κανονισμοί, ε, διαδικασίε, α πούμε, για την εμπορική συμφωνία με τον Καναδά. Πριν από, ένα, από μια εβδομάδα πήγα στον Καναδά και συζήτησα και μίλησα με τον Υπουργό και λέω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Αυτό που κάνετε εδώ είναι φανταστικό και η Κομισιόν κάνει πολλά, αλλά η βασική ευθύνη αφορά τα κράτη-μέλη. Πρέπει δηλαδή τα κράτη-μέλη να φροντίζουν ώστε οι εθνικέ επιχειρήσει έχουν πρόσβαση σε όλε τι ε, πληροφορίε, ε, στι διάφορε γλώσσε και τόσο έτσι να διαδίδονται ε, οι πληροφορίε. Εμεί κάνουμε πολλά και φυσικά υπάρχουν και άλλα που πρέπει να γίνουν, ήδη όμω γίνονται αρκετά από την Κομισιόν. Τώρα, στο άλλο θέμα, αν θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ηγετική θέση η Κομισιόν. Χαίρομαι που απαντήσατε ναι. Διαφορετικά θα ήταν δύσκολο για μένα. Να σας πω ότι ο κύριος Λάνιε τόνισε τις διαφορές σε έναν κόσμο που πολλές ε, χώρες αναλαμβάνουν μονομερή δράση, αμφισβητούν το, το, το, το, το, το εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες που έχουμε θεσπίσει εδώ και πολλές δεκαετίες. Ε, τώρα λοιπόν εμείς, ναι, αναλαμβάνουμε ηγετική θέση έτσι ώστε να μεταρρυθμίσουμε ε, τους κανόνες, να, να βγάλουμε νέους κανόνες και να ε, συμφωνήσουμε και, στη, και στους, με τους κανόνες του ε, ΠΟΕ. Το εμπόριο μπορεί να είναι κάτι πολύ καλό και για σας και για εμάς, εφόσον γίνεται με διαφάνεια, με βιώσιμο τρόπο, το εμπόριο είναι κάτι πολύ καλό για τις εταιρείες, για τους καταναλωτές, για τους ε, πολίτες. Και αυτό κάνουμε μέσα από τις διάφορες εμπορικές συμφωνίες μας και προσπαθούμε να αντικατοπτρίσουμε και κάποιες από τις ανησυχίες που ακούστηκαν. Κύριε Πρόεδρε, κάθε εμπορική συμφωνία που έχουμε στο Ευρωπαϊκό ε, και το φροντίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό, είναι πολύ ε, φιλόδοξο όσον αφορά την εμπορική και βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν μιλάμε για κοινωνικά πρότυπα με τους εταίρους, γιατί δεν είναι κοινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν κάποια πρότυπα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους κανονισμούς του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Αυτά φροντίζουμε να τα τηρούμε. Τώρα, όσον αφορά τα, ε, τις συμφωνίες ε, ελεύθερης συναλλαγής, ε, ωραία, αυτό έχει μπει στο ψυγείο λίγο. Δεν έχουμε ακόμα τι προποθέσει για να ξεκινήσουμε ξανά τι διαπραγματεύσει με τη ΣΥΠΑ. Αυτό που είπαμε στη ΣΥΠΑ είναι ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε μία, να φτιάξουμε μία ατζέντα με κάποια θετικά σημεία που θα μα δώσουν μία όθηση. Έχουμε πολλά δηλαδή κοινά. Να ψάξουμε λοιπόν μόνο σε κάποιε μικρότερε ε, συμφωνίε ε, για κάποια βιομηχανικά προϊόντα και εκ παραλίλου σε εθελοντική βάση να δούμε αν μπορούμε να θέσουμε κάποια πρότυπα ε, και να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα που είναι δύσκολα για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν μπορούν εύκολα να τα ξεπεράσουν. Να βασιστούμε σε κάποια από την εμπειρία και τη δουλειά του παρελθόντος και να δούμε αν μπορούμε κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε και πάλι. Ε, είναι συζητήσεις, δεν έχουμε αρχίσει ακόμη διαπραγματεύσεις για τίποτα. Εξάλλου θα χρειαζόμασταν και την εντολή των κρατών μελών για να το κάνουμε αυτό. Αλλά μιλάμε με τη ΣΥΠΑ και να δούμε αν υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε για να διευκολύνουμε το εμπόριο, ε, το οποίο θα είναι επωφελές για αμφότερες πλευρές. Επόμενη ερώτηση στο Brexit. Εδώ νομίζω ότι τα κράτη-μέλη και εμείς ε, ε, επιδείξαμε ισχυρή ενότητα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, έσπασε σε διάφορα κομμάτια, όπως όλοι πίστευαν ε, ότι θα γίνει μετά το δημοψήφισμα. Ο κύριος Μπαγνέο που θα έρθει όπου να είναι, που είναι ο βασικός διαπραγματευτής, νομίζω ότι κάνει ό,τι μπορεί με την ομάδα του έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι έχουμε μια συμφωνία εξόδου και έναν ε, τρόπο συνεργασίας για το μέλλον. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο, αλλά ευελπιστώ ότι σύντομα θα έχουμε σαφέστερο τοπίο και θα διαπραγματευτούμε κάποιο είδος εμπορικής συμφωνίας ανάλογα με τις ε, συνθήκες εξόδου προκειμένου να μην ε, χάσουμε ε, καθόλου από το σημαντικό εμπόριο που έχουμε με τους αγαπητούς φίλους από το Ηνωμένο Βασίλειο, να συνεχίσουμε δηλαδή να έχουμε συνεργασία. Ευελπιστούμε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Τέλος, όσον αφορά το σχέδιο υλοποίησης, η κάθε ξεχωριστή ε, συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ε, δεν είναι κάτι για την οποία ε, θα μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει πώς θα εφαρμοστεί κάθε μία στην κάθε χώρα, στη Σλοβενία, στην Πολωνία ή οπουδήποτε. Κάποιοι έχουν πολύ φιλόδοξα σχέδια. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε να παρακολουθήσουμε την υλοποίηση και εδώ είπαμε και πάλι ότι αυτό θα αποτελέσει προτεραιότητα στο μέλλον, να δούμε δηλαδή πώς υλοποιείται να, δούμε, να βλέπουμε συχνά πυκνά τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά, πώς μπορούμε να λύσουμε κάποια προβλήματα, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με τις μικρές επιχειρήσεις εφόσον είναι απαραίτητο και να έχουμε δηλαδή τακτικές αξιολογήσεις. Θα έχουμε μια ε, καινούρια έκθεση ε, μετά από κανένα δύο εβδομάδες και θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα, θα είναι και online βεβαίως. Θα ε, δούμε όλες τις υπάρχουσες ε, συμφωνίες, πώς γίνονται, πώς εφαρμόζονται, ποια είναι τα προβλήματα, ποια είναι τα πλεονεκτήματα, πώς πάνε τα πράγματα και αυτό μαζί με τη βάση δεδομένων πρόσβασης στην αγορά, να εντοπίσουμε τα μέτρα προστατευτισμού ε, έτσι ώστε να έχετε κι εσείς ένα εργαλείο στα χέρια σας και να το χρησιμοποιείτε. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι απάντησα τις ερωτήσεις ψηφοφορίας και συμπεριλαμβάνω Πάνονται εδώ και κάποια θέματα που έθεσαν οι συνάδελφοι στο ε, κοινό. Δύο-τρία σχόλια σύντομα. Η Κομισιόν την επόμενη εβδομάδα θα υιοθετήσει τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Βιετνάμ και θα στείλουμε κατευθείαν στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την αγγλική έκδοση προκειμένου να ξεκινήσουν οι προετοιμασίε Ελπίζω, αλλά εντάξει δεν είναι στα χέρια μου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο θα κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να υπάρξει μια ομαλή έκβαση αυτής της υπόθεσης ε, και να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία. Στον Ιρλανδό φίλο για το Μερκοσούρ γνωρίζουμε το, το, το, ευαίσθητο κομμάτι που είναι το, ε, το βοδινό. Ε, φυσικά υπάρχει το θέμα της κατανάλωσης κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές, διαπραγματευόμαστε με το Μερκοσούρα, αλλά αν καταφέρουμε να έχουμε συμφωνία μαζί τους, θεωρώ ότι ε, έτσι θα, θα, θα δημιουργήσουμε εξαιρετικές δυνατότητες για τις εταιρείε μας σε όλους τους τομείς, στον αγροτικό τομέα, στις δημόσιες προμήθειες, στις υπηρεσίες, αλλά και, στη, και η, στρατηγική, η στρατηγική σημασία μιας συμφωνίας με αυτές τις χώρες δεν θα πρέπει να υποτιμάται. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν, υπάρχει πολλή χρηματοδότηση, η οποία είναι διαθέσιμη για μικρές εταιρείες, για startups και όλα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σας, πρέπει να σας πω ότι δεν έχουμε κάνει πολλά για να προωθήσουμε την ύπαρξη αυτών των, ε, να κάνουμε γνωστή την ύπαρξη αυτών των ταμείων. Ε, θα έχουμε περισσότερες επενδύσεις ε, την επόμενη περίοδο. Κάποιοι από μπορείτε να ενοχλήσετε και τις κυβερνήσεις σας ε, για να τους επιστήσετε την προσοχή να προσέχουν όταν θα διαπραγματευτούν τον επόμενο ε, προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, υπάρχουν περιορισμοί, αλλά υπάρχουν και δυνατότητες να συνδράμουμε τις μικρές ε, εταιρείε, κυρίως τις νέες εταιρείε, τις start-up και τις πολύ μικρές. Αυτά λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να σχολιάσω, κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και που είχαμε αυτό τον επικοδομητικό διάλογο μεταξύ μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και δεδομένης της αντίδρασης του κοινού ε, άκουσα για την επόμενη εμπορική συμφωνία που θα συναφεί ο Νούπο. Βλέπω ότι όλοι μοιραζόμαστε την αισιοδοξία σας και όντως πιστεύουμε ότι το εμποριο είναι win-win κατάσταση για όλους. Ε, Επικερδής δηλαδή για όλους. Ε, να χειροκροτήσουμε εδώ τους εκπροσώπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. And now we go for our third session. Περνάμε τώρα στην ε, τρίτη συνεδρία. Είναι η συνεδρία που αφορά το μέλλον της Ευρώπης και θα ήθελα εδώ να καλωσορίσω ε, στο πάνελ τους τρεις εισηγητές μας, την Αν Μέτλερ, τον Στίβεν Κλάρκ και τον Βλάντιμιρ ε, Βλάουι. I would like to start with a video for this session. Και θέλω να ξεκινήσω με ένα βίντεο για τη συνεδρία αυτή. Throughout the first half of 2018, the European Parliament led ε, του αιώνα έγιναν συζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ασφάλεια, για το περιβάλλον, για το προσφυγικό. Μοιράστηκαν όλοι τις απόψεις τους σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Μία από αυτές τις προκλήσεις είναι η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης μιλήσανε τα μέλη για κοινέ δράσεις από όλα τα κράτη-μέλη, οικονομικές ε, λοιπόν ε, προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν πιστούν. Το Κοινοβούλιο ε, ψήφισε για τις ε, αγορές online ε, σε διασυνοριακό επίπεδο. Η ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων και αυτό ψηφίστηκε και ο ίδιος μισθός για ίδιες παροχές είναι κάτι το οποίο επιδιώκεται ένεργα, τουλάχιστον 32% τουλάχιστον αυτό θα είναι το ποσοστό της ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο στόχος είναι η χρήση των νέων ε, τεχνολογιών, των έξυπνων τεχνολογιών. Ε, επίσης, καταπολέμηση ε, των περιβαλλοντικών αλλαγών. Έχει αναβαθμιστεί το σύστημα όσον αφορά τις, δια... τις εκπομπές, την αποφυγή εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ενθαρρύνονται επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Το Κοινοβούλιο έθεσε ε, και νέες προτεραιότητες ως προς ε, την ανακύκλωση, ως προς την κατάργηση των χωματερών. Οι νέοι κανόνες ε, θέλουν να μειωθούν τα διατροφικά απόβλητα κατά το ίμιση στο προσεχές μέλλον. Η κυκλική οικονομία, οι έξυπνες πρακτικές, η έρευνα και η καινοτομία είναι βασικές προτεραιότητες. Επίσης, Φροντίζουμε για τη διατροφή, τα τρόφιμα και την ε, γεωργία. Τώρα έχουμε μια καλή ευκαιρία να κάνουμε μια συζήτηση με τον ε, Διευθύντη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για, ε, που ασχολείται ιδιαίτερως με τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια και τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όντως είμαι υπεύθυνο για την υλοποίηση της, της ε, θεσμικής ε, επικοινωνίας όσον αφορά την ε, προεκλογική εκστρατεία για τις επικείμενες εκλογές. Ο Ζαν Κλοντιούλκερ ήρθε κάποτε και μίλησε πρόσφατα και είπε «Αυτή είναι η Κομισιόν της τελευταίας ευκαιρίας». Φαντάζομαι ότι ο καθένας μπορεί να κρίνει το πώς το έζησε και πώς αντιμετώπισε την πρόκληση αυτή η Κομισιόν. Αλλά νομίζω ότι αυτό που τονίζει είναι η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η Ευρώπη σε εκείνη τη φάση και ίσως είναι και ακόμη σε αυτή τη φάση. Ε, ε, κάποιοι σαν και εμένα θα πούν ότι οι επόμενες εκλογές είναι πολύ σημαντικές. Θεωρώ όμως ότι αυτές είναι ιδιαίτερως διαφορετικές και πάρα πολύ σημαντικές. Και αυτό εξαιτία της κατάστασης στην οποία βιώνουμε. Ε, περάσαμε μια δεκαετία κρίσης, πάμε στο 2008, όπου Εκεί ξεκίνησε η δημοσιονομική κρίση. Εν τω μεταξύ είχαμε το θέμα του μεταναστευτικού, του προσφυγικού και ε, βεβαίως αντιμετωπίσαμε και τον Brexit στο μεταξύ. Είμαστε λοιπόν σε μια δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή και η διάθεση του κόσμου δεν είναι πολύ καλή. Είδαμε επίση ε, κατά το ίδιο διάστημα μεγάλε αλλαγέ στην τεχνολογία, στου διάβλου επικοινωνία. Υπήρξε μεγάλη έτσι αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουν την άποψή τους οι πολίτες και κάποια πολιτικά δεδομένα ε, ε, και αυτά άλλαξαν τελείως. Έχουμε νέους παίκτες και αυτοί οι παίκτες συχνά αμφισβητούν πάρα πολλές μορφές πολιτικής ε, συνένεσης. Πολιτικές δομές και διευθετήσεις που υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό έχουν αρχίσει να αμφισβητούνται. Η εδρεωμένη πολιτική και θεσμική δομή και αυτή τίθεται ένα αμφιβόλο. Και ακόμη και η ίδια δημοκρατία, αν θέλετε, τουλάχιστον έτσι όπως εμείς την κατανοούσαμε, σε πολλές περιπτώσεις αυτή τη στιγμή αμφισβητείται και υπάρχει και συγκεκριμένη έρευνα από αυτού. Τώρα, αν εξετάσουμε λιγάκι τα θέματα όπως είναι η απασχόληση, η ανάπτυξη, η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, το εμπόριο, οτιδήποτε. Είναι αυτονόητο ότι όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, ταυτόχρονα υπάρχουν πολλές φωνές οι οποίες αμφισβητούν τις διάφορες δομές που έχουμε δημιουργήσει προκειμένου να διαχειριστούμε την κατάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και όντως θα το έχετε αντιληφθεί ότι μια χώρα αποφάσισε μέχρι και να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα αυτό που λέω λοιπόν σχετικά με τις εκλογές είναι ότι τα διακυβεύματα είναι ιδιαίτερα σοβαρά και ε, τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα σχετικά με το πού γενικώ κατευθύνεται η Ευρώπη, η Ήπειρος, προς τα πού πηγαίνει. Και αυτό το ερώτημα στις συγκεκριμένες εκλογές τίθεται πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, άρα όσον αφορά τις ε, επικείμενες ε, ευρωεκλογέ, σαφώς θέλουμε να υπάρξει μεγάλο ποσοστό συμμετοχή. Είναι σημαντικό οι πολίτε να συμμετάσχουν στις ε, εκλογές, να κατανοήσουν τα διακυβεύματα και εδώ να ακουστεί η πραγματική φωνή των Ευρωπαίων και όχι η πιο δυνατή φωνή που ξέρετε κάνει θόρυβο και ακούγεται. Ακούγεται μέσα στο, στις χαοτικές επικοινωνίες τις οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο η Αρχέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσαν εντολή στη διοίκηση, και εγώ γι' αυτό είμαι εδώ, εκ μέρους τη διαχείριση τη διοίκηση, να ξεκινήσουμε μια εκστρατεία έτσι ώστε να ευνοήσουμε την συμμετοχή στι ευρωεκλογέ. Είπαμε επίση ότι θα πρέπει να έχουμε μια εκστρατεία η οποία θα, θα πρεσβεύει κάποιε αρχέ, όπω είναι η δημοκρατία στην Ευρώπη. Δημοκρατία έτσι όπω την ξέρουμε και έτσι όπω εκπροσωπείται εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο. το οποίο κάνουμε είναι Μία εκστρατεία πολύ απλή. Θέλουμε να προσελκύσουμε κόσμο να ψηφίσει. Θέλουμε κόσμο να ε, συμφωνήσει σε αυτή τη δήλωση που λέμε ότι αυτή τη φορά ψηφίζω. Είναι και η ιστοσελίδα, έτσι. Είναι αυτή, αυτή, ε, αυτή τη φορά ψηφίζω this time I ε, e Η όλη διαδικασία είναι σημαντική. Είμαστε ένας από τους θεσμούς που, ξέρετε, η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μας έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος δεν ακούνε απαραίτητα ανθρώπους σαν και εμένα, αλλά σίγουρα ακούνε ανθρώπους σαν και εσά και ανθρώπους σαν και τους ίδιους. Άρα τι προσπαθούμε να πετύχουμε με την εκστρατεία αυτή, να την διαδώσουμε. Χρειαζόμαστε πολίτες, επιχειρηματίες, ε, ανθρώπους που ασκούν επιρροή, να συμφωνήσουν και να σπαστούν αυτό το θέμα της συμμετοχής έτσι ώστε οι επόμενες ευρωεκλογές που θα ασκήσουν μεγάλη επιρροή στο μέλλον της Ευρώπης να αποτελέσουν ουσιαστικά τη φωνή των Ευρωπαίων γενικά. Χωρίς τη συμμετοχή τη δική σας και τη συμμετοχή άλλων, ε, δηλαδή χωρίς να ευνοήσουμε τη δημοκρατική συμμετοχή, θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα. Διότι σε αυτές τις εκλογές ε, διακυβεύεται και εξαρτάται το μέλλον της Ευρώπης. Thank you very much, Stephen Clark. Ευχαριστούμε πολύ τον Στίβεν Κλάρκ. Όπως είπατε και εσείς, η εκστρατεία ξεκίνησε και όπως σε κάθε εκστρατεία έχουμε και προγράμματα, έχουμε και όραμα και με μεγάλη χαρά θα δώσω το λόγο στον κύριο Βλάντιμιρ Λούι, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ε, Task Force Future of Europe στο Ευρωπημελητήριο, ο οποίος θα μοιραστεί μαζί μα το όραμά του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι η παρέμβαση του ΣΤΙΒ δεν θα μπορούσε να είναι η καλύτερη εισαγωγή για αυτά που θέλω και εγώ να σας μεταφέρω. Όντως, η Ευρώπη βρίσκεται ε, σε μια επικίνδυνη κατάσταση και οι επόμενε ευρωεκλογέ θα είναι ε, μείζονο σημασία. Ακούσαμε εδώ ότι η δημοκρατία η ίδια τίθεται υπό αμφισβήτηση και έχει γίνει λεπτομερής έρευνα επ' αυτού. Μα την έδειξε ο Στίβνο μερικέ εβδομάδε και είδαμε ότι σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε λιγότερο από 40 και 30% των ερωτηθέντων θεώρησαν ότι η, η φιλελεύθερη δημοκρατία είναι ο κατάλληλος τρόπος διακυβέρνηση. Οπότε, από αυτή την έννοια, όντω αντιμετωπίζουμε δυσκολίε και τα διακυβεύματα είναι μεγάλα. Υπάρχει δηλαδή εδώ μια δυσαρέσκεια η οποία αντανακλάται, αλλά εδώ έχω έρθει για να σας πω ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν. Όχι μόνο οι επιχειρήσεις αυτές καθ' αυτές, αλλά κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις είναι πολύ άριθμες. Αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο κομμάτι του ευρωπαϊκού εκλογικού κοινού. Δηλαδή κάποιοι σίγουρα ανήκουν στους δυσαρεστημένους που είναι έτοιμοι ας πούμε, να ψηφίσουν ε, τους λαϊκιστές. Οπότε, αν δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τότε θα συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη βελτίωση των προτύπων ζωής και όχι στην τελμάτωση, όπως πολλοί ε, στην Ευρώπη βίωσαν πρόσφατα. Ε, εδώ θέλουμε να πούμε επίσης ότι η εσωτερική αγορά είναι επιτυχημένη ε, παρά τα ελλείμματα που μπορεί να εντοπίζουμε ενίοτε. Και εντάξει, οι επιχειρήσεις καμιά φορά επικρίνουν αυτά τα ελλείμματα ε, και εδώ τα προβλήματα όντως μερικές φορές είναι πραγματικά. Το Ευρωεπιμελητήριο πάντα υπερασπίζονταν τα συμφέροντα των μελών του έχει δημοσιεύσει μια διακήρυξη των επιχειρηματικών δικαιωμάτων, 12 τέτοια δικαιώματα, τα οποία συνοδεύσαμε με συστάσεις όσον αφορά τις απαιτούμενες πολιτικές για να διασφαλίσουμε αυτά τα δικαιώματα, ότι, γίνονται δηλαδή σεβαστά. Τώρα, πριν από τις εκλογές ε, που είναι τεράστιας ε, σημασίας, το Ευρωεπιμελητήριο αποφάσισε να δημιουργήσει μια επιτροπή για το μέλλον της Ευρώπης που μαζί με το Πιέρ Γκογιάν, το φίλο μου από τη Γαλλία, συμπροεδεύουμε. Αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα position paper σχετικά με το ε, μέλλον της Ευρώπης και να είμαστε σαφείς για ε, όσον αφορά αυτά που σκεφτόμαστε. Θέλουμε ένα μέλλον της Ευρώπης ανοιχτό για τις επιχειρήσεις. Η Ευρώπη έχει πρόβλημα με κρυμμένο προστατευτισμό, με υπερβολικό κανονιστικό πλαίσιο Πρέπει να έχουμε προβλέψιμους και σταθερούς κανόνες. Ζητάμε δηλαδή για ε, μια ισχυρή ε, ενιαία αγορά που θα συνοδευτεί στο μέλλον από την ψηφιοποίηση καθώς επίσης και από κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά τους εμπορικούς εταίρους της Ευρώπης. Ο στόχος δεν είναι να συζητήσουμε το position paper στην ε, σε, με λεπτομέρειες, αλλά θέλουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες το όραμά μας να γίνει σαφές σε όλους τους εμπλεκομένους πριν από τις εκλογές και ευελπιστούμε ότι θα γίνει σαφές και για τη νέα κομισιόν που θα, γίνει μετά, που θα σχηματιστεί μετά από τις εκλογές. Και θέλουμε να υποστηρίξουμε το κατάλληλο περιβάλλον για εσάς, για τους επιχειρηματίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και για τις μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις στον τομέα των υπηρεσιών, διότι πιστεύουμε ότι η ενιαία αγορά, η εσωτερική αγορά που είναι δυνατή, που διέπεται από διαφάνεια, που είναι αποτελεσματική και δίκαιη, είναι το βασικό εργαλείο προκειμένου να αντιπαρέλθουμε την κρίση η οποία φαίνεται ότι ε, σκιάζει, επισκιάζει ακόμη την Ευρώπη. Και τέλος, προετοιμάζοντα αυτό το έγγραφο θέση, το Ευρωεπιμελητήριο σαφέστατα θέλει να δηλώσει ότι θέλει να ακουστεί η φωνή του και ότι θα ακουστεί η φωνή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Δική σε σειρά τώρα, συναδελφοί, να διατυπώσετε προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τον Στίον Κλάρκ και τους ε, συμπροεδεύοντες ε, Βλαντιμίρ Κλουί και Πια Γκογκέ. Ξεκινάμε με την Ιταλία, θέση 382, Αντρέα Τζανλάρη. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους. Ως Πρόεδρος ε, Ερευνητικού Κέντρου στην Πάρμα, θα ήθελα να πω ότι η Ευρώπη είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε ανάπτυξη και μπορούμε να έχουμε φιλοδοξίες. Άρα λοιπόν ε, η διάνοχη της Ευρώπης στον χώρο των τροφιμών είναι απαραίτητη για την επιβίωση της κουλτούρας διατροφής που έχουμε ως πολιτής, πολίτης και ως επιχειρηματίας. Το μήνυμά μου είναι ότι από την Ευρώπη στην ουσία δεν παίρνουμε αυτά που πρέπει να παίρνουμε, δεν παίρνουμε τις ευκαιρίες Δεν έχουμε επίσης δει από πλευρά των Ευρωπαίων ηθινών των αυτοκριτική. Για να υπάρχει ανάπτυξη χρειάζεται καλή επικοινωνία και σίγουρα θα πρέπει οι πολίτες να έχουν επαφή με περιεχόμενο επιστημονικά τεκμεριωμένο πληροφορίες και στοιχεία τέτοια που να μπορούν να τους ενημερώσουν. Ε, η φωνή, μια κοινότητα φωνή. Αυτό είναι που εμείς βλέπουμε και που πρέπει να βρουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Οι πόροι δεν μοιάζουν να είναι πρόβλημα δεδομένου ότι έχουμε διαθέσει τον προπολογισμό. Άρα χρειαζόμαστε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, να κάνουμε μια νέα σκέψη για ολόκληρο τον αγροδιατροφικό τομέα. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλτα 583 η θέση Σιμόντε Τσέζερε. Καλησπέρα σας. Η πρόσφατη οικονομική κρίση έδειξε ότι η σύγκληση που η Ευρώπη επαγγέλλεται έχει ανατραπεί και αναστραφεί. Έχουμε δει τεράστια αύξηση της ανεργίας. Πρέπει να προαγηθηθούν πολιτικές που να αναστρέψουν την λιτότητα. Κάτι που αποτέλεσμα είχε και απαξίωση της ποιότητας ζωής και ε, κακές συνθήκες απασχόλησης. Χρειαζόμαστε λοιπόν καλύτερη συνεργασία για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων που θα μας κάνουν δυνατότερους και πιο ανταγωνιστέ ανταγωνιστικού σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διαδικασία αυτή πρέπει να συνεκτιμά διάφορα πράγματα μεταξύ των οποίων καλύτερη και διαρκή ανάπτυξη και μια καλύτερη διασπορά περιφερειακά των επιχειρήσεων στα κράτη-μέλη. Ο χρόνος έχει σημασία και πρέπει να δράσουμε τώρα προκειμένου για τη σωστή εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα είναι οικονομικέ και όχι επώδυνες και θα σκοπό θα έχουν να αποτρέψουν κρίση στο μέλλον αντί να τι επαναλάβουν. Θέλουμε μια ένωση που να λειτουργεί μέσα από τρόπο ε, διαφανή και με δημοκρατικούς θεσμού με αυξημένη ανταγωνιστικότητα και μια καλύτερη, ένα καλύτερο όραμα για την ανταγωνιστικότητα. Πολλέ και καλύτερε θέσει εργασία, ολοκλήρωση ενιαία αγορά και τη μεγαλύτερο επιτεύγματο τη Ένωση και υλοποίηση των βασικών ελευθεριών ε, σε εμπορικό και αγοραίο επίπεδο, αυτέ τις αγορέ που σίγουρα πρέπει τώρα να κατοχυρούνται. Η Ευρώπη παραμένει ο καλύτερο τόπο για να ζει και να δουλεύει κανεί στον κόσμο, αλλά πρέπει ε, η ευρωπαϊκή διαδικασία να συνεχίσει να καλλιεργείται για να έχουμε και στο μέλλον εγγυημένη ε, πρόοδο και ευημερία. Ευχαριστώ πολύ. Ισπανία, θέση 6-7-3, Χωσέ Λουίς Μπονέ Φερέρ. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Η Ισπανία είναι χώρα βαθιά ε, πεπισμένη για την σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η στήριξη του πολίτη ε, προς ε, το ευρωπαϊκό σχέδιο είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι περίεργο το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισέφερε αποφασιστικά υπέρ της εγκαθίδρυσης της δημοκρατίας και της οικονομίας στην Ισπανία. Η συνεισφορά αυτή από πλευρά των πολιτικών και οικονομικών θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησαν κατά ένα μέρος ε, στην επιτυχία, την θεαματική επιτυχία της πανικής οικονομίας. Ναι μεν, αλλά να αναγνωρίσουμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ζει σήμερα στιγμές αβεβαιότητας. Έχουμε το Brexit, τον προστατευτισμό που απειλεί, καθώς και οι μεταναστευτικές ροές. Μεγάλη πρόκληση αυτές και άλλες. Θέλουμε και πρέπει αυτά τα προβλήματα να ξεπεραστούν γίνεται λόγος για το μοντέλο των 3-3 ε, ταλέντο, εργασία και ε, διεθνισμός. Αυτό σημαίνει ότι θα φτάσουμε αν τα εφαρμόσουμε σε περισσότερη Ευρώπη και πιο πολύ Ευρώπη σημαίνει περισσότερες φιλοδοξίες για το ε, ευρωπαϊκό όραμα, ένα όραμα που πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστικό, ένα ευρωπαϊκό σχέδιο πιο εξυγχρονιστικό, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που σίγουρα θα είναι αλληλέγγυο και τέλος ένα ευρωπαϊκό σχέδιο που θα μας οδηγήσει στο μέλλον τις ευημερίες των Ευρωπαίων. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Σερβία 765 Στράβκο Ιλίτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως Σέρβος πολίτης είναι κάπως παράξενο να μιλώ στο χώρο αυτό. Δεν παραδέχομαι, αλλά ως ε, εκπρόσωπο του σερβικού επιχειρηματικού κόσμου, τι το πιο φυσικό. Όταν εμπορευόμαστε με την Ευρώπη, εμπορευόμαστε. Όταν κάποιο επενδύει σε εμά, η Ευρώπη επενδύει πάντα σε εμά οι μεγαλύτερε οδικέ αρτηρίες, οι μεγαλύτεροι ποταμοί, όλα αυτά εντάσσονται σε εμά στο ευρύτερο σύστημα ευρωπαϊκών διαδρόμων. Τόσο είναι οι δεσμοί, ώστε και η μοίρα μα μας αλληλένδετη με εσά όταν περνάτε κρίση, περνάμε και κρίση και εμεί και αντίτροφα. Και όταν αναπτυσσόμεθα, ένθεν και θα αναπτυσσόμεθα. Το μέλλον της Ευρώπης είναι ο δικό μας μέλλον. Για το λόγο αυτό, για μας, η ένταξη στην Ένωση για τις επιχειρήσεις ε, στη Σερβία είναι ζωτική σημασία. Ε, από την ιστορία διδασκόμαστε και πιστεύουμε ότι το ίδιο σημαντικό και για εσά, γιατί είναι μια στρατηγική όπου όλοι κερδίζουν. Και εσείς ε, και από την εμπειρία σα έχει καταδειχθεί ότι η διεύρυνση τη Ένωση αποτελεί πραγματικά σενάριο στο οποίο όλοι κερδίζουν. Σήμερα ε, θέλουμε να μα υποστηρίξει γιατί πιστεύουμε ότι η κυβέρνησή μα και οι θεσμοί ε, στην Ευρώπη ξέρουν τι θέλουμε και τι χρειαζόμαστε. Θέλουμε η φωνή να ακουστεί πιο ε, στεναρά και να σταλεί το μήνυμα ότι η διεύνηση χρειάζεται και το μέλλον της Ευρώπης είναι περισσότερη η Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γερμανία 1-1-4. Ελίχιατ Βέμπα. Λέγομαι Ρίχιατ Βέμπερ. Προέρχομαι από την περιοχή της Ζάρ. Παράγουμε μπύρα και ποτά με βάση την μπύρα. Είμαστε παρόντες σε έξι διαφορετικές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν, είναι και παραμένει σημαντική για μας και τις επιχειρήσεις μας, ιδίως προκειμένου για τις υπηρεσίες που παρέχονται διασυνοριακά είναι εξαιρετική σημασία και αυτό διότι πρέπει να είμαστε σε θέση να δουλέψουμε με τρόπο εύκολο και ευέλικτο διοικητικά και γλωσσικά μιλώντας. Και αν πραγματικά θα μπορούσαμε να δουλέψουμε και στη δική μας γλώσσα σε άλλες χώρες, ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Και βέβαια η σχέση με τις γειτονικές χώρες είναι για μας μεγάλη σημασία και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενο που ακούω και ότι οι Σέρβοι ε, πήραν το λόγο και είπαν ότι είπαν σημαντικό να του έχουμε κοντά μα σήμερα γιατί και εμεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουμε να δώσουμε μια προοπτική τέτοια που να του βοηθήσει να καταλάβουν σαφώ ότι είναι κομμάτι τη ε, ε, Ευρώπη. Δεν θέλουμε. Ξέρετε, να έχουμε άλλες δυνάμεις από την Ανατολή. Η Κομισιόν πρέπει να δημιουργήσει την εσωτερική αγορά και να αποτελέσει αυτή το δυνατό σημείο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να εντατικοποιήσει του στενού δεσμού με του κοντινού μας γείτονε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από την Εσθονία, ο Κάουρο Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το, μέλλον της Ευρώπης κινείται αργά, αλλά μέχρι να τα συζητήσουμε, δηλαδή εδώ ο κόσμος έχει προχωρήσει. Υπάρχουν επικείμενες εκλογές, έτσι, ας τις περιμένουμε. Μήπως πρέπει να πάρουμε μια απόσταση και να περιμένουμε τα καλύτερα να συμβούν. Διότι πολλές φορές τρέχουμε από πίσω να προλάβουμε τις αλλαγές. Οι αντιδράση των νομοθετών πολλές φορές είναι αργοπορημένες και ε, βεβαίως έτσι εμποδίζουν τη δυνατότητά μας για καινοτομία. Πάνε χέρι -χέρι με τις Πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι με τις αναδυόμενε τεχνολογίες και με το ε, μέλλον, γιατί το μέλλον δεν μας περιμένει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η Γαλλία. Θέση 256. πια Η Ευρώπη είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, το ξέρουμε όλοι αυτό. Και σίγουρα οι γαλλικές επιχειρήσεις ε, είναι δεσμευμένες σε ένα πρόγραμμα διαβούλευσης με τους πολίτε γύρω από το μέλλον της Ευρώπης. Πάνω από 35 κύκλοι διαβούλευση έχουν διοργανωθεί από όλα τα γαλλικά επιμελητήρια, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Και αυτό επιτρέπει σήμερα πλέον να έχουμε μια πρώτη αποκατάσταση αυτού που οι επιχειρηματίε επιτόπου, οι νέοι ε, θέλουν και περιμένουν. Έχουμε μια πρώτη εικόνα. Τέσσερα μηνύματα έχω να καταγράψω. Φέρουν μια Ευρώπη της κινητικότητας για τους μαθητευόμενους, για τους σπουδαστέ και τους ε, μισθωτούς, ιδίως σε διασυριακές ζώνες την Ευρώπη της καινοτομίας με βιομηχανικά ευρωπαϊκά προγράμματα πιο ευπρόσβατα για τις μικρομεσαίες. Μια Ευρώπη πιο δεδηλωμένη και πιο ταγμένη στην αηφόρο ανάπτυξη που τις μεγάλες απαιτήσει της ε, μεταφράζει σε ευκαιρίες και ανταγωνιστικά προτερήματα. Και τέλος μια Ευρώπη εναρμονισμένη, θεμελιούμενη σε κοινωνική σύγκληση, δημοσιονομική σύγκληση, έτσι ώστε όλες οι επιχειρήσεις να μπορούν να ε, δραστηριοποιούνται με τους ίδιους κανόνες. Ε, από τα μηνύματα όλων αυτά είναι διαθέσιμα επιγραμμικά και έχουμε και ένα εθνικό αποθετήριο ε, δηλώσεων στη Γαλλία που θα είναι έτοιμα τις επόμενες εβδομάδες και θα σας ενημερώσουμε αργότερα. Ευχαριστώ πολύ. Turkey. Τουρκία 698 Μουλκιέ Αϊτά Καλησπέρα σας. Είμαι η Μουλκιέ Αϊτάρα από την Τουρκία η τρέχουσα θεώρηση των πολιτικών και στην Ευρώπη και ειδικά το θέματα της, ε, των, των πολιτικών γειτονία είναι που οδηγούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την εταιρική της σχέση ανά τον κόσμο και να αναζητήσει νέες ε, συμμαχίες. Κατά συνέπεια, χαιρετίζουμε την πρόσφατη πρωτοβουλία ε, στον χώρο των Δυτικών Βαλκανίων ε, δεδομένου ότι μας δίνει μια επιπλέον νέα ε, για τα Βαλκάνια θεωρούμε ότι οι βαλκανικές χώρες θα πρέπει να γίνουν όλες μέρη της Ένωσης. Παρά τα αυτά, θα ήθελα να υπογραμμίσω όλος ιδιαίτερα το γεγονό ότι η Τουρκία αποκλείεται από την πολιτική διεύρυνση και αυτό δεν είναι παραδεκτό, δεν είναι αποδεκτό. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι το εξή. Εν ώψη των νέων δυναμικών του διεθνού συστήματος βάσει του οποίου η Τουρκία αποκλείεται από την πολιτική διεύρυνση μήπως τελικά θα είναι από μόνο του ένα μεγάλο λάθος ή θα είναι μόνο πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι πιστεύετε. Thank you very much. Ευχαριστούμε. Βέλγιο. 64. Μπέρτ Ούγκο. Το ακούσαμε σήμερα κύριε Πρόεδρε ότι η ολοκλήρωση είναι και πρόκληση αλλά και μια πραγματικότητα πολύ συγκεκριμένη. Η ένταξη των ενέων στην χώρα των μεταναστών, στα διάφορα τη Ένωση κτλ. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν ε, τα διάφορα θρησκεύματα και οι κουλτούρες δημιουργούν πρόσκομα στην καλή ολοκλήρωση διότι για συστήματα αξιών, σημαντικών αξιών για καθέναν μας. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει πραγματικά να παίξει το ρόλο ε, του συγκεραστεί. Εάν δεν, δεν θέλουμε να μείνει χώρος για τους λαϊκιστές και τους εθνικιστές. Εξού και το ερώτημα, μήπως τελικά ήρθε ο χρόνος να γίνει ουσιαστικός διάλογος επί των αξιών. Ε, δεν αρκεί μια καμπάνια αξιών. Ε, πρέπει να συζητήσουμε τις αξίες με το κοινό των πολιτών και με τα επιμελητήρια για να ξέρουμε τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θέση θα πάρει στο μέλλον. Διαφορετικά ε, ρισκάρουμε ο πληθυσμό τη Ένωση να απομακρυνθεί και μέχρι τώρα τα αποτελέσματα των εκλογών είναι καταστροφικά. Έχω κατά νου τη Σουηδία αλλά και στην Ιταλία. Προσοχή, αν, ε, προσοχή τι θα κάνουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ελλάδα 3-2-7 Στέφανος Γεωργιάδη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι επιχειρηματία στον χώρο Παραγωγή ενέργεια από ανανεώσιμε πηγέ, Είμαι αντιπρόεδρο στην Ένωση Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιοχών και πρόεδρο του Μελιτηρίου Δράμα, καθώ και μέλο τη Δίκη Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδο. Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση διανύει μια κρίσιμη περίοδο αναζήτηση ταυτότητα και προσανατολισμού που ίσω δεν έχει προηγούμενο. Μετά την εφορία τη δεκαετία του 1980, με την ολοκλήρωση τη ενιαία εσωτερική αγορά και τη δεκαετία του 1990, με την επίτευξη τη νομισματική ένωση, το ευρωπαϊκό εγχείρημα δείχνει να έχει χάσει το δυναμισμό και τον προσανατολισμό του η αισιοδοξία ότι η σημερινή κρίση μπορεί να ξεπεραστεί δεν είναι κατάλληλη στάση για να συμβάλλει κανείς στην υπέρβασή της. αντίθετα ο προβληματισμός για το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι απολύτως αναγκαίος γιατί το μέλλον του ευρωπαϊκού οικοδομήματος μοιάζει σήμερα περισσότερο αβέβαιο από ποτέ. μήπως θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην κοινωνική συνοχή των κρατών μελών και να μην μπαίνουν σε προτεραιότητα ατομικές πολιτικές όταν τα συμφέροντα των σημαντικότερων χωρών μελών της ένωσης αποκλίνουν συστηματικά; μήπως οι καλές πρακτικές πρέπει να έχουν προτεραιότητα στις συνοριακές περιοχές με αποκεντρωμένες πολιτικές αυξημένης χρηματοδότησης ώστε τα σύνορα μεταξύ των κρατών μελών καθώς και τα εξωτερικά σύνορα να καταστούν χώρος ανάπτυξης δημιουργίας καινοτομία και πολιτισμού; ευχαριστώ. Thank you very much. Εμείς ευχαριστούμε. Ιταλία, 438 Γκλωριάνου Λαντσότη. Είμαι ο Γκλωριάνου Λαντσότη, πρόεδρος ε, του επιμελητηρίου του Τρεμόνο. Κύριε Πρόεδρε, προ, ε, φίλοι συναδελφοί, το μέλλον της Ευρώπης δείχνει να είναι οξύμορο. Το λέω γιατί πρέπει σίγουρα να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα και την ευκαιρία που μας παρέχεται να την ε, μετατρέψουμε σε μήνυμα αλλαγή. Οι κανόνε ε, τη Ευρώπη επηρεάζουν την καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, διαπιστώνω ότι πίσω από κάθε απόφαση για το μέλλον τη Ευρώπη υπάρχει πάντοτε μια αντιπαράθεση δύο αποκλίνουσων σχέσεων που δύσκολα γεφυρώνονται. Η αποδυνάμωση των ε, Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων Ιδίω Κομισιών και Κοινοβουλίου μα καταπλήσει, είναι καταφανή. Και απ' την άλλη, το λέμε ότι στην Ευρώπη θέλουμε θεσμού ευρωπαϊκού, σε επιχειρήσει και αρμοδιότητε ε, που να θα ενισχυθούν πρέπει να σκεφτούμε με προσοχή ποιε είναι οι μελλοντικέ φιλοδοξίε μα και να καταστήσουμε την Ευρώπη ένα συντελεστή που πραγματικά θα είναι ικανό να είναι ηγέτη των ε, εξελίξεων στην περιοχή μα, γιατί ε, η περιοχή μα είναι κρίσιμη συνεργασία για όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Η Ρουμανία 638 Αλεξάνδρου Τσόκαν. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε Είμαι Ρουμάνος επιχειρηματίας και σπουδαστή που αποφάσισε να ζήσει στο εξωτερικό και να μελετήσει στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι κοινότυπο, όχι μόνο στη χώρα μου, αλλά και σε άλλε νοτιοευρωπαϊκέ χώρε. Και είμαι ευγνώμων για το ότι μπορώ να συνδέομαι και να μαθαίνω από του ευφυεί τη Ευρώπη ε, δεν νομίζω ότι θα λυπήθηκα που έφυγα από τη χώρα μου. Το ταλέντο που ε, χρειά Ρουμανία για να έχει μέλλον επιλέγει το εξωτερικό για να βρει το δρόμο και να μπορέσει ίσως να γυρίσει πίσω με κάτι καλύτερο. Ε, δεν νομίζω ότι αυτό όμως θα ισχύσει για όλους. Για μένα το μέλλον της Ευρώπης δεν είναι μόνο ο αγωγός που θα δώσει ελεύθερο εμπόριο, ε, θέσεις και ενημέρωση, αλλά και μια ευκαιρία επιχειρηματικότητας για τους νέους στις χώρε προέλευσή τους. Πρέπει για να γίνει αυτό να έχουμε πρόσβαση σε καλύτερη χρηματοδότηση, να υπάρχει ενημέρωση για ευκαιρίε χρηματοδότηση για τι ε, νεοφυεί επιχειρήσει. Μην ξεχνάμε τα θέματα κατάρτιση και ε, επιμόρφωση. Άκουσα με ενδιαφέρον Ρωμάνου αδελφού να μιλούν για ένα διευρωπαϊκό σύστημα μέσα από το οποίο οι εταιρείε θα υποφελούνται φορολογικών ελαφρύσεων και κινήτρων για να μπορούν να απασχολούν εγχώριου ε, φοιτητέ και να αποτρέψουν τη φυγή στο εξωτερικό. Ευχαριστώ πολύ. Εμεί ευχαριστούμε. Σουηδία. 536 Στέφαν Μούσλα Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ευχαίρεια που μου παρέχετε να μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έστω και για 60 δευτερόλεπτα. Να χωρέσει εκεί το μέλλον μου πρέπει στα 60 δευτερόλεπτα. Εάν το ευρωπαϊκό σχέδιο το δούμε σαν προϊόν, ε, θα ήταν κάτι εξαιρετικό και όλοι θα ήξεραν τι να κάνουν και θα το πετύχαιναν. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι δεν το βλέπει έτσι το κοινό. Και για ποιο λόγο η κοινή γνώμη δεν το βλέπει. Νομίζω ένα από του λόγου είναι ότι δεν μπορέσαμε ε, ή δεν πετύχαμε αρκετά να προωθήσουμε το προϊόν μα και να πείσουμε τον κόσμο για την επιτυχία που θέλουμε να πετύχουμε. Τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον λοιπόν είναι να μπορέσουμε να προωθήσουμε διαφημιστικά και να κοινοποιήσουμε το μήνυμα αυτό, να πείσουμε για την ποιότητα του οράματό μα και ότι όλοι θα αποφεληθούν ε, και ότι όλοι θα μπορέσουν να είναι κοινωνίες στην ευημερία. Γι' αυτό ε, ζητώ από τους πολιτικούς να μην ε, βρίσκουν δικαιολογίε για να δημιουργούν ε, προγράμματα λιτότητας εσωτερικά, αλλά να πείσουν την χώρα και τον κόσμο. Είμαι Σουηδό. αυστηρός στον χρόνο και δεν τον υπερβαίνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. 521. 2 Ρομπέρτ Σεσπιολέτσι. Σεσπολέτσι. Διόρθωσε τον ομιλητή. Σχεδόν το είπα σωστά, λέει ο Πρόεδρος. Ε, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, άκουσα μια σειρά από βραχεία ε, ερωτήματα στην Αγγλική, αλλά παρακολουθώντας τη συζήτηση αυτή, θυμήθηκα ότι υπήρχε κάποτε εδώ κάποιος στο, στο ε, ακροατήριο που ήδη από την δεκαετία του 80 εστιαζόταν σε εργαλεία και σε μηχανισμούς, σε μηχανισμούς μέσα των οποίων θα δραστηριοποιούμασταν. Ε, η δική μου επιχείρηση έχει δύο άτομα προσωπικό, αλλά στην Πολωνία και άλλους 50 διασπαρμένους σε πάνω από 14 χώρες ε, στην Ευρώπη. Ε, εταιρεία πληροφορική είναι η επιχείρησή μου που συναλλάσσεται επιχειρηματικά με την Τουρκία και τη Σερβία. Τώρα, εάν μου επιτρέπετε, ε, δύο-τρία στοιχεία που έχουν μεγάλη σημασία νομίζω, γιατί στοχεύουν τόσο έπατα και είναι τροφή και σκέψη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διαφρόγαρα. Το 2006 ε, η οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών ε, τέθηκε σε ισχύ εναρμονίζουσα το 45% των ε, υπηρεσιών. Πάμε ένα βήμα παραπέρα λοιπόν τώρα πάνω από 50% ε, των, υπηρεσιών στην Ευρώπη παίρνουν να εναρμονιστούν για να υπάρχει πραγματική ελεύθερη ροή των υπηρεσιών. Και κάτι ακόμα θα πρέπει να αναλογιστούμε πώς θα μπορούσαμε ενδεχομένως να επιταχύνουμε την εναρμόνιση ε, της φορολογίας και αυτό να αφορά όλη την Ευρώπη. Γιατί ξέρετε ότι Πολλέ επιχειρήσεις αναγκάζονται να εγκατασταθούν στις ΗΠΑ. Ε, υπάρχουν διάφορες καταστάσεις που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μέσα από καταστάσεις. Η ενερμόνιση της φορολογίας έχει μάλιστα και κάτι ακόμα. Ε, υπό την επόμενη ε, χρηματοοικονομική προοπτική θα πρέπει να έχουμε γραμμή στον προπολογισμό ειδικά μεταξύ κρατών της Ένωσης Ειδικά ε, χώρε οι οποίες ε, έχουν μεταναστευτικέ ροέ είναι και χώρε πρόληψης μεταναστών. Κάποιοι. Yeah, thank you. Ε, νομίζω ότι ε, το οφείλουμε αυτό στου μεταναστέ. Now we continue with uh, German. Ε, συνεχίζουμε τη Γερμανία 3-4-4. Χριστίνα Λούτκε. Yes, Mr. President. Ladies. Ναι, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, ε, Είμαι πρόεδρος ε, του Γερμανικού Φορέα Ένωσης των ε, Μελτηρίων. Ε, έχω, είμαι επικεφαλής της τοπικής ε, αντιπροσωπείας της ΚΙΑ. Μικρή, αλλά θαυματουργή όπως λέμε, έντονα ρυθμισμένος ο τομέας. Επιτυχημένος επιχειρηματές είναι εκείνο που κάνει την ιδέα πραγματικότητα και επιτυχής διακυβερνητικό ή διεθνής οργανισμό, είναι εκείνο που δίνει προστιθέμενη αξία στα μέλη του. Οι νέοι επιχειρηματίε θα πρέπει να βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ω ένα θεσμικό φορέα που παρέχει ευκαιρίε για το επιχειρήν και όχι ω φορέα που σου αναστέλει την διάθεσή σου να διοικεί μια επιχείρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει ενδυναμωτής και όχι πρόσκομα. Ε, για τις νεοφυείς, για τις οικογενειακές, μικρομεσές και όλους αυτούς ε, χρειαζόμαστε όλοι μια νέα ευελιξία και όλο αυτό θα είναι δοκιμή για το μέλλον. Θέλουμε νέου κανόνε και πρέπει να ενθουσιάσουμε του νέου για την ευρωπαϊκή ιδέα και να προάγουμε το επιχειρηματικό πνεύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δίνει το ρυθμό για την ηλεκτρονική και διακυβέρνηση και περαιτέρω να προάγει την εκπαίδευση των επιχειρηματιών. Είναι μεγάλε αυτέ προκλήσει και πρέπει να τι αντιμετωπίσουμε. Σα ενθαρρύνω να ξεκλειδώσετε το δυναμικό των οικονομιών σα με το να ξεκλειδώσετε το πνεύμα των επιχειρηματιών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Αλβανία 7-7-1 Ήλι Μπράκα. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και κάποιες φορές να καταλάβουμε εμένα και τους δε όλη την ημέρα σήμερα παρακολούθησα όλους όσους πήραν το βήμα, όλους τους συναδέλφους να έρχονται εδώ και να καταθέτουν προβλήματα. Πολλά προβλήματα ε, να καταθέτουν την εμπειρία τους. Αλλά η εμπειρία αυτή μας βοηθεί να είμαστε μια ομάδα, ένα σώμα. Και για να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου, Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει υπόψη του όλα τα προβλήματα που κατέθεσαν εδώ οι συνάδελφοι. Είμαστε συντελεστέ σε αυτή τη διαδικασία. Όλοι συνεισφέρουμε σε αυτήν. Και ξέρουμε ότι πίσω από εμά υπάρχουν πολλοί που περιμένουν από εμά να προχωρήσουμε. Κάθε φορά χρειαζόμαστε πρόγραμμα. Πρόγραμμα που σημαίνει ώρες και ώρες δουλειάς. Ώρες και ώρες δουλειά ανθρώπων επιχειρήσεων, ενώσεων, χωρών Κοιτούμε λοιπόν ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την θεωρούμε ένα μεγάλο σπίτι για μας και μια υπόσχεση. Για το λόγο λοιπόν αυτό και για να μπορέσουμε λοιπόν να δώσουμε ένα βήμα στο οποίο εισακούγονται τα ζητήματα για την Ευρώπη πρέπει καταρχήν να καταλάβουμε ποιοι είναι οι βασικοί συντελεστές ε, ποιοι είναι αυτοί που θα παίξουν το βασικότερο ρόλο για το μέλλον αυτό. Και ένας από αυτούς τους συντελεστές, όπως το έχετε προτείνει, νομίζω ότι όλο αυτό είναι μεγάλη δοκιμασία αλλά και μεγάλο, μεγάλη πρόκληση για σας. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Η ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορεί να κάνει τίποτα από μόνη της Γι' αυτό και θα ήθελα να αναφέρω στη μνήμη σας τρία βασικά ζητήματα. Λυζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, πρέπει να σας διακόψω γιατί δεν έχετε χρόνο. Περνάμε στον επόμενο μιλήτη. We continue with number seven. Αριθμός 773. Πάμπελ Ραντοβάνοβιτς. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μια κάποια προοπτική ιδιότητα μέλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλη σημασία ε, ένα ζήτημα μεγάλη σημασία για την οικονομία του Μαυροβουνίου και των γειτονικών χωρών. Η διάνοιξη ε, επιμέρους κεφαλαίων έχει μεγάλη σημασία για την καλή διαδικασία ένταξης και επιβεβαίωση του ότι το Μαυροβούνιο είναι μια προοδευτική και σταθερή χώρα. Αξίζει το Μαυροβούνιο να αξιοποιήσει σωστά τι ευκαιρίε που του παρέχονται για να γίνει κομμάτι τη κοινή ευρωπαϊκή αγορά. Έχουμε την ικανότητα να είμαστε αξιόπιστο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα δεν είναι λόγο για αναβολή Τη διαδικασία διεύρυνσης γιατί η αντίδραση του Μαυροβουνίου και άλλων κρατών της περιοχής απέναντι στην οικονομική κρίση και τη μετανάστευση αποδεικνύει ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε ουσιαστικά στην επίτευξη ευρωπαϊκών στόχων. Η διαδικασία διεύρυνσης ε, είναι προ το συμφέρον όλων των Ευρωπαίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ε, χώρες της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης ε, είναι κομμάτι ενό ολοκληρωμένου σχεδίου. Προσοχή στην τήρηση των αρχών όμω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Γαλλία, αριθμός 312, Φανή Ρουίνα. Φανή Ρουίνα. ε, έχω συστήσει την επιχείρηση Φανή Στυλ Χάλιβα στην Πικαρδία και πρόεδρο ε, του ομιλού ε, Φλάν. Ως επικεφαλής επιχείρησης δημιουργούμε θέσεις εργασία και αναπτύσσουμε την οικονομία. Παρά τα αυτά, το 52% του πληθυσμού ε, είναι μόνο 30% ε, ε, επικεφαλής επιχειρήσεων. Ως γυναίκα μιλώ, αλλά και ως συντελεστής της οικονομίας ζυγίζω καλά τα λόγια μου. Δεν εκπροσωπούμαστε αρκετά και αυτό είναι βλάβη για την οικονομία της Ευρώπης. Οι αρμόδιοι λήψη αποφάσεων στην Ευρώπη πρέπει να απελευθερώσουν αυτή τη δυνατότητα. Οι πολιτικοί δεν πρέπει να προσπαθούν να παμβλύνουν όλε τι διαφορέ. Δεν γίνεται αυτό, το καταλαβαίνουμε. Αλλά η διαφορετικότητα, η συμπληρωματικότητά μα είναι αυτό που μα ενώνει και μα δίνει δύναμη. Και δεν μιλάμε μόνο ε, σε επίπεδο φύλου. Εδώ δουλεύοντα σε επίπεδο επικοινωνικού συστήματο έχει μεγάλη σημασία. Α δώσουμε επιθυμία για δημιουργία να μην περιοριζόμαστε, ιδίω όσον αφορά τον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα, του ανθρώπους. Πρέπει να παράσουμε τα χέγγυα για πολιτικές δημιουργίες οικογενειών, δημοσιονομικές και άλλες πολιτικές χωρίς διακρίσεις. Εμείς οι επικεφαλής επιχειρήσεων εκλεγμένοι και εμείς θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα για τη δημιουργία επιτυχίας που θα είναι παράδειγμα. Έχουμε ρόλο να παίξουμε. Ας μοιραστούμε καλές πρακτικές μέσω των εμπορικών επιμελητηρίων. Ας δώσουμε επιθυμία. Η Ευρώπη είναι υπέροχη ευκαιρία για όλους και όλες. Ας αναπτύξουμε από κοινού τις δυνατότητές μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Εμείς ευχαριστούμε. Ουκρανία, αριθμός 703, Βαρετίνα Σουρτικόβα Γκέπνα. Καλησπέρα σας. Εκπροσωπώ το Ουκρανικό Εμπορικό και Μηχανικό Επιμελητήριο Σέβομαι τη ρίζα μου που είναι γερμανική, γι' αυτό και θα ήθελα να συνεχίσω τη γερμανική γλώσσα, λέει ο μιλήτρια. Ε, κατά τον τρέχοντα μήνα και μέχρι το Μάρτιο του 19 οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποφασίσουν ε, σχετικά με το ποιος θα τους εκπροσωπήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε 27 χώρες και στη συνέχεια θα αποφασίσουν για τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ποια είναι η Ευρώπη των Ευρωπαίων πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προφανώς είναι στην καρδιά της συζήτηση αυτής. Τελικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να καταστεί ένας, ε, μια ευρωπαϊκή περιφέρεια ή αν θέλετε πολυομοσπονδικό κράτος όπως είναι η αν θελετε πολυ ομοσπονδικο κρατος οπως ειναι η ελβετια οι Ηνωμένες Πολιτείες ή ενδεχομένως μια Ευρώπη των διαφόρων ε, κρατών που και εθνών ε, που συνδέονται μέσω ενός κοινού συντάγματος τέλος πάντων ή συνθήκων. Εμείς έχουμε την εξής ερώτηση. Πότε θα μπορέσει πραγματικά η Ουκρανία να αποκτήσει σαφή και περίφραστη ένταξη ε, όπως οι υπόλοιπες βαλκανικές χώρες ε, των Δυτικών Βαλκανίων. Πόσο χρόνο ακόμα θα θεωρούμε, θα θα απλά μια γειτονική χώρα το Εμπορικό Επιμελητήριο ελπίζει να έχουμε μια θετική απάντηση συντόμω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. From Ireland, number 495, Fiona Fiona Kandan. Η Fiona Kandan, είμαι από την Ιρλανδία, από το Εμπορικό Επιμελητήριο, υπό το φως του Brexit. Εμείς στην Ιρλανδία δεν πάμε πουθενά. 92% των Ιρλανδών θεωρούν ότι το να είμαστε μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η καλύτερη ευκαιρία που μα έχει δοθεί ποτέ. Ήρθα εδώ γιατί όπω και οι υπόλοιπε μικρομεσαίες επιχειρήσει θέλω να αναπτυχθώ περαιτέρω και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα με βοηθήσει και θα με διευκολύνει να το καταφέρω. Υπάρχει μόνο μία βεβαιότητα όσον αφορά την επιχείρηση, την επιχειρηματικότητα. Δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο. Όλα είναι ρευστά και αβέβαια. Το διεθνέ ε, περιβάλλον ε, κινείται με ηλικιώδεις ρυθμούς Υπάρχει ο αντίκτυπος των ε, νέων τεχνολογιών, η πολιτική αβεβαιότητα σε ολόκληρο τον κόσμο και πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα. Εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προετοιμαστούμε συλλογικά για να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει αυτέ. Αυτό θα ε, ε, πρέπει να σημαίνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσει θα ανταμείβονται για την καινοτομία του και για τι προτάσει του. Τώρα, η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο ενεργή όσον αφορά τις αρχές της. Πρέπει να διευκολύνουμε τους κανονισμούς και το γραφειοκρατικό βάρος που βαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έτσι ώστε να έχουμε τους πόρους και το χρόνο να καινοτομούμε και να αναπτυσσόμαστε. Ζητάμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη να ε, συνεργαστούν με τα επιμελητήρια ώστε η Ευρώπη να καταστεί το καλύτερο μέρος στον κόσμο για να κάνει κανείς ε, δουλειές και να αναπτύξει την επιχειρηματικότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ήρθε η στιγμή της ψηφοφορίας. Σας ε, θυμίζω ότι πρέπει να βάλετε το, την κάρτα σας ε, στο μηχάνημα. Ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση. Η ενιαία αγορά είναι ε, αρκετά εδρεωμένη έτσι ώστε να επιτρέπει στην εταιρεία σας να λειτουργεί και να ανταγωνίζεται ελεύθερα. Υπάρχει την ψηφοφορία. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Λήξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν 416, 111 είπαν ναι, αρκετά, 250 είπαν όχι. Ευχαριστούμε. Ερώτηση 2. Παρά τους γενικούς προϋπολογιστικούς περιορισμούς, η Κομισιόν έχει δίκιο να προτείνει αύξηση της χρηματοδότησης για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία για την, ε, για το, ε, για την επόμενη πολιετή ή δημοσιονομική περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψηφίστε. Ευχαριστούμε. Ψήφισαν 425, 402 είπαν ναι. Έχει δίκιο η Κομισιόν. Ερώτηση 3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εστιάζεται περισσότερες, περισσότερο σε πρωτοβουλίες με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ψηφίστε. Thank you very much. The vote is closed. Ευχαριστούμε. η ψηφοφορία. Έχουμε 124 ψήφισαν, 387 ναι, 6 μείον. Άρα είπατε ότι ναι, θέλετε να εστιαστεί περισσότερο σε περισσότερη προστιθέμενη αξία και 31 πήγαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερώτηση παριθμών 4. Ε, εξακολουθεί να έχει σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση για εμένα και την επιχείρησή μου Αρχίζει η ψηφοφορία. Παρακαλούμε, ψηφίστε. Ευχαριστώ πολύ. Περαιούται ψηφοφορία. 426 ψήφισαν, των οποίων 381 καταφατικά είπαν ναι, έχει σημασία η Ένωση για την επιχείρησή μου. 19 είπαν όχι και 26 απήχαν. Τελευταίο ερώτημα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τους επιχειρηματικούς δεσμούς με τις τρίτες χώρες ανοίγοντας το δρόμο για πρόσβαση αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανοίγει η ψηφοφορία. Ευχαριστούμε πολύ. Περαιούται ψηφοφορία. Ψήφισαν 425. 300 είπαν ναι, θα πρέπει να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύει του επιχειρηματικού θεσμού με τι τρίτε χώρε, ανοίγοντα τον δρόμο για τη μελλοντική του ένταξη. Ευχαριστώ όλου και όλε. Με χαρά δίνω το βήμα στην ΑΝΜΕΚΛΑ. Είναι επικεφαλής ε, του Κέντρου Ευρωπαϊκής Στρατηγικής, Πολιτικής Στρατηγικής Ε, είναι το εγκέφαλο σκέψης ε, του Ζων Κλοντ Γιούνκερ. Ευχαριστώ πολύ, ε, μεγάλη μου χαρά είμαι εδώ σήμερα. Ε, ξέρω ότι είναι εδώ ήδη και ο Σβαρνιέ, οπότε θα είμαι πολύ σύντομη. Απλά ήθελα να πω ότι σα μιλώ σήμερα όχι μόνο με την ιδιωτά μου Γενική Διευθύντρια ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ω αναλήτρια, αλλά και ω κάποιο που υπήρξε επιχειρηματία και προέρχεται από επιχειρηματική οικογένεια. Ε, κάτι για το οποίο είμαι περήφανη. Υπήρξα αυταπασχολούμενη για 11 χρόνια πριν να λάβω την ε, θέση αυτή και μπορώ να πω πόσο πολύ αξιολογώ το ότι προσφέρετε χρόνο από το πολυάσχολο πρόγραμμά σα για να έρθετε μέχρι εδώ να μας μιλήσετε και να απαντήσετε τα ερωτήματα αυτά που για μας έχουν μεγάλη χρησιμότητα. Απλά επιτρέψτε μου να δώσω ένα γενικότερο πλαίσιο για το πώ βλέπουμε το μέλλον τη Ευρώπη. Το λέω αυτό γιατί η συγγραφή ήταν πάρα πολύ μακρύ μέχρι ότου η Ευρωπαϊκή Ένωση έμαθε ότι ε, το Ηνωμένο Βασίλειο θα εγκαταλείψει την Ένωση και περιμένουμε ε, κλιμακωτές αντιδράσεις ιδιαίτερα έντονες τις επόμενους μήνες. Ε, είπαμε λοιπόν τι θα γίνει με αυτό, πώς θα το αντιδράσουμε. Κάναμε λοιπόν ε, μια συγγραφή πέντε διαφορετικών σενάριων που με πολύ σκόπιμο τρόπο διαμορφώθηκαν και είπαμε δεν θα πούμε εμείς προς τα που πρέπει να πάει η κατάσταση αλλά σίγουρα θα δρομολογούσαμε μια συζήτηση επί της οποίας όλοι οι άλλοι θα σκέπτονται. Θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν μια καλή προσέγγιση και τη χαιρέτησατε όλοι. Επίσης θα ήταν απαραίτητο να γίνει. Πρέπει να σας πω ότι κάποιες φορές οι προσδοκίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο υψηλέ και μάλιστα σε μια εποχή όπου οι ικανότητές μα και τα μας, ε, οι οικονομικέ μα δυνατότητε είναι τόσο πολύ περιορισμένα, ώστε κάποιε φορέ υπάρχει ε, μια αίσθηση ματέωσης στην Ευρώπη. Τα σενάρια αυτά βοήθησαν όλου να καταλάβουν ότι ναι, εμεί ξέρουμε ότι θέλουμε, θέλετε να κάνουμε πιο πολλά, αλλά θέλουμε πιο πολλά χρήματα και πιο πολλέ ε, αρμοδιότητε. Εξού και η σημασία για αυτή τη συζήτηση, που πέρα από το δυνόμιο του υπέρ κατά της Ευρώπης, μαύρο και άσπρο, πιο πολύ ή πιο λίγο, μπήκαμε έτσι σε πιο πολλές αποκεχρωσμένες λεπτομέρειες και στις γκρίζες ζώνες εκείνες οι οποίες θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να κάνουμε πιο πολλά πράγματα μαζί, πιο αποτελεσματικά, μέσα από την ενιαία αγορά. Γενικότερα λοιπόν αυτή η προσέγγιση υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχημένη και ευχαριστώ όλους και όλες εκείνες που συμμετείχαν ε, μετά από ανάγνωση της συγγραφή των διάλογο. Για όσους δεν το έχουν πράξει τους σας παροτρύνω γιατί έχει μεγάλη σημασία για το σημερινό μας διάλογο. Δεν θέλω να επιμείνω περαιτέρω. Έχω διάφορα σχόλια επί των παρεμβάσεων που λάβαμε, αλλά από όλα αυτά θέλω να συγκρατήσετε κάποια πράγματα πριν κλείσω. Είναι γεγονός ότι η Ευρώπη ε, έχει μια... Ε, ένα, ε, η Ευρώπη δεν είναι το σύμπαν, έχει ένα μικρό μερίδιο της παγκόσμιας πραγματικότητας και η δημόσια πολιτική δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Πρέπει να ετοιμαστούμε για μια συρρήγνωση και ο μόνος τρόπος για να μπορέσει η Ευρώπη να βγει προς τα εμπρός είναι να είμαστε μαζί και ενωμένοι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αυτό είναι ο μόνος τρόπος. Κατά δεύτερο λόγο, η Δύση πλέον δεν ε, έχει το μονοπόλιο της καινοτομίας και των ε, πρωτοποριακών τεχνολογιών. Έχουμε ε, στην Κίνα έναν ανταγωνιστή εκπληκτικό. Μια πρόκληση που πέρα από την οικονομία θα μπορούσε κάποτε να είναι και ιδιαίτερα διαβροτική για τις οικονομίες μας γιατί ε, υπάρχουν άνθρωποι που αναρωτιούνται πώς γίνεται οι Κινέζοι να έχουν τόσα χρήματα να χρηματοδοτούν τόσα πολλά στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης γιατί εμείς πάμε τόσο αργά στις δημοκρατίες μας πού, πού κολλάμε τέτοια ερωτήματα δεν είναι σωστό να τα θέτετε είναι ε, δύναμη η δημοκρατία να υποβάλει ερωτήματα και να ζητεί ευθύνε. μην παραπονιέστε συνέχεια είτε πόσο αργά πάνε τα πράγματα Προσπαθείτε να καταλάβετε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρί συζήτηση, χωρί διάλογο, χωρί αντιπαράθεση και χωρί να μην τεθούν όλα τα πράγματα πάνω στο τραπέζι. Η δημοκρατία αυτή καθεαυτή σίγουρα τώρα υπονομεύεται, την κατηγορούν και την επιτίθενται. 12 χρόνια τώρα βλέπουμε να συρρυκνούνται η δημοκρατία και, στη, και η ελευθερία στον κόσμο. Είναι αλήθεια και ουδέποτε είχαμε τέτοια πόλωση στι κοινωνίε όπω σήμερα ζούμε. Αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο εσεί ω επιχειρηματίε και επικεφαλή επιχειρήσεων πρέπει να γίνετε η φωνή του, του ορθολογισμού. Πρέπει εσεί να βοηθήσετε ότι όλοι θα δεχτούν την αλλαγή και την γενοτομία χωρίς ε, διάσπαση. Εσείς, η δική σα φωνή είναι αυτή που πρέπει να ακουστεί Όσο για μένα, εγώ δεν μπορώ παρά να σας ενθαρρύνω να ψηφίσετε, αλλά να σας ενθαρρύνω επίσης να ενθαρρύνετε και άλλους να ψηφίσουν. Στις επόμενες ευρωεκλογέ, τα πάντα διακυβεύονται, μα τα πάντα ε, είναι η πιο κρίσιμη καμπή της Ευρώπης. Και αν η Ευρώπη ε, πάρει μια στροφή αρνητική και επικίνδυνη προς ε, λιγότερη ελευθερία και προς το λαϊκισμό, αυτό σίγουρα θα έχει αρνητική επίπτωση επάνω σας. Το μέλλον της Ευρώπης λοιπόν σε εμά να να το διαμορφώσουμε. Είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Είμαστε ε, πολύ μεγάλη εμπορική δύναμη στον κόσμο με συμφωνίε με πάνω από 70 χώρε σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε μεγάλο συντελεστή. αλλά μόνο όταν είμαστε όλοι μαζί ω ενιαία αγορά. Εξεκολουθούμε να είμαστε ακόμα αρκετά δυνατοί για να μπορέσουμε να είμαστε οι διαμορφωτέ του πεπρωμένου μα. Και πραγματικά σε εσάς ανάγεται να το διαμορφώσετε μετά και από την εμπειρία που είχαμε και όλοι στρέφονται απέναντί μου και μου λένε είμαι η Ευρώπη, εγώ είμαι η Ευρώπη, εσείς είστε η Ευρώπη, εμείς είμαστε η Ευρώπη. Είναι το δικό μας λογικό πεπρωμένο. Εμείς πρέπει να το διαμορφώσουμε σήμερα και όταν όλοι τελικά πάμε στην ε, κάλπη να ξέρουμε τι κάνουμε και να το έχουμε κατά νου αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ, Άννα. Στίβ, ε, η Άννα νομίζω θα σου έχει πάρει τη δουλειά. Τι έχω να προσθέσω εγώ. Αυτό που έχω να πω είναι αυτή φορά ε, θα πρέπει όλοι να ψηφίσουμε. Είναι θέμα της Ένωσης, μην το ξεχάσουμε. Ε, παρακαλώ να συγχαρούμε όλους τους ε, ομιλητές και τους διαμορφωτές και καθώς αλλάζει η σύνθεση θα έχουμε ένα σύντομο βίντεο γύρω από τις ευρωεκλογές.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 Με μεγάλη χαρά χαιρετίζω ανάμεσά μας την παρουσία του κυρίου Μισελ Μπαρνιέ. Δεν χρειάζεται πια κάποια ιδιαίτερη παρουσίαση. Όλοι ξέρουν τον κύριο Μπαρνιέ. Καταρχήν, αν μου το επιτρέπετε, στη μητρική μου γλώσσα θα παρέμβω και θα πω στα γαλλικά, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Κρίστοφ Λάιτερ, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα καταρχήν να σας χαιρετήσω, να χαιρετήσω την ε, διαφορετικότητα και την ποικιλότητα, το βαθμό υπευθυνότητα που επιδεικνύεται στις επιχειρήσεις σας. Ε, οι χώρες από τις οποίες προέρχεστε, με 45 ε, χώρες μέλη του Euro Chambers, αποτελείται μια εξαιρετική δύναμη, μια μεγάλη ευκαιρία. Και το ότι εδώ μπορούμε να βρισκόμαστε όλοι μαζί σε αυτό το κοινοβούλιο των επιχειρήσεων, είναι τεράστια δυνατότητα που παρέχεται στην καρδιά της ε, Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ δεν είμαι υπερτεχνοκράτης της Ευρω... της... Ε, των Βρυξελών, πολιτικός είμαι, που εδώ και μερικό καιρό ε, δουλεύει και δεν έχει ξεχάσει τίποτα από ό,τι έχει μάθει επί τόπου στην περιφέρεια πρόεδρος της οποίας ήμουν εδώ και 20, ε, για 20 και πλέον χρόνια την Άνω Σαβοία, ορεινή περιοχή της Άλπης ε, και αργότερα υπουργό στη χώρα μου και τα όσα έμαθα μετά από δύο θητείες επιτρόπου, καταρχήν επικεφαλής περιφερειακής πολιτικής και στη συνέχεια ε, αρμόδιος για ένα θέμα που άπτεται της ε, δικής σας δραστηριότητα, ε, οι κοινέ σας προκλήσεις και η δέσμευσή μας σήμερα εδώ το αποδεικνύουν, το είδα άλλωστε και από την σφιγομέτρηση που ακούσαμε. Πέντε χρόνια λοιπόν ως ε, επίτροπος της εσωτερικής αγοράς. Ε, και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Τίποτα δεν ε, ξέχασα από τόσα έμαθα από την συχνότατη επαφή που είχα, πάντοτε επικοδομητική, ποτέ ε, θεωρητική, αλλά πάντοτε ουσιαστική με τις μικρομεσαίες και, και μεγάλες επιχειρήσεις σε αποστολές μου. Αυτό πάντοτε έχω κατά νου και το σκέφτομαι εν ώψη της αποστολής που μου ανέφερε ο κύριος Γιούνκερ ε, έχοντας μιλήσει με 27 διαφορετικούς επικεφαλής κρατών και με καλή συνεννόηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια αυτής της εξαιρετικής φύσεως και περιπλοκότητας ε, διαπραγμάτευσης ε, που ε, έχει να κάνει με, με την διασφάλιση τακτικού, αν μπορούμε, διαζυγίου με μια μεγάλη χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάρηκα ε, που μπορώ να ανταποκριθώ στην πρόσκλησή σα για να μιλήσουμε για κάποιε επιθέσει μου και κάποια στοιχεία που έχω να σα δώσω σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Τουλάχιστον ε, για εσά, εδώ από κοινού έχει μεγάλη σημασία να πάρουμε το λόγο γιατί πιστεύω ότι όπως και η Άννα το είπε προηγουμένω, ουδέποτε στην ιστορία της Ένωσής μας δεν βρεθήκαμε αντιμέτωποι ε, εντός και εκτός συνόρων ανατολικά, δυτικά, βόρεια, νότια με τόσες προκλήσεις, με τόσες απειλές που κάποτε φτάνουν στο σημείο να είναι τεράστιες challenges στα αγγλικά. Είναι λοιπόν η καλύτερη στιγμή να συναντηθούμε, να μιλήσουμε, να ακούσουμε οι mentors και για εμάς ε, από την πλευρά των Βρυξελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λάβουμε υπόψη μας την άποψη και τα αιτήματα των επικεφαλής των επιχειρήσεων, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε όλη την ποικιλότητα. Κύριε Πρόεδρε, αν κρίνω αγαπητέ Χριστιαν και Χριστόφ ε, από το μέχρι τώρα έργο που έχει επιτελεστεί σήμερα βρίσκεστε στον πυρήνα αυτών των διακύβευμάτων τόσο όσον αφορά τα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας την πρόκληση ε, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων της ε, κατάρτισης, της κινητικότητας και εκπαίδευσης των μεταναστών, την καταπολέμηση κατά της ανεργίας των νέων, την εξέβραση νέων αγορών μέσα από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες. Η Σίλια Άρμστρονγκ το είπε αυτό και κάτι που θα θελήσει και τις μικρομεσαίες, όχι μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντας βέβαια και την υφόρο ε, ανάπτυξη και προκειμένου από κοινού να μπορέσουμε να επενδύσουμε στις τεχνολογίες του μέλλοντος, να εμβαθύνουμε την ενιαία μας αγορά και να την προσαρμόσουμε στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Ορίστε ε, παραδείγματα θετικών ε, σχεδίων που απηχούν τις δεσμεύσεις και τις πρωτοβουλίες του Jean-Claude Juncker έτσι όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της είχε ενστερνιστεί. Ε, το θέμα αυτό των 27 χωρών που θα παραμείνουν μαζί κοντά η μία στην άλλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα τους οδηγήσει να επικεντρωθούν στη δόμηση μιας ε, στενανότερης ένωσης ριδόμενες κυρίες και κύριοι σε αυτό που κατ' εμέ τουλάχιστον συνιστά ε, το βασικό μας προτέρημα, το μεγάλο μας ατού αν θέλετε, ε, το, τη σερμαγιά μας, το κεφάλαιό μας αυτό που δεν είναι από την ενιαία αγορά. Η ενιαία αγορά που δεν είναι απλά μια αγορά, είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών που έτσι ξεκίνησε βέβαια, δεν λέω, αλλά μεταξελίχθηκε και έγινε κάτι πολύ παραπάνω. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα που όλοι από κοινού δομήσαμε ή κάτω από την όθηση και των δικών σας επιμελητηρίων και των επαγγελματικών σας αντιπροσώπων με κοινά όνοματα, κοινέ προδιαγραφές, κοινέ πιστοποιήσεις, δικαιώματα, κοινά δικαιώματα επίσης, ε, του καταναλωτή τα δικαιώματα, ε, κοινή νομοθετική ρύθμιση, εποπτεία και πάνω απ' όλα ε, κοινή δικαιοδοσία. Ε, αυτό είναι το σημαντικό και αυτό ακριβώς το πετύχαμε και έτσι ακριβώς το δομήσαμε εδώ και 20 χρόνια με τους Βρετανούς δίπλα μας. Πολύ να ξέρετε, δούλεψα με τα Euro Chambers και τους εκπροσώπους στην εποχή που είχα την τιμή να διατελέσω επίτροπος για την ενιαία αγορά και έχω κατά νου σημαντικά ζητήματα όπως η απλοποίηση των ε, πληστηριασμών και δημοσίων διαγωνισμών προμηθειών ή ακόμα το θέμα της επιτέλους ε, σύστασης ενιαίου ευρωπαϊκού διπλωμάτων ευρασιτεχνίας. Ε, ήταν μια πολύ θετική αυτή όλη η εξέλιξη, μια ατζέντα προόδου και εξέλιξη για την Ευρώπη και για τους Ευρωπαίους ε, και θα το πούμε ότι πραγματικά ε, και 27 υποφελήθηκαν Πολλά ακούστηκαν από τότε που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση που τώρα βιώνουμε για την ενότητα των 27 που εφαινόταν να διαρριγνύεται ε, μόνο που υπήρχε προσωπική θέληση για τη δέσμευση των 27 επικεφαλή κρατών του κυρίου Γιούγκερ, του Τούσκ, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά έχει να κάνει και με μια δουλειά που επιτελέσαμε και που θα συνεχίσω να επιτελώ προκειμένου να ακουστούν όλες οι γνώμες και να μιλήσουμε σε όλους ουδέποτε στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξήφθη διαπραγμάτευση τόσο κρίσιμη σε τέτοιο βαθμό διαφάνειας με τα 27 κράτη-μέλη και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα διατηρήσω μέχρι τέλους αυτή την αντιμετώπιση της διαφάνειας γιατί αποτελεί κλειδί της εμπιστοσύνης των 27 χωρών και του Κοινοβουλίου και στο πνεύμα αυτό είναι που θα συνεχίσω να εξηγώ, να ακούω ε, σε κάθε μία από τις πρωτεύουσες όχι μόνο ε, την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό που ξαναβρίσκω κάθε φορά με ευχαρίστηση γύρω από το τραπέζι των ε, συζητήσεων, αλλά και τις εργατικές και επαγγελματικέ ενώσεις, τα συνδικάτα και τις οργανώσεις χώρα προς χώρα. Θα συνεχιστεί αυτή η δουλειά γιατί αποτελεί κλειδί στην ενότητα. Θεωρώ ότι έτσι μέσο και μακροπρόθεσμα είναι που θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις που έχει μπροστά της η Ευρώπη ανάμεσα από τις οποίες προκλήσεις είναι και το Brexit, μοιραία. Ένα Brexit που όπως ξέρετε δημιουργεί πάρα πολύ άγχος. Ε, έχω κατά νου τους πολίτες και τι καθεστώς θα διέπει αυτούς. Μεγάλη ανησυχία για πολλούς επιχειρούντες ε, και πολλούς συλλογικού φορείς που ανησυχούν από τις αβεβαιότητες που επιστρεί το Brexit. Θα ήθελα εν ώψη αυτών των ανησυχιών να σας πω σαφέστατα πού βρισκόμαστε και τι μένει ακόμα να επιτελεστεί προκειμένου να καταλήξουμε μια συμφωνία τουλάχιστον στην τρέχουσα φάση με τους Βρετανούς ε, γύρω από τον Brexit και για να υπάρξει μια τακτική παρά μια άτακτη αποχώρηση. Περνάω τώρα στα αγγλικά, Χάιμε. Κυρίες και κύριοι, την 29η Μαρτίου του χρόνου, του επομένου χρόνου, που είναι και τα γενέθλιά σας, ε, κατά σύμπτωση. Μπα, το θυμάστε, το θυμάστε, με εκπλήσει. Δεν κάνω καμία σύνδεση, αλλά ξέρω ότι είναι τα γενέθλιά σας εκείνη την ημέρα. Για σε λιγότερο από 6 μήνες λοιπόν κυρίε και κύριοι, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποσυρθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανέκαθεν ε, σεβαστήκαμε την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση, ακόμα κι αν βαθιά μας λυπεί αυτή η απόφαση. Ωστόσο, σεβόμαστε την απόφαση του να φύγει από την ενιαία αγορά, ε, την απόφαση του να αποχωρήσει από την Τελωνική Ένωση και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία ε, έτσι ώστε η αποχώρησή του να είναι τακτική. Από την αρχή των διαπραγματεύσεων αυτών, έχουμε σημειώσει αρκετά καλή πρόοδο. Πράγματι, πολλά από τα κεφάλαια ε, του Συμφώνου αποχώρηση έχουν τύχει τη αποδοχή του Νομιμονού Συμβουλίου. Ορίστε το έκτυπο αντίγραφο του σχεδίου της συνθήκης 168 άρθρα το αποτελούν και τρία πρωτοκολλά. Γιβραλτάρ, Κύπρος και Ιρλανδία. Λίγο πολύ 80 με 85% του περιεχομένου αυτού του σχεδίου έχει ήδη τύχει συμφωνίας. Το πράσινο δείχνει ότι έχει υπάρξει συμφωνία με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Επί του παρόντος, παρά τα αυτά, υπάρχουν ακόμα κάποια τεχνικά θέματα και κρίτησιμα, μάλιστα που τα έχουμε πει το τέλος. Πρέπει να αποφασίσουμε περί της διακυβέρνησης για την εφαρμογή τη συμφωνία και το κέριο ε, θέμα της αγροτικής οικονομίας των γεωγραφικών ενδείξεων και των προστατευμένων ονομασιών στα 28 κράτη-μέλη. Πάνω απ' όλα πρέπει να αποφασίσουμε για το πώς θα αποφευχθεί το, ε, τα σύνορά μας μεταξύ των δύο Ιρλανδιών να δημιουργήσουν πρόβλημα για πολλούς λόγους πολιτικούς, ανθρωπιστικούς και οικονομικούς. Κυρίε και κύριοι, το Εμένο Βασίλειο επιθυμεί να αποχωρήσει ε, να αφήσει εμάς την ενιαία αγορά και την Τελωνική Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν και πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι στα προϊόντα που διακινούνται μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλεγχοι που σήμερα δεν υφίστανται. Έλεγχοι ΦΠΑ, τελωνική έλεγχη και έλεγχοι συμμόρφωσης που ε, αφορούν την ανάγκη να προστατευτούν οι καταναλωτές μας και οι εταίροι μας στο εμπόριο αλλά και οι επιχείρησει. Συμφωνήσαμε με το Βασίλειο ότι αυτοί οι έλεγχοι δεν είναι δυνατόν να διενεργούνται στα σύνορα μεταξύ Βορείου και Νοτιού Ιρλανδίας. Ε, κέριο ερώτημα λοιπόν παραμένει πού θα συμβαίνουν αυτοί οι έλεγχοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να σέβεται την εδαφική ακαιρεότητα και τη συνταγματική τάξη του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως ακριβώς και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευθεί να σέβεται την ακαιρεότητα της δική μα ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένη και τη Ιρλανδίας. Θυμάμαι την Φιώνα Κάντερμαν που κάτι προηγουμένω. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει την διεξαγωγή αυτών των ελέγχων με τον λιγότερο διζητικό τρόπο, όσο πιο λιγότερο διζητικά γίνεται, έτσι ώστε οι έλεγχοι η τελωνιακοί και του ΦΠΑ να, να γίνονται μέσα από τις τρέχουσες διαδικασίες διαμετακόμισης για να αποφευθούν έλεγχοι στα φυσικά ε, σύνορα. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος ως προς αυτό γιατί πιστεύω ότι πολλέ από τι επιχειρήσεις σας θα μπορούσαν να εμπλακούν σε αυτές τις μελλοντικέ διαμορφώσει των σχέσεων. Οι εταιρείε ε, στο Ενωμένο Βασίλειο που θα συμπληρώνουν επιγραμμικά τις ε, τελωνιακέ δηλώσει των προτέρων για την απαστολή ε, προϊόντων προ τη Βόρεια Ιρλανδία. Η μόνη ορατή συστηματική έλεγχη μεταξύ Βορείου Ιρλανδία και του Ηνωμένου Βασίλειου θα έχουν να κάνουν με την σάρωση, scanning των ε, γραμμικών κωδικών, barcodes, ε, στα ε, φορτηγά και τα εμποερματοκιβώτια. Αυτό μπορεί να γίνεται είτε στα ferry boats είτε στους λιμένες διαμετακόμισης. Αυτές οι διευθυντήσεις ήδη υπάρχουν εντός των κρατών μελών και πολλές από τις χώρες μας, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά την Ισλανδία, ε, αλλά και μεταξύ της υπηρετικής Ισπανίας και των Κανάριων νησιών το πράττουν αυτό, δεν είναι κάτι παλιό. Κατά δεύτερο, ε, ρυθμιστική ελεγχή βιομηχανικών ε, προϊόντων που μπορούν να διεξάγονται από τις αρχές ε, επαγρύπνησης της αγοράς. Αυτό και πάλι δεν χρειάζεται να συμβαίνει στα σύνορα, αλλά απευθείας στην αγορά ή στις εγκαταστάσεις ε, εταιριών στη Βόρεια Ιρλανδία ε, μένουν έξω οι έλεγχοι ζών των ζώων και φυτογειονομικών προϊόντων καθώς και προϊόντων ζωικής προέλευσης. Γιατί εκεί ισχύουν άλλοι κανόνες που είναι σαφέστατοι και γνωρίζω πολύ καλά ε, ε γιατί έχω κάποτε διατελέσει και υπουργό Γεωργία στη Γαλλία. Αυτοί οι έλεγχοι κυρίως συμβαίνουν στα σύνορα λόγω δεκιβευμάτων σχετικών προς την ασφάλεια της ε, διατροφικής ασφάλειας και της υγείας των ζώων. Ε, βέβαια, ε, στο μέλλον η Ιρλανδία παραμένει και πρέπει να παραμείνει μια ενιαία επιδημιολογική ε, περιοχή. Προφανώς αλλά αυτοί οι έλεγχοι ήδη ισχύουν και ασκούνται στον λιμένα του Λάον, στο Μπέλφαστ και στη Βόρεια Ιρλανδία. Οπότε ε, θα πρέπει να είμαστε σε άλλο ποσοστό. Όχι στο 10% των ζώων των ζώων και των ζωικών προϊόντων. Αυτό συμπεριλαμβάνει μια ουσιαστική αλλαγή όσον αφορά την κλίμακα πλέον. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλουν να υπάρχει φυσική μεθόριος μεταξύ Βορείου Ιρλανδία και Ιρλανδίας. Άρα λοιπόν, ό,τι φτάνει στη Βόρεια Ιρλανδία θα φτάνει και στη δική μα ενιαία αγορά. Ε, θα υπάρχουν διοικητικέ διαδικασίε οι οποίε σήμερα δεν υπάρχουν προκειμένου για προϊόντα τα οποία ε, μετακινούνται ε, προ την Βόρεια Ιρλανδία από την υπόλοιπη Βασίλειο. Πρόκλησή μα είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτέ οι διαδικασίε θα είναι όσο πιο ε, εύκολε γίνεται και όχι ιδιαίτερα επαχθεί, ιδίω για τι μικρέ επιχειρήσει. Κατανοώ για ποιο λόγο αυτές οι διαδικασίες πολιτικά είναι ευαίσθητες, αλλά επιτρέψτε μου τρεις παρατηρήσεις επ' αυτού. Πρώτον, το Brexit δεν ήταν κάτι που εμείς θελήσαμε, είναι κάτι που θέλησε το Ενωμένο Βασίλειο. Η πρότασή μα προσπαθεί ε, να βοηθήσει το Ενωμένο Βασίλειο να διαχειριστεί τις αρνητικέ επιπτώσεις ε, του Brexit στο, στη Βόρεια Ιρλανδία έτσι ώστε να ε, τηρείται και η εδαφική ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης η πρότασή μα περιορίζεται στο απολύτω απαραίτητο προκειμένου να ε, κατοχυρούνται τα σύνορά μα, οι τελωνιακέ ε, διαδικασίε και η τήρηση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών για τα προϊόντα. Δεν περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν την ελεύθερη ε, διακίνηση υπηρεσιών, προσώπων και προϊόντων ή κοινωνική ή περιβαλλοντική πολιτική. Ε, ισχύει πάντοτε η κοινή περιοχή ταξιδιωτικών μετακινήσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας. Και πάλι, η πρότασή μα παρέχει στη Βόρεια Ιρλανδία ωφέλη που καμία άλλη τρίτη χώρα δεν απολάβει. Ιδίως ε, ε, υπάρχει ε, η διαρκή επαφή στην κοινή αγορά των αγαθών και υπηρεσιών και εξακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βόρεια Ιρλανδία να αποφελούνται από τα ωφέλη της Τελωνιακή Ένωσης θα συνεχιστεί και η ενιαία αγορά ηλεκτρισμού στην Βόρεια Ιρλανδία όπως το Βασίλειο ζήτησε. Την περασμένη εβδομάδα συναντηθήκαμε με τον επικεφαλή επικεφαλεί όλων των βασικών πολιτικών κομμάτων στη Βόρεια Ιρλανδία. Είχα ήδη μαζί του συναντήσει και παλιότερα. Η πόρτα μου υπήρξε, είναι και θα παραμείνει πάντα ανοιχτή. Και η ομάδα μου συναντήθηκε τη Δευτέρα με μια ομάδα από επικεφαλής ε, πολιτικούς της Βόρειας Ιρλανδίας ακριβώς για ερωτήσεις και η πρότασή μα και για τον Brexit γενικότερα. Αλλά οι πιο πολλέ συζητήσει ε, έχουν προστιθέμενη αξία τη Βόρεια Ιρλανδία έτσι ώστε να επαμβληθεί το βάρος ε, του ελέγχου. Third, our proposal is just a safety net. Είναι λοιπόν πρότασή μα τη δημιουργία ενό δικτύου ασφαλείας. Χρειάζεται γιατί οι λεπτομέρειε τη μελλοντική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεγάλη Βρετανία θα, θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευση μετά την έξοδο τη Ευρωπαϊκή της, ε, Μεγάλη Βρετανία. Οπότε μπορεί να γίνουν κάποιοι έλεγχοι να καταστούν μια απαραιτητη Π.χ. μια ε, ε, κτηνιατρική συμφωνία μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα χρειάζονται τόσο συχνή έλεγχη και βεβαίως παραμένουμε ανοιχτοί στην ιδέα του να έχουμε μια τελωνιακή ένωση με το Ηνωμένο ε, Βασίλειο, όπως γιατί αυτό, ξέρετε, θα μας απαλλάξει από μια σειρά ελέγχων που δεν είναι Ε, Υπάρχει το θέμα της ε, Βόρειας ε, Ιρλανδίας και βεβαίως θα συμπεριλάβουμε στη συμφωνία όλα τα θέματα τα οποία πολλά από αυτά έχουμε ήδη συμφωνήσει με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά είναι σημαντικά, μερικές φορές είναι ιδιαίτερο σημαντικά και για τις δικές σας επιχειρήσεις, για τους εργαζόμενούς σας και για τις περιοχές σας, τις περιφερειές σας. Και συγκεκριμένα συμφωνήσαμε ήδη ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες που έφτασαν, κατέφθασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από το τέλος ε, του 2020, ε, δηλαδή ε, μέχρι και το 2020, 2,3 εκατομμύρια ξένοι υπάρχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και εργάζονται σε αυτό. Εντάξει, φυσικά το ίδιο ισχύει για τους Βρετανούς πολίτες που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσοι λοιπόν μετακινήθηκαν σε ευρωπαϊκέ χώρε πριν από αυτή την ημερομηνία θα μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν κανονικά τη ζωή του όπω και πριν. Θα παραμείνουμε σε στενή συνεργασία με τι οργανώσει που εκπροσωπούν του ε, σχετικού ε, πολίτε και κυρίω για να συζητήσουμε την υλοποίηση της συμφωνίας απόσυρσης. Ε, δεύτερον, όλες οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί από τα 28 κράτη-μέλη θα τηρηθούν σε επίπεδο 28. Αυτό σημαίνει ότι παραδείγματο χάρη για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή για την πολιτική συνοχής, για την περιφερειακή πολιτική, όλα τα τρέχοντα προγράμματα θα συνεχίσουν με τη συμμετοχή της Μεγάλης Βρετανίας και στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού προγράμματος. Και το Ηνωμένο Βασίλειο θα διατηρήσει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις ε, για τη μεταβατική περίοδο μέχρι το τέλος του 2020, ε, όπως ζήτησε εξάλλου. Και αυτό θα αφήσει χρόνο στις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν και θα αφήσει και χρόνο να ολοκληρωθεί η μελλοντική σχέση. Αλλά για να είμαστε σαφείς έτσι και ξεκάθαροι, Όλα αυτά θα ισχύσουν υπό την προϋπόθεση ότι θα, συμφωνήσουν, θα συμφωνήσουμε γενικά τη συμφωνία απόσυρσης η οποία θα πρέπει να επικυρωθεί. Ελπίζω στις αρχές του επόμενου έτους, μετά όταν θα υπογραφεί από το Ηνωμένο Βασίλειο, να επικυρωθεί λοιπόν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τη Μεγάλη Βρετανία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει τον τελευταίο λόγο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ε, κυρίες και κύριοι, πέρα από αυτό το χωρισμό που είναι δύσκολος όπως όλα τα διαζύγια και που θέλουμε να γίνει μετάξι, το πιο σημαντικό ε, φυσικά για το κοινό συμφέρον των χωρών μας, για την οικονομική σταθερότητα, για την ανάπτυξη, θα είναι προφανώς η μελλοντική εταιρική μας σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η μελλοντική σχέση θα πρέπει να προσδιοριστεί τώρα, να βρούμε το πλαίσιο που θα την εντάξουμε και τις παραμέτρους που θα τη διέπουν. Δηλαδή, για να είμαστε σαφείς, αυτή η μελλοντική σχέση θα αποτελέσει αντικείμενο νέων διαπραγματεύσεων αργότερα, πολλών διαπραγματεύσεων συγκεκριμένα. Θα έχουμε παράλληλες διαπραγματεύσεις, καμιά δεκαριά, που θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο του 2019 κατά τη στιγμή που θα έχει εξέλθει από τους θεσμούς το, Ευρωπαϊκό, το Ηνωμένο Βασίλειο, θα είναι τρίτη χώρα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν βάσει της ε, διακήρυξης που ετοιμάζουμε και η οποία ορίζει το ε, πλαίσιο τις διαπραγματεύσεις σε καμιά δεκαριά τομεί για να καταλήξουμε στο τέλος του 2020, πολύ σύντομα δηλαδή, σε μια ολοκληρωμένη διαπραγμάτευση με ε, τη νέα σχέση, με την έτερη σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με τους Βρετανούς εκ παραλίλου ε, πάνω σε αυτή την κοινή ε, δήλωση διακήρυξη που θα περιγράψει το πλαίσιο της μελλοντικής μας σχέσης. Πέρσι το Μάρτι, η αρχική κρατών κυβερνήσεων, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Ντόναλτ Τούσκ, ο Ζαν Κλοντ Ιουνκέρ, όλοι εξέφρασαν τη βούλησή τους να υπάρξει φιλόδοξη εταιρική σχέση, πολύ φιλόδοξη, με το Ηνωμένο Βασίλειο για το μέλλον. Είναι κάτι το οποίο το μοιραζόμαστε και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος, ο Αντώνιο Ταγιάννη, συμφωνεί απολύτω. Τώρα, στη συζήτηση με το Ηνωμένο Βασίλειο, βεβαίω λαμβάνουμε υπόψη τι θέσει οι οποίε εκφράστηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίω το έγγραφο αυτό που ονομάζεται Λευκή Βίβλο, η οποία προέκυψε από την ε, ε, συνεδρίαση τη σχετική και των Τσέκερς λεγόμενων και ε, συζητάμε πολύ για τα κεφάλαια με τους ε, Βρετανούς διαπραγματευτές για το, και, για το, και στο πολιτικό και σε τεχνικό επίπεδο. Γιατί λοιπόν αυτή η λευκή βίβλος πάντα θεώρησα ότι είναι χρήσιμη ε, διότι μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το benchmarking, τη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των δικών μας προτάσεων για το μέλλον και των ετοιμάτων ή των προτάσεων Ηνωμένου Βασιλείου, έτσι ώστε να βρούμε όλα τα σημεία σύγκληση. Έχουμε βρει πολλά π.χ. στον τομέα της, της εσωτερικής ασφάλειας, της ε, εξωτερικής πολιτικής, της στρατιωτικής συνεργασίας για θέματα άμυνας. Έχουμε βρει πολλά σημεία σύγκλησης ε, ε, όσον αφορά τις κλαδικές συνεργασίες που αφορούν πολλές από τις δικές σας επιχειρήσεις, κυρίως σε θέματα μεταφορών, αερομεταφορών π.χ. Επίσης, βρήκαμε κοινά σημεία ως προς την συμμετοχή της Μεγάλης Βρετανίας στις πολιτικές της Ένωσης, όπως το κάνουμε και με άλλες τρίτες χώρες, με την Νορβηγία, την Ελβετία, το Ισραήλ. Π.χ. σε θέματα έρευνας χρησιμοποιούμε τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για τις σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες. Και τέλος, έχουμε επίσης ε, βρει κοινά σημεία με στόχο σε κάποιους ε, τομείς να χρησιμοποιήσουμε τα μονομερή εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, ώστε να συνεργαστούμε καλύτερα με το Ηνωμένο Βασίλειο, π.χ. σε θέματα οικονομικών υπηρεσιών ή ε, προστασίας δεδομένων. Τώρα, ως προς την οικονομική μας εταιρική σχέση, πέρα από όλα τα σημεία σύγκλησης τα οποία είναι κεκτημένα, Απομένουν κάποιες βρετανικές θέσεις στη Λευκή Βίβλο που δεν αντιστοιχούν στις κατευθυντήριες γραμμές και στη εντολή που έχω εγώ από την από ευρωπαϊκή πλευρά. Συμφωνούμε και είναι σημαντικό για το Ευρωπημελητήριο και για εσάς έτσι ώστε να, να χτίσουμε τις μελλοντικέ μας σχέσεις για, την... Ε, για το τομέα του ελεύθερου εμπορίου χωρίς ε, τα ρήφες, χωρίς ποσοστώσεις. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό Πέρα λοιπόν από αυτό το ε, τομέα έχουμε δύο σημεία διαφοράς με την, Ευρωπαϊκή, με την Μεγάλη Βρετανία γιατί υπάρχει μια αντίφαση εδώ και μια αντίθεση σε σχέση με τα θεμέλια της ενιαίας αγοράς μας, της δικής σας ε, ενιαίας αγοράς. Καταρχάς, όσον αφορά ε, το, το, τα, τα, θέματα τα τελωνιακά, το μεγάλο... Η Μεγάλη Βρετανία θέλει να μπορεί να διαπραγματεύεται μόνο τι συμφωνίε τη με του Κινέζου, του Αμερικανού κτλ. παραμένοντα στην, ε, ε, στον τελωνιακό χώρο, ε, οπότε να μπορεί να επιβάλλει ταρίφες χαμηλότερες από τις δικές μας, δηλαδή εξωτερικά σύνορα, παραμένοντας στην ενιαία αγορά και υποφελούμενοι από τα ωφέλη. Αυτό κατά την άποψή μας θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα κίνδυνο που θα επιβαρύνει τις δικές μας επιχειρήσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να εφαρμόσει τις δικές του εξωτερικές ταρίφες, συλλέγοντας όμως για εμάς τα δικαιώματα των Ευρωπαϊκών Τελωνίων. Αυτό θα σήμαινε για μας απώλεια ελέγχου. Πρόκειται για τα τελωνικά δικαιώματα για το, Ευρωπαϊκ... για, το... για το ΦΠΑ και τα λοιπά. Εξάλλου, το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να ξαναβρει τον έλεγχο των συνόρων του. Ήταν και ένα θέμα στο δημοψήφισμα. Εμεί σεβόμαστε την επιλογή των Βρετανών. Αλλά η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας πρέπει υπό το ίδιο πνεύμα να αποδεχτεί ότι και εμείς θα διατηρήσουμε την ε, διαχείριση και τον έλεγχο των δικών μας εξωτερικών σύνορων και των τελωνιακών σύνορων μας. Ένα άλλο σημείο απόκλησης ε, αφορά πέρα από το τελωνίο ε, το, το, το ρυθμιστικό πλαίσιο, το κανονιστικό πλαίσιο για τα αγαθά. Θέλησε το Ηνωμένο Βασίλειο να ευθυγραμμιστεί με τα δικά μας πρότυπα, αλλά μόνο εν μέρη προκειμένου να διατηρήσει μια ε, ίδια συμμετοχή για την ε, εσωτερική αγορά, αλλά μόνο για τα αγαθά. Ταυτόχρονα θέλει να είναι ελεύθερο, να κάνει ό,τι θέλει σχετικά με το σύνολο των ε, κανονισμών που αφορούν την παραγωγή των αγαθών, είτε πρόκειται για υπηρεσίες, για απασχόληση, για κεφάλαιο, για κοινωνικούς κανόνες ή για περιβαλλοντικούς κανόνες. Ο καθένας εδώ καταλαβαίνει ότι ένα τέτοιο σύστημα ενιαίας αγοράς αλακάχτ θα προσφέρει μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους της ενιαίας αγορά. Δύο παράδειγματα για να γίνω σαφής. Ας πούμε στα χημικά προϊόντα. Ε, πολλές εταιρείες θα χρησιμοποιούν. Το 31% της, ε, της ε, τιμής, όχι της ε, ρυθμιστικής τιμής, όχι της πρώτης ύλης, σχετίζεται με το σεβασμό των κανόνων του προϊόντος, όπου ούτως ή άλλως ο κάθε εξαγωγέας πρέπει να σέβεται προκειμένου να εισέλθει στην αγορά μας. Είναι ο κανονισμός REACH. Αλλά το 69% της ρυθμισμένης τιμής του χημικού προϊόντος προκαλείται από το σεβασμό των άλλων κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγματος χάρη των περιβαλλοντικών κανόνων. Και αυτό το κομμάτι ε, η Μεγάλη Βρετανία θέλει να το αποφύγει και θέλει να διαφέρει από εμάς. Και εντάξει, τα νούμερα είναι ακόμη πιο χαρακτηριστικά. Μιλάνε από μόνα τους. Ξέρετε κυρίες και κύριοι ότι σε έναν οικονομικό τόμο από τα περιθώρια είναι πολύ ε, δύσκολα. Οι παραμικρές αποκλήσεις μπορούν να προκαλέσουν ε, πολύ σημαντικό ε, συγκριτικό πλέον και το Ηνωμένο Βασίλειο εφόσον παραμείνει στην ενιαία αγορά των αγαθών και όταν μπορεί να αποφεύγει όλα τα υπόλοιπα. Για τον λόγο αυτό, πολλοί ε, επικεφαλής ε, επιχειρήσεων, διευθυντές επιχειρήσεων και ο κύριος πρόεδρος εδώ, ζητήσαμε λοιπόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην κάνουν τίποτα που θα κάνει πιο εύθραυστη αυτή τη διαπραγμάτευση για την ε, εσωτερική αγορά. Η εσωτερική αγορά μετά τον Brexit θα συνεχίσει να, απο... να εκπροσωπεί πάνω από το 60% των εμπορικών συναλλαγών μας και ε, δείξατε κι εσείς τη δέσμευσή σας και το δέσιμο που έχετε με αυτή την αγορά. Λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις αρχές, ε, ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς, σεβασμός των αρχών, αυτονομία των 27 κρατών μελών, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπόψη και τις κόκκινες γραμμές της Μεγάλης Βρετανίας, με αυτά τα, το προτείναμε μια εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο που θα βασίζεται σε μια φιλόδοξη ε, συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών θα υπάρχει τελωνιακή συνεργασία, κανονιστική συνεργασία και επίσης και στο Levin Playing Field ε, θα ε, γίνει μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Αυτή την, ε, τη συνεργασία, την εταιρική σχέση θέλουμε να δημιουργήσουμε με τους Βρετανούς και θα αποτελέσει το, τη βάση των μελλοντικών οικονομικών μας σχέσεων. Και τίποτε δεν μας εμποδίζει στη συνέχεια να εμπλουτίσουμε τη σχέση αυτή κατά τη διάρκεια μιας διαπραγμάτευσης εκ νέου ε, με το σεβασμό βεβαίως όλων των βασικών αρχών. Θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας απλώς δύο πραγματάκια ως προς τις ε, συνθήκες αυτής της διαπραγμάτευσης που συνεχίζεται εντατικά αυτή την εβδομάδα νυχθημερών. Με βάση το στόχο μας που ορίστηκε από τις 27 αρχικούς κρατών και από το Κοινοβούλιο να, να, να έχουμε μια συμφωνία αύριο και προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε ε, τις δυνατότητες για μια τακτική έξοδο και να μειώσουμε βεβαίως το κόστος και για τις επιχειρήσεις και ε, για, ε, για, το μεγάλο, για τη Μεγάλη Βρετανία. Γνωρίζουμε ότι το κόστος θα είναι πολύ υψηλό, κυρίως για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και για κάποιους άλλους τομείς οικονομικούς. Γι' αυτό το λόγο το no deal ποτέ δεν υπήρξε σενάριο που τέθηκε επιτάπητος. Έστω και αν είναι ευθύνη μας να είμαστε προετοιμασμένοι για όλες ε, τις δυνατότητες. Ήθελα να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ακόμη και στην περίπτωση μιας συμφωνίας, εγώ δουλεύω σκληρά για μια α, συμφωνία, θα γίνουν προσαρμογές για πολλές ε, ε, από τις επιχειρήσεις σας εξαιτία των επιλογών της Μεγάλης Βρετανίας. Δεν θα είναι business as usual θα πρέπει, για να βοηθήσουμε λοιπόν, τι εταιρείε να αντιμετωπίσουν αυτέ τι προσαρμογέ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Γραμματέα, δημοσίευσε πάνω από 70 σημειώματα τα οποία είναι στη διάθεσή σα και τα οποία αφορούν όλου του ε, τομεί ε, που του αφορά ε, το Brexit. Θαλάσσιες μεταφορέ, ηλεκτρονικό εμπόριο, οικονομικέ υπηρεσίε. Ευχαριστώ λοιπόν το Ευρωεπιμελητήριο για τη στήριξη που μα έδειξε. Μα συνοδεύσατε σε αυτή την προετοιμασία. Η Task Force που διευθύνω παραμένει επίση στη διάθεσή σα. Αυτά ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσω και με ένα προσωπικό στοιχείο κυρίε και κύριοι. Ε, στη θέση μου ω υπεύθυνο αυτών των διαπραγματεύσεων και υπό τον έλεγχο των Ευρωπαίων Ιθινόντων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλω να πω αυτό που πιστεύω εγώ. Ω κάποιο ο οποίο όταν πρωτοψήφισε στη χώρα του κάποτε το 1972 ήμουν 21 ετών Είχαμε τότε ένα δημοψήφισμα στη Γαλλία για, το, για την ένταξη της Ιρλανδίας, της Δανίας, της Νορβηγίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Και εγώ ψήφισα ναι. Και μάλιστα έκανα και εκστρατεία για το ναι. Γιατί και τότε μέλη του ε, κόμματος ε, του, Ντεγκόλε δεν συμφωνούσαν. Δεν το μετάνιωσα γιατί πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να ξέρουμε να έχουμε κατά νου είναι η ισχύ εν τη ενώση. Ε, είμαστε λοιπόν 28, 27, καλύτερα να είμαστε 27 για να μπορούμε να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας, τις αξίες μας, να γίνουμε ε, σεβαστοί, να ακουστούμε τα επόμενα 30-40 χρόνια. Λυπάμαι λοιπόν ε, για αυτή την κατάσταση. Θεωρώ ότι καλύτερα είναι να είμαστε μαζί. Νομίζω ότι το Brexit δεν έχει καμία προσθέμενη αξία. Καμία. Είναι μια αρνητική διαπραγμάτευση lose-lose game. Δεν είναι win-win, είναι lose-lose. Χάνουμε όλοι. Και η έκβαση αυτή τη διαπραγμάτευση είναι σημαντική πέρα από τη σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο για το μέλλον όλη τη Ευρώπη. Ε, και είμαι πεπισμένο. Από την πλευρά μα προσπαθούμε να καταλέξουμε σε πιο δίκαιη, δυνατή και συγκεκριμένη συμφωνία για αυτό το διαζύγιο και είμαστε φιλόδοξοι. Για το μέλλον θέλουμε να προσπιστούμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών, των επιχειρήσεων και θέλουμε να διατηρήσουμε και τα θεμέλια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Και για να τα καταφέρουμε κύριε και κύριοι, όσον με αφορά, θα συνεχίσω βεβαίω με τις διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος. Εξ ονόματο τη Ένωσης θα συνεχίσω να σέβομαι τις αρχές που μόλι ανέφερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Ευρωπαίων Ιθινόντων, έτσι όπω ε, ε, έγιναν γνωστά ακόμη και κατά το δημοψήφισμα. Και κύριε και κύριοι, χωρίς κανένα εκδικητικό πνεύμα, χωρίς ε, καμία επιθετικότητα, με τον ίδιο σεβασμό, με πολύ σεβασμό για μια μεγάλη χώρα η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνει σύμμαχός μας και εταίρος μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μισελ Μπαρνιέ. Και τώρα θα κηρύξει τη λήξη ο πρόεδρος ο Κρίστοφ Λάιτεν. Αγαπητά μέλη του Επιχειρηματικού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακούσαμε. Συγχαρητήρια. Πολύ σκληρό το έργο σας. Πολύ δύσκολο. Και νομίζω ότι για να βρούμε μια διέξοδο και για να έχουμε τις καλύτερες επιλογές για το μέλλον, αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι και το αποτέλεσμα. Εσείς είδατε το χειροκρότημα που λάβατε, πιστεύω ότι χαίρετε του πλήρου σεβασμού μας για όλη σας την προσπάθεια. Κινηθήκατε μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση και θέλω να σας συγχαρώ γι' αυτό και βλέπουμε τι κάνουν οι επιχειρήσεις, βλέπουμε ποια είναι τα προβλήματά τους και προσφέρουμε ιδέες σχετικά με το πώς θα το διαχειριστούμε όλο αυτό με έναν ε, ρεαλιστικό και πρακτικό τρόπο. Κυρίες και κύριοι, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ψηφίσατε και έτσι λοιπόν με τις ψήφους σας επηρεάζετε τον οργανισμό σας, το Ευρωεπιμελητήριο. Ψηφίσαμε ναι κατά περισσότερο από 80% για μια πολιτική ενσωμάτωσης, πάνω από 70% υπέρ ενός συμβουλίου με αποφάσεις πλειοψηφίας και πάνω από 80% να παραμείνουμε ενωμένοι και να το αντιμετωπίσουμε καλύτερα το πρόβλημα που θα ε, μας έλθει από το εξωτερικό. Έχουμε λοιπόν περισσότερη ενότητα και αυτό είναι σημαντικό, είναι ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα της σημερινής ε, ημερίδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θέλω να προσθέσω μια κουβέντα. Ευχαριστούμε για την πειθαρχία που επιδείξατε. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ μαζί μας. Είχαμε τρεις ενότητες και είστε επιχειρηματίες, είστε απασχολημένοι, πρέπει να κάνετε τη δουλειά σας, αφήσατε τη δουλειά σας για να έρθετε εδώ και ήρθατε. Και μία συμβουλή μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. δεν είναι ωραίο να μιλάει ο πρόεδρος της Κομισιόν σε ένα φόρουμ που είναι σε μια αίθουσα που είναι άδεια. Αυτές οι εικόνες πάνε σε όλη την Ευρώπη και βοηθούν αυτούς οι οποίοι εξαρτώνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους θεσμούς Πρέπει να το γνωρίζουμε. Είναι σαφές ότι μπορεί να είναι παρόντα τα μέλη του Κοινοβουλίου σε όλες τις ολομέλειες. Πολλές ε, συνεδριάσεις, ε, ε, επιτροπές, το ένα το άλλο, αλλά όταν ο πρόεδρος της Κομισιόν εξηγεί την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάξει, θα πρέπει να είναι όπως της είπα όπου η γερουσία είναι κατάμεστη. Θα πρέπει να είναι όπως σε άλλες χώρες, όπου ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης κάνει μια σημαντική δήλωση, δίνει ένα σημαντικό μήνυμα. Η Ευρώπη πρέπει να το έχει αυτό επίσης. Αυτό θέλουμε να καταφέρουμε και νομίζω ότι ο πρόεδρος Ταγιάννη και ο ίδιος υποφέρει από αυτό και θα πρέπει να του δείξουμε τι κάνουμε εμείς και να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκφράσατε επίσης, ε, εκφραστήκατε με τις παρεμβάσεις σας, ε, συμβάλλατε στις συζητήσεις. Το ευρωπαϊκό ιδεώδες είναι σημαντικό. Βοηθάμε όλοι τον επιχειρηματικό κόσμο. Ε, δεσμευόμαστε να αναλάβουμε την κοινωνική μας ευθύνη. Αναφέρθηκαν οι ανάγκες μας, αλλά αναφέρθηκαν και οι δυνατότητές μας. Δυνατότητες εξυπηρέτησης των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τα πήγατε περίφημα. Τελικώς, θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό και την ομάδα που έκαναν εξαίρετη δουλειά, εξαιρετική διοργάνωση και ευχαριστούμε και τον Αρνάντο. Κηρύττουμε λοιπόν τη λήξη της συνεδρίασής μας.